Well, good afternoon. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίζω τα μέλη, τους προσκεκλημένους ομιλητές και το κοινό στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Τάξη 3 με θέμα την καταπολέμηση των επιζήμιων φορολογικών πρακτικών. Θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων καταρχήν με τη διαμεσολαβήτρια, την κυρία Οράιλη, που θα ήθελα να ευχαριστήσω που δέχτηκε την πρόσκλησή μας. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Οράιλη. Οι προηγούμενες ειδικέ και εξεταστικές επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξέφρασαν την ανησυχία τους ως προς τη διαφάνεια ε, στο Συμβούλιο σε θέματα φορολογικά. Όπως γνωρίζετε, πρόσφατα η διαμεσολαβήτρια εξέδωσε συστάσεις για τη διαφάνεια ε, της νομοθετικής διαδικασίας στο Συμβούλιο. Η Επιτροπή μας, ΤΑΞ 3, επιθυμεί να μάθει πώς αξιολογεί μεταξύ άλλων η κυρία Ορέιλη ε, τον πιθανό αντίκτυπο των προσφάτων συστάσεων ε, για τη διαφάνεια στις μεθόδους λειτουργίας του Συμβουλίου πάντα στα φορολογικά ενδεχομένως και του συμβουλευτικού οργάνου και τι γίνεται με τον κώδικα διοντολογίας για τη φορολόγηση των επιχειρήσεων. Ακολουθεί πάνελ ε, ε, με θέμα Ευρωπαϊκός Κατάλογος Μη Συνεργάσιμων Κρατών για φορολογικά θέματα ε, που θέσπισε η Ένωση τον περασμένο Δεκέμβριο. Φιλοδοξεί να είναι ο κατάλογος αυτός αποφασιστικό εργαλείο στην καταπολέμηση αυτών των φορολογικών πρακτικών. Ο κώδικας συμπεριφοράς για τη φορολόγηση των εταιριών υπήρξε κομβικός για την κατάρτιση αυτού του καταλόγου αρχικά και στη συνέχεια την τροποποίησή του. Γι' αυτό ε, προσκαλέσαμε τον πρόεδρο της ε, λόγω ομάδας που δυστυχώς ε, για λόγους αλλημένων υποχρεώσεων δεν κατάφερε να δεχθεί την πρόσκληση. Αλλά η κυρία Φαμπρίτσα Λόπε Κορέρα μας είπε ότι πριν δεχτεί την ε, πρόσκλησή μας θέλει να διαβλεφθεί με την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων, Κορεπέρ. Θέλουμε να δούμε και τον Υπουργό ε, Βλάντισλαβ Κοράνοφ, Υπουργό Οικονομικών της ε, Βουλγαρίας και Προεδρεύοντα του Συμβουλίου ΕΚΟΦΗΝ για τα θέματα αυτά των επιζήμιων φορολογικών πρακτικών και τις προθέσεις της Βουλγαρίας για τη μελλοντική φορολόγηση των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, το γραφείο του Υπουργού ε, δήλωσε αδυναμία και πριν από λίγη ώρα μας είπε ε, ο Υπουργός, ε, πήραμε επίσημη απάντηση από το γραφείο του όπου ε, αρνείται και απορρίπτει την πρόσκληση και είπε ότι έχει παρουσιάσει ήδη τις ε, προτεραιότητες της Βουλγαρικής Προεδρίας στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων ΕΚΟΝ και θεωρεί ότι αυτός είναι ο βασικός του συνομιλητής από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μάλλον δεν καταλαβαίνει την κατάσταση για το τι επικρατεί στο Κοινοβούλιο και στις σχέσεις Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Και η κυρία Λιάννα Παύλοβα, υπουργό, καθώς και η κυρία Μόνον Παναγιώτοβα, ε, αναπληρώτρια υπουργό ε, Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Προσεκλήθησαν και δύο σε περίπτωση που δεν θα ε, δύνατο ο κύριος Γκουράνοφ να παρευρεθεί. Δυστυχώς δεν δέχθηκαν την πρόσκληση αυτή οι δύο κυρίες. Θεωρώ λοιπόν αυτό βαθύτατα ανησυχητικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο που εκπροσωπείται ε, προκειμένου από την Προεδρία του θα πρέπει να δίνουν το παράδειγμα αγαστής συνεργασίας και καταπολέμησης κατά ε, των εγκλημάτων ε, των οικονομικών φοροαποφυγής και φοροδιαφυγή και όχι το αντίθετο. Θα ήθελα να ενημερώσω τα μέλη της Επιτροπής μας ότι αυτό το θέμα το συζητήσαμε σήμερα το πρωί στους συντονιστές και θα λάβουμε κάθε απαραίτητο μέτρο έτσι ώστε να εμπλακεί και το Συμβούλιο στις εργασίες μας. μετά από τις βασικές αποκαλύψεις που έκαναν οι δημοσιογράφοι και τις συστάσεις οποίες προέβη οι προηγούμενοι και άλλες επιτροπές του Κοινοβουλίου και μετά από τις πρωτοβουλίες που έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει το Συμβούλιο να κάνει ό,τι μπορεί για να ε, ανταπεξέλθει και στη δική του ε, υποχρέωση. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα καλωσορίζουμε τέσσερις εμπειρογνώμονες, την καθηγήτρια Έλιφαντε Βέλντε από το Πανεπιστήμιο του Χάσελ του Βελγίου, Έχουμε τον κύριο Άλεξ Κόπχαμ, Διευθύνοντα Σύμβουλο του ε, Δικτύου για τη Φορολογική Δικαιοσύνη. Έχουμε τον κύριο Γιώχαν Λάγκεροκ τη Oxfam και τον κύριο Βαλέχ Μουταλιέ, Διευθυντή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριος Βαλέχ Μουταλιέ, ε, σας καλωσορίζω όλους. Θέλουμε να ακούσουμε και πώς θα βελτιωθεί ο κατάλογος αυτός με τις μη συνεργαζόμενες χώρες για να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Στείλαμε και ερωτηματολόγιο. Βέβαια, δεν απάντησαν όλοι οι ε, ενδιαφερόμενοι γιατί ήταν αργά, μπορούν να απαντήσουν σήμερα γραπτός. και στην ιστοσελίδα τη ε, Επιτροπής μας θα βρείτε απαντήσει, αλλά και μετά τη συνεδρία σε άλλε γραπτέ. Καλωσορίζω θερμά την κυρία Έμιλι Ορέιλι, Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια. Σας στείλαμε διάφορες ερωτήσεις για διάφορα θέματα που μας ενδιαφέρουν είναι μεγάλη μας τιμή το γεγονός ότι μπήκατε στον κόπο και βρήκατε το χρόνο ε, να μας απαντήσετε γραπτός. Θα τα διαβιβάσουμε αυτά στα μέλη της Επιτροπής μας. Και τώρα κυρία Ορέλη σας καλώ να κάνετε την εισαγωγή σας μέχρι 10 λεπτά παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την πρόσκληση που μου απίφθηνε προκειμένου να συζητήσουμε σήμερα το απόγευμα την ε, καταπολέμηση των επιζήμιων φορολογικών πρακτικών καθώς και το έργο μου σχετικά με, το, με τις μεθόδους εργασίας του Συμβουλίου. Θα σας δώσω μια επισκόπηση της έρευνάς μου όσον αφορά τη λογοδοσία του Συμβουλίου και την πρόσβαση στα έγγραφα που άνοιξα πριν από ε, ένα χρόνο και που έκλεισε αυτή την εβδομάδα και στη συνέχεια μπορώ να απαντήσω σε ερωτήσεις τα έγγραφα παραδείσου του 2017, η μεγαλύτερη διαρροή εγγράφων που αφορούν ε, επιζήμιες ε, φορολογικές πρακτικές εταιριών μετά τα έγγραφα του Πανανά, επανεπικέντρωσε την συζήτηση σε ζητήματα φορολογικών παραδείσων, φοροαποφυγής, φοροδιαφυγής και τις αντίστοιχες προκλήσεις που σχετίζονται με, την, ε, με τις ανισότητες όσον αφορά το εισόδημα. Γι' αυτό και καταλήξαμε στην δημιουργία αυτής της ε, επιτροπής που ακολουθεί το έργο παλαιότερων επιτροπών ε, προκειμένου να παρακολουθείτε το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν γίνονται αρκετά προκειμένου να υπερασπιζόμαστε τα κοινά συμφέροντα, τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου όσον αφορά τα φορολογικά ζητήματα. Η διαφάνεια προφανώς και αποτελεί κομβικό στοιχείο σε, αυτή, σε αυτό το έργο. Αυτοί που θέλουν να αποφύγουν τον δημόσιο έλεγχο ε, των φορολογικών τους πρακτικών έχουν ε, συμφέρον βεβαίω να ε, διασφαλίσουν την εμπιστευτικότητά του. Οι εταιρείε που βοηθούν λοιπόν αυτούς ε, μπορούν αντίστοιχα να έχουν παρόμοια συμφέροντα. Η Appleby ε, απέσυρε την, ε, την ε, μήνυση που είχε, καταστήλει, που είχε υποβάλει κατά των δημοσιογράφων Guardian και Independent που, ε, έφεραν στη δημοσιότητα αυτό το θέμα. Προφανώς η, η εμπιστοσύνη των πελατών αποτελεί στοιχείο της εταιρική ανάπτυξης, αλλά αυτό δεν μπορεί να αποκλείει ότι οι εμπιστευτικές δράσεις θα πρέπει να συνάδουν με τον νόμο και τις βέλτιστες πρακτικές. Οι, δημόσιοι θεσμοί επίσης πρέπει να λογοδοτούν για τις δικές τους αποφάσεις στον τομέα αυτό. Οι απλοί άνθρωποι, οι απλοί πολίτες δεν ε, έχουν έλεγχο επί των ιδιωτικών εταιρεών και γι' αυτό το λόγο βασίζονται στους δημόσιους θεσμούς προκειμένου να υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους. Και αυτό είναι το έργο που κάνει η δική σας Επιτροπή. Η λογοδοσία λοιπόν όμως καθίσταται δυνατή μόνο εφόσον υπάρχουν έγκαιρα ε, οι σχετικές πληροφορίες. Κάτι που είναι αόρατο που προφανώς δεν μπορεί να μετρηθεί και δεν μπορεί και να αξιολογηθεί. η οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν λοιπόν ένα, γενικά ένα υψηλό επίπεδο προσβασιμότητας των εγγράφων τους, αλλά το Συμβούλιο συγκεκριμένα χρειάζεται να κάνει βήματα βελτίωσης. Δεν έχουμε λάβει συγκεκριμένα παράπονα όσον αφορά τη διαφάνεια της ομάδας για τον κώδικα διοντολογίας για, τις, ε, για τη φορολόγηση των επιχειρήσεων, αλλά η ομάδα αυτή για την φορολόγηση των επιχειρήσεων αποτελεί ένα επίσημο προπαρασκευαστικό όργανο του Συμβουλίου που ε, προετοιμάζει ε, διοικητικά έγγραφα και γι' αυτό το λόγο εμπίπτουν στη δική μου αρμοδιότητα. Ο πιο απλό τρόπο για να χειριστώ το ζήτημα της διαφάνειας σχετικά με αυτήν την ομάδα θα ήταν μέσω ενός, μιας καταγγελίας ε, σε περίπτωση που υπάρχει άρνηση πρόσβαση σε έγγραφα ή σε περίπτωση που χορηγηθεί μόνο εν μέρη πρόσβαση. Γι' αυτό και σε αυτές τις περιπτώσεις θα μπορούσα να καταλήξω στο αν η, άρνηση, η εκάστοτε άρνηση ήταν ε, σύνομη ή όχι. Τα υψηλά πρότυπα βεβαίω δεν σημαίνει ότι πρέπει τα πάντα να είναι διαφανή ή να είναι άμεσα διαφανή και προσβάσιμα. Κάποιε φορέ είναι προ το συνδημόσιο συμφέρον κάποια έγγραφα να μην δημοσιεύονται ή να μην δημοσιεύονται έω τον κατάλληλο χρόνο. Όμω, ο κανονισμό για τη διαφάνεια, ο 1049 του 2001, ε, λαμβάνει ως αφετηρία την υπόθεση ότι τα έγγραφα που έχει στην κατοχή της Ευρωπαϊκή Ένωση θα δημοσιευθούν εκτός ε, αν υπάρχει συγκεκριμένη εξαίρεση που εφαρμόζεται. Κάποιες εξαιρέσεις επίσης υπόκεινται σε έλεγχο ε, δημόσιο. Σε άλλα με άλλα λόγια, αν υπάρξει δηλαδή για παράδειγμα μια εμπορική ζημία, ακόμη και αν υπάρξει, μπορεί το δημόσιο συμφέρον να υπερισχύει. Κάποιες ε, εξαιρέσεις βεβαίως θεωρούνται υποχρεωτικές. Πρόκειται για αρχεία που σχετίζονται με τη δημόσια ασφάλεια, ζητήματα άμυνας και ασφάλειας, διεθνείς σχέσεις, καθώς και την πολιτική, την νομισματική και δημοσιονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι θεσμοί και πάλι πρέπει να ετυλογούν όμως την, ε, την εξαίρεση αυτή. Σε ό,τι αφορά τα τα, τα, τους τρίτους, όπως είναι για παράδειγμα χώρες που μπορεί να διευκολύνουν τη φοροαποφυγή, τότε η τρίτη αυτή χώρα ε, πρέπει να ε, τύχει διαβούλευσης, όμως κάθε απόφαση θα πρέπει να συνάδει με τον κανονισμό 1049. Αντίστοιχα, αν το κράτος, αν κάποιο κράτος μέλος ζητήσει να μην δημοσιευθεί κάποιο έγγραφο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε θα πρέπει να αξιολογηθεί αν πράγματι συνάδει ε, μια τέτοια εξαίρεση με τον κανονισμό. Η φορολόγηση είναι προφανές ότι είναι ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα και αμφιλογόμενο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα ζήτημα ευαίσθητο και εσωτερικά στα κράτη-μέλη, αλλά και για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τις εμπορικές και διπλωματικές σχέσεις με τρίτες χώρες, κάποιες, ε, από τις οποίες έχουν φορολογικά καθεστώτα τα οποία μπορεί να βλάψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα οικονομικά της συμφέροντα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η δυναμική ε, να αντιμετωπίζονται αυτά τα ζητήματα με αδιαφανή διπλωματία μπορεί να έρχεται σε σύγκρουση με τις αρχές του 1049. Η ομάδα για, την, ε, για τον κώδικα διοντολογία για την φορολόγηση των επιχειρήσεων έχει ε, αναλάβει να ασχοληθεί με μια σειρά από πολύ σημαντικά ζητήματα συμπεριλαμβανομένων των, ε, της εξέτασης επιζήμιων πρακτικών φορολογικών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατάρτιση ενός καταλόγου τρίτων χωρών που παρουσιάζουν προβλήματα και συμβουλεύει το Συμβούλιο για το ποιε χώρε πρέπει να είναι σε αυτόν τον κατάλογο, ποιε πρέπει μπορούν να βγουν και τι ακριβώς ε, αιτιολογεί την προσθήκη ή την αφαίρεση μια τέτοια χώρα από αυτόν τον κατάλογο. Και αυτό χρειάζεται υψηλό επίπεδο διαφάνεια αν θέλουμε οι πολίτε να διαβεβαιωθούν ότι πράγματι ε, αναλαμβάνονται σημαντικέ δράσει για να προστατευτούν τα συμφέροντά του. Όμω, σε κάποιε ε, περιπτώσει αντιμετωπίζουμε σημαντικέ προκλήσει διαφάνεια. Όπω είπα, δεν έχω λάβει ε, κάποιο συγκεκριμένο, παράπονο ή καταγγελία όσον αφορά την ομάδα αυτή. Όμω, έχουμε λάβει παράπονα γενικά για το Συμβούλιο που σχετίζεται και με, την μικρή, με το χαμηλό επίπεδο γνώσης που έχουν οι Ευρωπαίοι πολίτε για αυτό το θεσμικό όργανο. Γι' αυτό και επικεντρωθήκαμε σε συζητήσεις για νομοσχέδια που συζητούνται στις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου και στην ε, Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσωπιών. Ε, ξεκίνησα λοιπόν το Μάρτιο του 2017 αυτή τη στρατηγική έρευνα με δεδομένο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είναι συνομοθέτες όμως αυτός ο δεσμός ε, δεν, εξασφαλίζει ίδιο επίπεδο λογοδοσίας και των δύο θεσμικών οργάνων. Ενώ το Κοινοβούλιο έχει ανοιχτά την, ε, και προσβάσιμα τα στοιχεία του όσον αφορά την διαδικασία και τη συζήτηση που ακολουθείται κατά την εξέταση ενός νομοσχεδίου το, το ίδιο δεν ισχύει για το Συμβούλιο. Αυτό που εμείς επιμένουμε είναι ότι θα πρέπει η νομοθετική διαδικασία να είναι επαρκώς διαφανής προκειμένου οι Ευρωπαίοι πολίτες να μπορούν να συμμετέχουν στην ε, νομοθετική διαδικασία ε, στον ε, προβλεπόμενο βαθμό και για να μπορούν να το κάνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες αυτοί θα πρέπει έγκαιρα να γνωρίζουν ποια είναι η θέση που το κράτος μέλος τους έχει υιοθετήσει για ένα συγκεκριμένο νομοσχέδιο που συζητείται. Αν ε, σε αυτό το πράγμα, σε αυτή τη ε, διαδικασία υπάρχει αδιαφάνεια, τότε υπάρχει πρόβλημα. Και αυτό σχετίζεται και με το γεγονό ότι ε, υπάρχει αυτή η διάχυτη αίσθηση στου Ευρωπαίου πολίτε ότι κάποιοι γραφειοκράτε καταρτίζουν την νομοθεσία και όχι τα ίδια του τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό και επιμένω ότι η ε, η έγκαιρη ε, και πλήρης δημοσίευση ε, των εγγράφων μπορεί να βοηθήσει στην εγγένη άποψη και εικόνα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους της. Προφανώς η, η, η ισορροπία ανάμεσα στις... αν, μάλλον η νομοθετική διαδικασία ακολουθείται πίσω από κλειστέ πόρτε, δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπερασπιζόμαστε τα, τα δημόσια συμφέροντα. Και αυτό βεβαίω σχετίζεται και με τον τομέα τη φορολογία. Θεωρώ ότι η η τρέχουσα πρακτική του Συμβουλίου είναι πλημελής γιατί ακόμα και η αδυναμία να καταγράφονται τα κράτη-μέλη που τοποθετούνται σε ομάδες εργασίας και λόγω του περιορισμού της πρόσβασης σε νομοθετικά έγγραφα με ε, τη διαβάθμιση αποτελούν μεγάλο πρόβλημα. Στις 9 Φεβρουαρίου 2018 έκανα τρεις συγκεκριμένες συστάσεις και διάφορες προτάσεις προς το Συμβούλιο για το πώς μπορεί να βελτιώσει τον, το επίπεδο λογοδοσίας του. Το Συμβούλιο δεν απάντησε στις συστάσεις αυτές εντός της τρίμηνης περίοδου που, προβλέπεται που εξέπνευσε στις 9 Μαΐου 2018. Όμως λόγω της πολύ μεγάλης ανάγκης ε, που, υπάρχει για νομοθετική διαφάνεια θα συνεχίσω την έρευνά μου και μάλλον θα συντάξω μια ειδική έκθεση σχετικά με την έρευνα αυτή στο Κοινοβούλιο αυτή την εβδομάδα. Θεωρώ ότι οι επιτροπέ ΑΦΚΟ και ΠΕΤΗ θα συντάξουν σχετική έκθεση και όλα τα, όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου θα μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία και το επιτελείο μου βεβαίω ε, είναι στη διάθεσή σα για να σα ενημερώνουμε για τα επόμενα βήματα. Πρέπει επίση, βεβαίω να σα ενημερώσω ότι η δουλειά μου αφορά την νομοθετική διαδικασία του Συμβουλίου. Τα νομοθετικά έγγραφα έχουν ειδικό καθεστώ ε, υπό τον κανονισμό 10 49 και πρέπει να καθίστανται δημόσια από την ε, νομοθετική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γενικά ε, ένα υψηλότερο επίπεδο διαφάνειας αφορά τα νομοθετικά ε, έγγραφα από ότι τα άλλα διοικητικά έγγραφα για Παρ' όλα αυτά η δική μου έρευνα δεν αφορά συγκεκριμένο τομέα πολιτικής ή κάποια συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση. Οι φάκελοι που ερεύνησα υιοθετήθηκαν ε, με την, κατά τη συνήθεια νομοθετική διαδικασία, αλλά η έρευνά μου αφορά όλε τι νομοθετικέ διαδικασίε και οι συστάσει μου αφορούν όλε τι συζητήσει σε όλα τα προβασπαστικά όργανα, συμπεριλαμβανομένων των ε, ε προτάσεων ε, που αφορούν σε αφορολογικά ζητήματα όπω είναι η καταπολέμηση τη νομοποίηση παράνομων εσόδων. Όσον αφορά τα μη νομοθετικά έγγραφα, καταλαβαίνω ότι η ομάδα για, την, για τον κώδικα διοντολογία του Συμβουλίου ακολουθεί μια πιο συμβουλευτική ε, προσέγγιση που αφορούν πολιτικές ε, συμβουλές προκειμένου τα κράτη-μέλη να μπορούν να εκφράσουν μια πολιτική θέση και δεν είναι νομικά δεσμευτικά. Αυτές οι συζητήσεις δεν είναι νομοθετικές από τη φύση τους και γι' αυτό και δεν αφορούν την τωρινή μου έρευνα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι η δημόσια πρόσβαση σε αυτού του είδους τα έγγραφα ε, δεν μπορεί να χορηγηθεί με βάση τον κανονισμό 1049. Όπω γνωρίζετε, οι προηγούμενες επιτροπέ επιτροπές του Κοινοβουλίου για τη φορολογία ε, αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα όσον αφορά την πρόσβασή του σε έγγραφα του Συμβουλίου. Γενικά, όλα τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσφέρουν ε, πρόσβαση στα έγγραφά του εκτό αν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη εξαίρεση. Και αυτό αφορά και την ομάδα κώδικα δεοντολογίας για, για τη φορολόγηση των επιχειρήσεων του Συμβουλίου. Και το ελεγκτικό συνέδριο τόνισε ότι ο κανονισμό 1049 αποσκοπεί να εξασφαλίζεται η δημόσια πρόσβαση σε ολόκληρο το περιεχόμενο των εγγράφων του Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένου εμείς αυτή σε αυτή την περίπτωση της ταυτότητας εκείνων που κάνουν την ε, εκάστοτε πρόταση, των κρατών μελών δηλαδή. Και ενώ το ελεγκτικό συνέδριο επιμένει στα νομοθετικά έγγραφα, εξακολουθεί και τονίζει ότι ε, η δημόσια πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα αποτελούν το γενικό κανόνα, εκτός αν υπάρχουν συγκεκριμένες εξαιρέσεις, η ερμηνεία και η εφαρμογή των οποίων θα πρέπει να είναι αυστηρή. Κάποιες φορές έχω την αίσθηση όμως ότι το Συμβούλιο ακολουθεί την αντίθετη λογική, όπου η μη αποκάλυψη είναι ο βασικός κανόνας και η αποκάλυψη ή η πρόσβαση σε έγγραφα αποτελεί την εξαίρεση. Και για να ολοκληρώσω, Πρόεδρε, η υπηρεσία μου έχει αποστολή να ελέγχει τη διαφάνεια των, της δραστηριότητας και των διαδικασιών που ακολουθούνται στα θεσμικά όργανα και βάσει αυτών των ερευνών ε, ε, αξιολογώ ε, αν πρέπει ένα έγγραφο να δημοσιευθεί ή όχι. Τις περισσότερες φορές πράγματι και εγώ συμφωνώ όταν κάποιο θεσμικό όργανο αποφασίζει να μην δημοσιεύσει κάποιο έγγραφο. Κάποιες φορές όμως διαφωνώ. Δεν έχω, ξαναλέω, λάβει συγκεκριμένη καταγγελία, όμως θα αξιολογήσω άμεσα και σε βάθο οποιαδήποτε καταγγελία λάβω. Μπορούμε να λάβουμε ε, Καταγγελίε από ε, ευρωβουλευτές αλλά και επιτροπέ του Κοινοβουλίου. Και όλα τα παράπονα που πλέον λαμβάνουμε σχετικά με την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα ε, τα χειριζόμαστε γρήγορα και αποτελεσματικά εντό 40 ημερών. Όπω είπα, απουσία συγκεκριμένης καταγγελίας, οι παρατηρήσει μου προφανώ είναι γενικέ. Όμω, ε, αν έχετε ερωτήσεις είμαι στη διάθεσή σας και αν θέλετε βεβαίως υπάρχει και το επιτελείο μου, η υπηρεσία μου η οποία με μεγάλη χαρά θα σας βοηθήσει. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Οράιλη. Σας ευχαριστούμε για την αρχική σε αυτή παρέμβαση, για όλες τις προσπάθειες που έχετε καταβάλει και βλέπουμε ότι ε, ο βασικός λόγος για τον οποίο δεν λάβατε καταγγελίες όσον αφορά την ομάδα του κώδικα δεοντολογίας είναι ότι ε, πολλοί μπορεί να μην γνωρίζουν καν ότι υφίσταται μια τόσο ισχυρή ομάδα εργασίας στο Συμβούλιο και για την οποία υπάρχουν ε, ανησυχίες διαφάνειας. Ας ακούσουμε τώρα ερωτήσεις. Θα κινηθούμε ένα πέντε λεπτά. Μία ερώτηση θα πρέπει να λαμβάνει ένα λεπτό και ο υπόλοιπος χρόνος θα είναι για την απάντηση. Και εν συνεχεία, εφόσον μείνει χρόνος, μπορείτε να θέσετε και επιπλέον ερωτήσεις καλό καταρχάς τους εισηγητές να πάρουν το λόγο, καταρχάς τον κύριο Νίντερ Μάιερ εξ ονόματος ε, του ΕΛΚΑ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ κύριε Οράιλη που βρίσκεστε εδώ, ιδίω ε, έχοντας ακούσει ε, τον λόγο σας αυτό, την αρχική παρέμβαση που μας εμπνέει τόσο πολύ και πραγματικά λυπούμεθα που οι υπόλοιποι καλεσμένοι δεν βρίσκονται εδώ. Το ζήτημα της φορολόγησης μας έχει απασχολήσει εδώ στο Κοινοβούλιο για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί ουσιαστικά είναι ένας παράγοντας ο οποίος δεν είναι μόνο οικονομικός, αλλά και πολιτικός και κοινωνικός και πραγματικά πολύ συχνά μας προκαλεί αγανάκτηση το γεγονός ότι δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε σημαντική βελτίωση όσον αφορά τον φορολογικό τομέα και ακριβώς μέσω, του, μέσω της ομάδας του κώδικα δεντολογίας θα έπρεπε να προωθηθούν βελτιώσεις και πολύ φοβάμαι ότι αν η διαδικασία που ακολουθείται δεν ορθεί στον κώδικα δοντολογία, εκεί πέρα μπορεί να ξεκινήσουν και κάποιε κακέ συνήθειε όσον αφορά τη φορολογία. Πέρα από αυτό, θα ήθελα να ασχοληθώ γενικότερα με την στάση σα απέναντι στο Συμβούλιο πραγματικά βλέπουμε ότι το Κοινοβούλιο κινείται με έναν τρόπο πολύ πιο διαφανή, ενώ το Συμβούλιο λαμβάνει δράση με εντελώ διαφορετικό τρόπο. Ορισμένοι από την άλλη μπορεί να πούνε ότι το χαμηλό επίπεδο διαφάνεια στο Συμβούλιο δικαιολογείται από την απόπειρα επίτευξη συμβιβασμών. Άλλοι πάλι διαφωνούν με την προσέγγιση αυτή. Θα ήθελα δυνατόν να σα θέσω δύο-τρία ουσιώδη ερωτήματα για τα οποία θα ήθελα να είχα την προσωπική σας άποψη. Πρώτον, προωθείτε, μας είπατε όλο και περισσότερο, την διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρείτε πάντως ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η ενίσχυση της διαφάνειας οδηγεί σε πιο αποτελεσματική λήψη αποφάσεων ή μπορεί τελικά να είναι και αντιπαραγωγική. Δεύτερον, υπάρχει λόγος για τον οποίο το πρότυπο διαφάνειας είναι διαφορετικό ή μπορεί να είναι διαφορετικό με βάση το αν οι χώρες αποφασίζουν με ομοφωνία ή με ειδική πλειοψηφία. Και τρίτη ερώτηση. Μερικές φορές μας προκαλεί αγανάκτηση το γεγονός ότι υπάρχουν διάφορα νομοθετήματα, διάφορες προτάσεις που μπλοκάρονται στο Συμβούλιο χωρίς να γνωρίζουμε επίσημα ή ακόμα και ανεπίσημα τι ακριβώς συμβαίνει. Θεωρείτε ότι ένα υψηλότερο επίπεδο διαφάνειας θα μπορούσε να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στο Συμβούλιο προκειμένου να πάρει μια τελική τελικά απόφαση, να προωθήσει, να προωθήσει ένα φάκελο, να βρει συμβαστικέ λύσει ή ακόμα και να απορρίψει, αλλά τουλάχιστον να προχωρήσει. Κυρία Ράιλι, σας ευχαριστώ πολύ. Όντω τα ζητήματα τα οποία θίγεται είναι ζητήματα τα οποία μας έχουν υποβληθεί και στο παρελθόν και με τα οποία έχουμε ασχοληθεί και στα πλαίσια τη έρευνα στην οποία ανέφερα. Για δύο λόγους κάναμε την έρευνα αυτή όσον αφορά τη διαφάνεια του Συμβουλίου. Πρώτον, διότι κρίναμε και εμείς ότι υπήρχαν πολλά διαφορετικά επίπεδα διαφάνειας μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και δεύτερον γιατί το Συμβούλιο ως θεσμικό όργανο είναι περισσότερο αδιαφανές και λιγότερο γνωστό στους Ευρωπαίους πολίτες, μολονότι σε αυτό συμμετέχουν κρατικοί φορείς, αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Και ξέρετε ότι ε, πολλοί δεν συνειδητοποιούν τελικά ότι στα πλαίσια του Συμβουλίου είναι οι ίδιες οι κυβερνήσεις οι οποίες συνομοθετούν συνεργαζόμενες με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου διάβασαν επιστημονικά άρθρο σε σχέση με την διαφάνεια και τη στάση του Συμβουλίου στους τριμερούς διαλόγου, διαλόγους και ακριβώς θίγεται και το ζήτημα αυτό μεταξύ λογοδοσίας και αποτελεσματικότητας στα πλαίσια των τριμερών διαλόγων. Ο συντάκτης του επιστημονικού αυτού άρθρου εξέτασε τη στάση του Συμβουλίου τα τελευταία δέκα χρόνια και κατέληξε στο συμπέρασμα τελικά ότι η διαφάνεια εξαρτάται από το θέμα το οποίο τίθεται κάθε φορά προς συζήτηση. Για παράδειγμα, για, τα νομοθετη... για τις νομοθετικές εκείνες προτάσεις όπου διακυβεύονται πολύ σημαντικά χρηματικά ποσά τότε είναι περιορισμένη η διαφάνεια. Ενώ για ζητήματα τα οποία, μάλλον για ζητήματα τα οποία είναι πολιτικά ευαίσθητα και για αυτά είναι μειωμένη διαφάνεια. Από την άλλη ζητήματα τα οποία δεν έχουν μια κάποια πολιτική ευαισθησία, για παράδειγμα κοινωνικά μέτρα, περιβάλλον κτλ τότε στις περιπτώσεις αυτές το επίπεδο διαφάνειας είναι πολύ υψηλότερο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι οι πολιτικές ευαισθησίες αυτές οι οποίες καθορίζουν το επίπεδο διαφάνειας. Αυτό το οποίο μας έχει απασχολήσει εμά τη έρευνά μας είναι να δούμε τι θα έπρεπε να γίνεται από νομικής πλευράς, αλλά και τι θα έπρεπε να γίνεται σύμφωνα μετά όσο επιτάσσουν οι ίδιες οι συνθήκες. Το ότι δηλαδή ο Ευρωπαίο πολίτης θα πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένος και ότι θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε έγγραφα, σε συζητήσει αν το αποφασίσει αυτό. Από την άλλη, υπάρχουν ορισμένοι που λένε, αυτό το οποίο αναφέρατε κι εσεί, ότι ενδεχομένω αν είναι υπερβολική η διαφάνεια, τότε δύσκολα να επιτυγχάνονται και συμβιβασμοί. Αλλά ξέρετε ότι όλες οι νομοθεσίες, ακόμα και ο καονισμός 1049, προβλέπουν ένα τέτοιο περιθώριο ευελιξίας. Δηλαδή, δίδεται τη δυνατότητα ακόμα και με τον κανονισμό αυτό να γίνεται μια ανταλλαγή απόψεων πιο μυστική προκειμένου να μπορεί τελικά να καταλήξει πιο εύκολα ο νομοθέτης ή εμπλεκόμενη σε ένα συμβιβασμό και προφανώς εμείς δεν το αμφισβητούμε αυτό σε καμία περίπτωση. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να προβλέπετε και αυτή η δυνατότητα αλλά σε σχέση με ένα πιο συγκεκριμένο ζήτημα, δηλαδή να γνωρίσουμε ακριβώς ποια είναι η τοποθέτηση των κρατών μελών, των κατοχωρών, της Ισπανίας, οποιασδήποτε άλλης χώρας. Για το ζήτημα αυτό, εμείς αυτό το οποίο ζητάμε δεν είναι να κοινωνοποιείται άμεσα η τοποθέτηση μιας χώρας στα πλαίσια της Κορεπέρη σε μια ομάδα εργασίας, αλλά να καταγράφεται, να καταγράφεται. Επομένως, να είναι δυνατό κάποιος να γνωρίζει, εφόσον το επιθυμεί, ακόμα και να κάνει μια ιστορική αναδρομή στην στάση που έχουν κρατήσει ορισμένες χώρες. Τώρα, η νομολογία του δικαστηρίου στην οποία αναφέρθηκα όσον αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα, λέει ότι δεν θα πρέπει να προβλέπεται καμία απόλυτο εξαίρεση. Εφόσον έχουν τηρηθεί πρακτικά, θα πρέπει αυτά να κοινοποιούνται. Αυτό το οποίο ανακαλύψαμε και το οποίο βέβαια δεν μας προκαλεί μάλλον έκπληξη βλέποντας τι κάνει το Συμβούλιο και η επιμέρους ομάδα εργασίας και η ΚΟΡΕΠΕΡ είναι ότι σταμάτησαν μετά την απόφαση αυτού του δικαστηρίου να καταγράφουν τις τοποθετήσεις των κρατών μελών. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ε, αν δεν καταγράφεται η τοποθέτηση αυτή δεν είναι προσβάσιμη από κανένα, δεν υφίσταται πολύ απλά. Οι δύο βασικές λοιπόν ε, συστάσεις ή μάλλον η βασική σύσταση που έκανα προς το Συμβούλιο είναι ότι θα πρέπει η τοποθέτηση των κρατών μελών, αν μη τι άλλο, να καταγράφεται. Βέβαια τα πράγματα δεν είναι απόλυτα, τίθενται όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία θίξατε, αλλά θα πρέπει να εξισορροπήσουμε τον πιθανό κίνδυνο στον οποίο αναφερθήκατε με τον υφιστάμενο κίνδυνο τον οποίο ζούμε και βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Το ότι υπάρχουν όλοι και περισσότεροι πολίτε οι οποίοι δεν εμπιστεύονται πλέον τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση που αντιμετωπίζουν το Συμβούλιο ω ε, μη εκλεγμένου γραφειοκράτε οι οποίοι αποφασίζουν για την τύχη του. Ευχαριστώ. Ε, από και Δημοκράτες, ο συνεισηγητής κύριο Κόφωτο. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ και σας κυρία Ορέιλη. Εξαιρετική και άκρως ενδιαφέρουσα η παρουσίαση. Ενησυχώ πάρα πολύ ακούγοντα σα να λέτε ότι από ό,τι φαίνεται ε, η νοοτροπία του Συμβουλίου είναι μάλλον η μία αποκάλυψη παρά η δημοσιοποίηση. Κανονικά το αντίθετο θα πρέπει να συμβαίνει. Εμείς είμαστε άμεσα εκλεγμένοι από τους Ευρωπαίους πολίτες εδώ στο Κοινοβούλιο και έχουμε κάθε δημοκρατικό δικαίωμα να γνωρίζουμε τι κάνουν οι εκπροσωποί μας. Ο λαός δηλαδή θέλει να γνωρίζει τι κάνουμε εμείς και αντίστοιχα και τι κάνουν κυβερνήσεις στο Συμβούλιο. Ίσως ε, έτσι ενισχυθεί και η εμπιστοσύνη και στα μάτια των πολιτών, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Σας ευχαριστώ για τις ε, απαντήσεις σας, Τι διάβασα πολύ προσεκτικά. Λέτε λοιπόν στη γραπτή σας απάντηση ότι το Συμβούλιο δεν κατάφερε να ε, τηρήσει την προθεσμία της 9 η Μαου και δεν θα απαντήσει πριν τον Ιούλιο. Αυτή είναι μια προθεσμία που έθεσαν μόνοι του Και τι θα γίνει αν δεν σεβαστούν για τη νέα προθεσμία. Εσεί ω διαμεσολαβήτρια τι προτίθεστε να πράξετε. Και στη συνέχεια λέτε επίση ότι, και μάλιστα ξεκάθαρα στα συμπεράσματά σα, ότι, και σα παραθέτω στη γραπτή σα απάντηση, το Συμβούλιο, οι ομάδε εργασίες του Συμβουλίου υπολείπονται στα όσα αναμένουμε από το Συμβούλιο για την νομοθετική διαφάνεια. Πράγμα που συνιστά ε, κακή πρακτική και κακοδιαχείριση. Αυτή ήταν η δική σας ε, λοιπόν παράθεση. Έχετε διαπιστώσει έκτοτε αλλαγές ε, στις εργασίες του Συμβουλίου και στις μεθόδους από τότε που αρχίσατε τις ερευνές σας και έχετε δεχτεί καμία κρούση από το Συμβούλιο ε, για το κατά πόσο θα σταματήσουν ε, αυτή την κρυψίνο πρακτική και για την ομάδα επαφών για τη φορολόγηση των επιχειρήσεων. Κοιτάξτε, είμαστε σε μία ενιαία αγορά εσωτερική και τα φορολογικά ζητήματα, όπως αυτές οι επιζήμιες φορολογικές πρακτικές, ανησυχούν πάρα πολύ τον κόσμο ε, σε μια εσωτερική αγορά με τις τέσσερις γνωστές ελευθερίες, στην κυκλοφορία των προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων. Δεν μπορεί μια ομάδα να, έτσι, να δρά με ένα τέτοιο μυστικοπαθή τρόπο για θέματα φορολογικά. Δεν καταπατούν την εντολή τους για την υποχρέωση που έχουν να υπηρετούν τους ευρωπαϊκούς λαούς και τις χώρες. Απάντηση. Εμείς τους δώσαμε μια προθεσμία 9 Μαΐου που κατά σύμπτωση είναι και η επέτειος της η μέρα της Ευρώπης. Είναι εντελώς τυχαίο, δεν υπήρχε καμία πρόθεση. Ε, είπαμε ότι μπορούσε να παρατεθεί, αλλά είπαμε επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα και επειδή καλπάζει ε, ο χρόνος και φτάνουμε στο 2019, δεν πρόκειται να δεχθούμε ε, και άλλη παράταση. Πριν από λίγες εβδομάδες ήρθαν και μας είπαν αν θέλουμε παράταση και εμείς είπαμε όχι. Οπότε νομίζω αυτή την εβδομάδα θα κάνω μια ειδική έκθεση στο Κοινοβούλιο και θα ζητώ την υποστήριξη του Κοινοβουλίου γι' αυτό. Θα είναι η δεύτερη έκθεση προς το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της θητείας μου. Είναι σοβαρό το θέμα και καταδεικνύει το δημόσιο ενδιαφέρον που διαπιστώνουμε κι εμείς. Βελτιώσεις, έχουν γίνει κάποιες βελτιώσεις. Έκανα και μια ακόμα σύσταση Ε, ε, έτσι συστηματικά ε, χαρακτηρίζουν διαβαθμισμένα τα έγγραφα. Γράφει «limité» στα γαλλικά. Και στη συνέχεια πάνω από 80% των εγγράφων αυτών από την πάροδο κάποιου χρονικού διαστήματος δημοσιεύονται. Οπότε για ποιο λόγο να είναι διαβαθμισμένα και Υπάρχουν κάποια έγγραφα που είναι τελείως ανώδυνα και ε, χωρίς καμία ιδιαίτερη ευαισθησία. Γιατί τα χαρακτηρίζεις ε, διαβαθμισμένα, ενώ πρέπει να δημοσιεύονται από την αρχή. Και βάσει του κανονισμού 1049 εδώ δεν πρόκειται περί εξαίρεσης. Και στην περασμένη επιτροπή είχα έρθει, τάξη 2, και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η συζήτηση και τα σκληρά λόγια που άκουσα και από την πλευρά του Συμβουλίου. Η διαφάνεια είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί όταν βγαίνουν αυτά στον αέρα και αποκαλύπτονται διάφορα Panama Papers και άλλα, ενδιαφέρεται ο κόσμος και βλέπει και τι γίνεται εδώ στο Κοινοβούλιο, σε αυτή την Επιτροπή. Χρειάζεται συμμαχία εδώ δυνάμεων για να αλλάξουν αυτά τα ε, ε, θέματα και καταστάσεις. Ο κύριος Ρωσάτη από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Οράλη, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ σήμερα το απόγευμα και για την παρουσίασή σας. Με χαρά άκουσα ότι η υπηρεσία σας και το Κοινοβούλιο τάσσονται υπέρ της μεγαλύτερης διαφάνειας να εξασφαλίζεται η πρόσβαση των Ευρωπαίων πολιτών σε πληροφορίες και αυτό αποτελεί μια θετική πλατφόρμα για τη συνεργασία μας. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πώς μπορείτε εσείς να μας βοηθήσετε ώστε να έχουμε μεγαλύτερη πρόσβαση σε ευαίσθητα, διαβαθμισμένα ε, ή προστατευόμενα στοιχεία τα οποία δεν μας δίνει το Συμβούλιο. Σε προηγούμενες εξεταστικές επιτροπές, μάλλον στην Επιτροπή Πάνα, ζητήσαμε μια σειρά από έγγραφα και αυτό που λάβαμε σε πολλές περιπτώσεις ήταν απλώς λευκές σελίδες ή σελίδες από τις οποίες είχαν διαγραφεί τα σημαντικότερα και τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία. Αυτό βεβαίως ε, έδωσε την ε, εντύπωση ε, μιας ιδιαίτερης μεταχείρισης που θα μπορούσε κανείς να την, χρησιμοποιήσει αποκαλέσει και κρυψίνο. Ε, στην συνεργασία μας μεταξύ Κοινοβουλίου δηλαδή και Δημοσιογραφήτρια θα μπορούσαμε ίσως να καταλήξουμε στην έκδοση συστάσεων για το πώς πρέπει να, να γίνεται ο χειρισμός φορολογικών πληροφοριών ή αποφάσει φορολογικού χαρακτήρα που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη, πώς αυτές θα δημοσιεύονται ή πώ μπορούμε να χειριστούμε ζητήματα που σχετίζονται με τον ε, τελικό δικαιούχο μιας απόφαση ή ωφελούμενο από μια, από μια φορολογική απόφαση. Πώς μπορούμε δηλαδή με άλλα λόγια να συνεργαστούμε καλύτερα προκειμένου να ενισχύσουμε τη διαφάνεια σε αυτούς τους τομείς που είναι τόσο σημαντικοί για μας, για σας και για τους πολίτες μας. Δεύτερη ερώτηση. Το Φεβρουάριο του 2018 ξεκινήσατε μια ταχεία διαδικασία σε σχέση με την ε, επεξεργασία καταγγελιών που σχετίζονται με την πρόσβαση σε έγγραφα. Μπορείτε να μας δώσετε μια κάποια προκαταρκτική ε, αξιολόγηση για το αν έχετε επιτύχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ίσως είναι νωρί, το καταλαβαίνω, αλλά ίσως θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποια πρώτα, κάποιες πρώτες ε, παρατηρήσεις στις οποίες έχετε καταλήξει. Ευχαριστώ πολύ. Με βάση το καθεστώ ε, διαφάνεια που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα θεσμικά όργανα μπορούν πραγματικά να ανοιγοκλίνουν τη βρύση αυτή όσον αφορά την ε, έκδοση και τη δημοσίευση συγκεκριμένων αρχείων εγγράφων. Μπορούν τα ίδια να αποφασίσουν αν αυτό θα το δημοσιεύσω ή όχι. Στη συνέχεια, βεβαίω, αν κάποιο δεν είναι ευχαριστημένο με την απόφαση του θεσμικού έργου, μπορεί να προσφύγει σε μένα ή στα δικαστήρια. Ο καλύτερο τρόπο, λοιπόν, ε, που μπορώ εγώ να χειριστώ μια τέτοια απόφαση είναι να λάβω συγκεκριμένη καταγγελία. Αν δεν έχετε δηλαδή πρόσβαση σε συγκεκριμένο έγγραφο ή σε συγκεκριμένο σύνολο εγγράφων και θεωρείτε ότι αυτό δεν είναι σωστό ή υπάρχουν έγγραφα από τα οποία έχουν διαγραφεί συγκεκριμένα στοιχεία που σα ενδιέφεραν, το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε είναι για, για εμένα να μου, δώσετε, να μου κάνετε μια καταγγελία ε, επίσημη ώστε να μπορώ να ξεκινήσω έρευνα. Προφανώς βεβαίω, ε, κανένα θεσμικό όργανο δεν είναι υποχρεωμένο να ακολουθήσει τη δική μου σύσταση αν και στις περισσότερες περιπτώσεις το κάνουν. Αυτό που μπορώ να κάνω όμως είναι ε, να ενθαρρύνω αυτό το, το, εν λόγω θεσμικό όργανο μέσω της πίεσης που θα ασκήσω εγώ ε, προκειμένου να προχωρήσει στη δημοσίευση αυτού του εγγράφου που σα ενδιαφέρει. Αν δηλαδή μπορείτε, μπορώ εγώ να σας βοηθήσω, μπορείτε και εσείς να με βοηθήσετε. Αυτό σας λέω, να μου κάνετε μια καταγγελία για να μπορέσω να ξεκινήσω τη διαδικασία. Ευρύτερα τώρα, υπάρχει ένα, επίτροπο, ένα δίκτυο ε, ε ανθρώπων που σχετίζονται με την προσβασιμότητα συγκεκριμένων πληροφοριών που εξετάζουν βεβαίως ε, τι υποθέσεις που σχετίζονται με αυτά τα θέματα, τη πρόσβαση σε έγγραφα και σε πληροφορίε. Αυτό ε, ε, είναι, είναι ένα δίκτυο επιτρόπων που, που ασχολούνται ακριβώ με αυτό το θέμα και αυτό μας βοηθά να αξιολογούμε ε, το πού πηγαίνουν τα πράγματα στα φορολογικά ζητήματα. Για την ταχεία αυτή διαδικασία ε, ευτυχώς μέχρι στιγμής τα πράγματα πάνε καλά. Αυτό που κάναμε είναι το εξής. Αντιληφθήκαμε ότι οι καταγγελίες για τη διαφάνεια είχαν ένα διαφορετικό χαρακτήρα από τις άλλες καταγγελίες. Γιατί έως ότου λάβουμε εμεί την καταγγελία και μπορέσουμε να την επεξεργαστούμε, το Συμβούλιο έχει ήδη καταλήξει ε, στην τελική του απόφαση χωρίς να μπορούμε εμείς να παρέμβουμε στη διαδικασία. Ε, στο παρελθόν δηλαδή ερχόμαστε και κάναμε μια αναδρομική δουλειά. Ζητούσαμε να δημοσιεύσουν πληροφορίε, οποίες όμως δεν, δεν, οι οποίες όμως δεν ήταν χρήσιμε ούτε ενδιαφέρουσε πια γιατί το θέμα είχε ολοκληρωθεί. Από αυτή την άποψη λοιπόν το σημαντικό είναι να λάβουμε καταγγελία για να μπορέσουμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε τη διαδικασία και να λάβουμε απάντηση γιατί, γιατί δεν έχουν δημοσιευθεί συγκεκριμένε πληροφορίε ακόμα. Στι περισσότερε περιπτώσει, λοιπόν, η ταχεία διαδικασία φαίνεται ότι φέρνει καλύτερα αποτελέσματα, αν και όπω είπατε και εσεί είναι αρκετά νωρί για να καταλήξουμε σε οριστικά απο, ε, πορίσματα. Ευχαριστούμε. Ο κύριο Σάρντ Κόν το λόγο εξ των Σοσιαλιστών. Θα μιλήσω γερμανικά, κύριε Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και σας κυρία Ωραίλη για την παρουσία σας. Και πραγματικά είναι καλό να σας βλέπουμε στο πλευρό μας και να γνωρίζουμε ότι μας συμπαρίσσεστε στην συνεργασία με το Συμβούλιο, όχι μόνο στην απαλλαγή για τον προπολογισμό, το έζησα στην Επιτροπή Ελέγχου του Προεπολογισμού, αλλά και στην ομάδα για τον κώδικα δεοντολογίας. Υπάρχουν πολλά στραβά Εσείς έχετε περισσότερες αρμοδιότητες και εξουσίες να ζητάτε έγγραφα από ότι εμείς ως Εξεταστική Επιτροπή, Ειδική Επιτροπή του Κοινοβουλίου. Εσείς αυτό το θεωρείτε θεμητό και δικαιολογημένο ή πιστεύετε ε, ότι θα πρέπει να κάνουμε και εμείς το ίδιο, να έχουμε περισσότερες αρμοδιότητες και να ζητούμε τα έγγραφα, ακόμα και αν πολλές φορές έχουμε ε, επικαλύψεις. Ε, γνωρίζω ότι αυτό το θέμα έχει ζητηθεί πολύ και στην περασμένη Επιτροπή τα θίγει αυτό το θέμα, έχω την ε, αίσθηση. Και αυτό πραγματικά επανέρχεται ξανά και ξανά στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, ιδιαίτερα όταν ε, έχουν ένα έργο ευαίσθητο και ερευνητικό, όπως το έργο με το οποίο έχετε επιφορτιστεί εσείς αυτό το καιρό. Νομίζω εσείς το είπατε, Πρόεδρε, ότι οι, τα θεσμικά όργανα κατά τη συνθήκη θα πρέπει να εργάζονται σε, σε ειλικρινή ή αγαστή συνεργασία, δεν απατώ με ειλικρινή συνεργασία φέρει η συνθήκη. Αλλά απαντώντας και σε προηγούμενη ερώτηση, είπα ότι σε ό,τι αφορά το δικό μου έργο, αυτό που θα με βοηθάει είναι να γίνονται καταγγελίες, να έρχονται καταγγελίες για να ε, μπορώ να προχωρώ, να το ερευνώ και να απευθύνομαι στο Συμβούλιο. Και όχι αυτεπάγγελτα, χρειάζομαι καταγγελίες για να το κάνω αυτό. Αλλά και το Κοινοβούλιο έχει τη δική του δουλειά και την έρευνα να κάνει. Ως πολίτης, ε, βέβαια δεν είμαι ε, αρμόδια για τη φορολογικά, ως πολίτης ε, σοκαρίστηκα ε, ε, μετά από αυτά που διάβασα ότι ετησίως η Ευρωπαϊκή Ένωση χάνει ένα τρισεκατομμύριο ευρώ από φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή και οι περισσότεροι πολίτες ε, όταν ακούν για φοροδιαφυγή δεν το αντιλαμβάνονται, δεν το βλέπουν σε αυτή την τάξη μεγέθους. Σκέφτονται το, τον τόπιο δισεκατομμυρίουχο ή πολυεκατομμυρίουχο και πώς κλέβει την εφορία ή πώς γλιτώνει την εφορία. Ευχαριστούμε. Νίλ Στόλβαρτς, τώρα από του ελευθέρους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν κάθομαι στη συνήθι μου θέση. Συχνά όταν προσπαθώ να περιγράψω τι κάνουμε εμείς στα πλαίσια της αποφυγής φοροδιαφυγής είναι το αντίστροφο δίλημα που έχει ένας φυλακισμένος. Γιατί ξέρετε ότι πολλές φορές οι εγκληματίες συνεργάζονται γιατί πιστεύουν ότι μπορούν κάτι να κερδίσουν από αυτό. Στην περίπτωση αυτή, στο αντίστροφο αν θέλετε σενάριο, δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή για εγκληματίες, αλλά για ένα θεσμικό όργανο, το οποίο ουσιαστικά κρατεί μια εντελώς διαφορετική στάση. κρατάει μια στάση η οποία τελικά γυρίζει λίγο μπούμεραν για το ίδιο, γιατί δημιουργεί μια αρνητική εικόνα για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι το θεσμικό αυτό όργανο με τη στάση του τελικά βάλει κατά της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζημιώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώς εμείς αυτό θα πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα προς τα έξω αλλά δυστυχώς από ό,τι φαίνεται δεν έχουμε την πυγμή προκειμένου να καταδικάσουμε τη στάση αυτή του Συμβουλίου. Χρειαζόμαστε λοιπόν τη δική σας συνδρομή. Πολύ ωραία. Συμφωνώ με το γενικότερο σχόλιο που κάνατε. Όντως, Κάθε δύο-τρεις εβδομάδες ακούμε έναν Ευρωπαίο ηγέτη ο οποίος αναφέρεται στο Συμβούλιο λέγοντας ότι υπάρχει ένα τεράστιο δημοκρατικό έλλειμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι αυτό τελικά συμβάλλει σε φαινόμενα όπως το Brexit κτλ. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε λίγο και τις επιπτώσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή αλλά και την καθημερινή, τον καθημερινό τρόπο με τον οποίο εργάζεται το Συμβούλιο αλλά βέβαια και το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να ασχοληθεί με αυτό. Καθότι ε, πλησιάζουν ε, οι ευρωπαϊκές εκλογές, βλέπουμε ότι αυξάνονται οι συζητήσεις που γίνονται παντού για το μέλλον της Ευρώπης. Νομίζω όμως ότι πέρα από τα λόγια θα πρέπει να περάσουμε σε κάτι λίγο πιο χειροπιαστό και νομίζω ότι και αυτή η πτυχή που θίξατε εσείς όντως θα πρέπει να τονιστεί. Τώρα, η όλη μυστικοπάθεια που μπορεί να υπάρχει, η στάση αυτή του απόρριτου στα πλαίσια του Συμβουλίου δεν νομίζω ποτέ ότι θα μπορούσε σε μια χώρα, σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο, να τεθεί μια ερώτηση, σε μια εκπομπή για παράδειγμα, σε έναν πολιτικό, από έναν πολίτη, από έναν δημοσιογράφο, ο οποίο να πει μπορείτε να αφαιρθείτε λίγο περισσότερο στην τάδε νομοθεσία, να μα δώσετε περισσότερα στοιχεία και αυτό να απαντήσει όχι, δεν αποκαλύπτω στοιχεία. Θα ήταν ε, αδιανόητο αυτό σε εθνικό επίπεδο, παρά αυτά το βλέπουμε να γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όντω. Ε, αυτό θα πρέπει να μας ανησυχήσει και θα πρέπει να το δούμε και από την οπτική γωνία της πολιτικής οριμότητος. Το Συμβούλιο, αντί να στρουθοκαμαλίζει, θα πρέπει πραγματικά να εμπιστεύεται περισσότερο τους πολίτες και αν μη τι άλλο να εξηγήσει προς τα έξω, προς τους πολίτες δηλαδή, ότι πολλές φορές τα πλαίσια της δημοκρατίας ή της λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης καλείται ή οφείλει να κάνει συμβασμούς. Νομίζω ότι θα ήταν θετικό αυτό να το πει προς τα έξω το Συμβούλιο ανοιχτά. Ευχαριστούμε. Εξ ονόματος των Πρασίνων, ο Μαξ Άντερσον έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ακούσαμε τόσες πολλές καλές ερωτήσεις και λάβαμε και πολύ καλές απαντήσεις. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι υπάρχουν ακόμα κάποια ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να θέσουμε. Πρώτον, δεν ξέρω αν έχετε λάβει μια κάποια εξήγηση από το Συμβούλιο. Για ποιο λόγο τελικά δεν απάντησαν στη δική σας την επιστολή μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, μέχρι την 9η Μαΐου δηλαδή. Έχετε καθόλου πληροφορίες για τις διαφορετικές στάσεις των κρατών μελών όσον αφορά αυτή την επιστολή. Και κάτι ακόμα. Ένα ακόμα σημαντικό ζήτημα που έχει να κάνει με την διαφάνεια της νομοθετικής διαδικασίας και πιο συγκεκριμένα το ζήτημα της διαφάνειας στα πλαίσια των τριμερών διαλόγων. Ξέρετε ότι έχουμε πάλι απόφαση του δικαστηρίου στην υπόθεση Καπιτώνη όσον αφορά την διαφάνεια στους τριμερείς διαλόγους. Μετά την απόφαση αυτή του δικαστηρίου, εσείς ποια δράση θα αναλάβετε προκειμένου και στα πλαίσια των τριμερών διαλόγων υπάρχει ένα πλήρες καθεστώς διαφάνειας σύμφωνα με όλα αυτά τα οποία ζητά το δικαστήριο. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Το Συμβούλιο πολύ απλά μου απάντησε ότι δεν είχαν το χρόνο να απαντήσουν εγκαίρως στην επιστολή μου. Δεν δώσανε συγκεκριμένα στοιχεία, ούτε κάποια πιο βαθιστόχαστη αιτιολόγηση. Σε σχέση με τους τριμερείς διαλόγους, όντως διεξήγαμε και για αυτούς μια έρευνα και προχωρήσαμε σε συγκεκριμένες συστάσεις. Την εποχή εκείνη το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο περίμεναν την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τη δημοσίευση αυτών των εγγράφων με τις τέσσερις στήλε που χρησιμοποιούνται στους τριμερείς διαλόγους. Και πριν από τρεις-τέσσερις εβδομάδες βγήκε αυτή η απόφαση του Δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία το δικαστήριο θεωρεί ότι δεν υπάρχουν λόγοι που να επαγορεύουν τη μυστικότητα του εγγράφου αυτού σύμφωνα με τον κανονισμό 1049. Η δικιά μου σύσταση ήταν ότι το έγγραφο αυτό θα πρέπει αν μη τι άλλο να δημοσιεύεται μετά το τέλος του τριμερούς διαλόγου. Μετά λοιπόν την επίσημη αυτή απόφαση του δικαστηρίου θα έλθουμε πάλι σε επαφή με τα θεσμικά όργανα για να δούμε τελικά πώς θα την εφαρμόσουν Ξέρετε ότι ε, ένα μέρος των πληροφοριών ήδη κοινοποιείται. Μπορούν να γνωρίζουν αυτή τη στιγμή οι πολίτες περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν πότε γίνονται τριμερείς διάλογοι ή με ποια ζητήματα καταπιάνονται. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή, εφόσον έχουμε την απόφαση την επίσημη του δικαστηρίου, μπορούμε να ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση για την ίδια τη δημοσίευση των εγγράφων αυτών και για την εφαρμογή των συστάσεων που έχω κάνει. <clears throat> Ο κύριο Σίρδεβαν, ευχαριστούμε κύριε Οράιλ για την παρουσίαση. Είπατε στι απαντήσει σα ότι ο κανονισμό εξασφαλίζει την πρόσβαση του κοινού σε ολόκληρο το περιεχόμενο των εγγράφων συμπεριλαμβανομένων των θέσεων των κρατών μελών. Και σε αυτή την επιτροπή, το έχουμε ξαναπεί και άλλε φορέ, ε, πολλές φορές έχουμε δεχτεί άρνηση από το Συμβούλιο να μας παράσχει πρόσβαση σε έγγραφα και πληροφορίε που θα, που θα αποκάλυπταν τη θέση των κρατών μελών και ε, στην έκθεσή σα του Φεβρουαρίου ε, προκύπτει ότι πολλές φορές δεν καταγράφονται καν αυτές οι θέσεις. Και τα πορίσματα αυτά ε, δείχνουν ότι το Συμβούλιο παραβιάζει το άρθρο 50 του κανονισμού που ορίζει ότι τα θεσμικά όργανα πρέπει να αναπτύσσουν καλέ ε, διοικητικέ διαδικασίε ώστε να εξασφαλίζεται το δικαίωμα πρόσβαση των πολιτών στι πληροφορίε. Χαιρετίζουμε τα πορίσματά σα σχετικά με την νομοθετική διαδικασία του Συμβουλίου. Σημειώνουμε όμω ότι το Συμβούλιο δεν ανταποκρίθηκε στην υποχρέωσή του να απαντήσει εντό προσθεσμίες Έχετε ε, σκοπό να δώσετε συνέχεια σε σχέση με τις σύστασή σας ότι τα, ότι τα κράτη-μέλη και οι θέσεις τους θα πρέπει να καταγράφονται στα έγγραφα. Θέλετε να, ε, σκοπεύετε να κάνετε κάποια έρευνα για αυτό το θέμα και υπάρχει κάποια γνώμη από την πλευρά σας σχετικά με πιθανή δικαστική δράση που μπορεί να αναλυφθεί σε περίπτωση που διαπιστώνεται κακή πλημελής διοικητική ε, πρακτική. Προφανώς μπορείτε να, μπορεί κανείς να προσφύγει ε, στο δικαστήριο σε περίπτωση που δεχτεί άρνηση πρόσβαση σε έγγραφα. Είναι κάτι που το οποίο το έχουν κάνει στο παρελθόν οι ευρωβουλευτές. Αυτό που κάνω εγώ είναι μια πολύ, ένα πολύ μεγάλο βήμα για την υπηρεσία μου η εκπόνηση αυτής της ειδική έκθεσης προς το Κοινοβούλιο και το αίτημά μου προς το Κοινοβούλιο να με υποστηρίξει. Όπως είπα είναι μόλις η δεύτερη φορά από το 2013 όταν ανέλαβα τα καθήκοντά μου που συντάσσω μια τέτοια ειδική έκθεση και πρόκειται για μια, η πρώτη μάλιστα ειδική έκθεση αποτελούσε συνέχεια που, που έδωσα σε, διαδικασία του προκατόχου μου. Ε, πρέπει λοιπόν να τονίσω ε, ότι ε, ε, ποιος μπλοκάρει ε, θέματα ή φακέλους στην, στο Συμβούλιο. Ε, βεβαίως αυτό το θέμα είναι πολιτικά ευαίσθητο, αλλά δεδομένου του χαρακτήρα της φορολογίας, των φορολογικών θεμάτων και επειδή μιλάμε για τρισεκατομμύρια, όχι απλά για δισεκατομμύρια, είναι προφανώς, προφανές ότι υπάρχει δημόσιο συμφέρον εδώ και εδώ το lobbying, η άσκηση πίεσης από συγκεκριμένε ομάδες παίζει ρόλο. Και αυτό πρέπει να, σε αυτό πρέπει να, να, να, φωτιστεί περισσότερο αυτό το θέμα. Και αυτό το, και το έργο μου επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στην, στο να φωτιστεί αυτό, αυτό το ζήτημα του lobbying στην Κομισιόν και στο Συμβούλιο. Και βεβαίως έχω μιλήσει και με διαμεσολαβητές ε, στα κράτη-μέλη για να ε, δω πώς ακριβώς ρυθμίζεται το θέμα αυτό νομοθετικά στα κράτη-μέλη. Παρ' όλα αυτά πρέπει να σας πω ότι ε, πρόκειται για έναν τομέα πολιτικής όπου ασκείται η μεγαλύτερη πίεση σε σύγκριση με όλους τους άλλους τομείς και στα κράτη-μέλη. Είναι κάτι υπαρκτό και είναι προφανές ότι αυτό επηρεάζει και τον τρόπο με τον οποίο σας έχουν μεταχειριστεί ως Επιτροπή. Αυτή όμως, αυτό ακριβώς θα είναι όμως και το θέμα της ε, ειδική έκθεσης που θα δημοσιεύσω αργότερα εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Ευχαριστώ κυρία Κάπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ε, κυρία Οράιλ για την ενδιαφέρουσα ε, παρουσίασή σας. Ήμουν μέλος της Επιτροπής ΠΑΝΑ και ε, όπως μια και λέτε ότι η καταγγελία θα μπορούσε να σας βοηθήσει ε, κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων σας προκειμένου να μπορείτε να στρέφεστε προς το Συμβούλιο ε, θυμήθηκα ε, αυτό που είχαμε αντιμετωπίσει πόσο δύσκολα ήταν τα πράγματα σε σχέση με την πρόσβασή μας σε, κατά την εξέταση των υποθέσεων της Επιτροπής ΠΑΝΑ. Ίσως θα μπορούσατε να μας είχατε βοηθήσει τότε αν είχαμε κάνει τέτοιου καταγγελίε καταγγελίες προς Θέλω να πω το εξή, ότι ε, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση που το Συμβούλιο δεν απάντησε μέχρι τις 9 Μαΐου στις συστάσεις σας. Ε, νομίζω ότι τους δώσατε αρκετό χρόνο για να απαντήσουν. Γι' αυτό και θα ήθελα να σας ρωτήσω, έχετε ένα γενικό περίγραμμα για το τι ακριβώς θα περιλαμβάνει αυτή η ειδική έκθεση, τι θα ζητάτε μέσα από αυτή την ειδική έκθεση από το Συμβούλιο. Δεύτερο, για την ομάδα για τον κώδικα διοντολογίας και στις συστάσεις της Επιτροπής Πάνα ε, είχαμε τονίσει ότι όταν μιλούμε για παράδειγμα για τον κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις μη συνεργάσιμες χώρες ε, υπάρχει μια έλλειψη, ένα έλλειμμα ε, διαφάνειας όσον αφορά την κατάρτιση αυτού του καταλόγου και όπως είπατε και εσείς, ε, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο χώρο, κάποια χώρα προστίθεται ή αφαιρείται από αυτόν τον ε, κατάλογο. Υπάρχει πολύ μεγάλη αδιαφάνεια. Γι' αυτό και θέλω να σας ρωτήσω, μήπως ε, έχετε συγκεκριμένες συστάσεις και προς αυτήν τη συγκεκριμένη ομάδα για τη φορολόγηση των επιχειρήσεων, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη καταγγελία για το πώς θα μπορούσε το έργο αυτής της ομάδας να καταστεί πιο διαφανές πώς θα μπορούσε να διαρθρωθεί με έναν πιο ε, δομημένο τρόπο η πρόσβαση στις πληροφορίες, πώς θα μπορούσε να, να εξασφαλιστεί η υποχρέωση λογοδοσίας και να μην έχουμε ε, διπλωματία πίσω από κλειστές πόρτες και μόνο. Νομίζω ότι για να εξασφαλιστεί κάτι τέτοιο χρειάζονται συγκεκριμένε συστάσει, συγκεκριμένε μέθοδοι ε, και πρακτικέ προκειμένου να μην γλιστρήσουμε πάλι προ τα πίσω προ μια κατάσταση αδιαφάνεια όπω αυτή που έχουμε συνηθίσει. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό που θα ζητήσω από, την, από το Κοινοβούλιο στις Επιτροπές ΑΦΚΟ και ΠΕΤΗ και στη συνέχεια και στην Ολομέλεια θα ήταν να εγκρίνουν τις συστάσεις που θα εκδώσω εγώ προκειμένου να ασκήσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πίεση στο Συμβούλιο για να ανταποκριθεί σε αυτές. Και αυτό θα γίνει πάρα πολύ σύντομα. Σας διαβεβαιώ. Όσον αφορά τα άλλα θέματα που θίξατε Όπω είπα, το, το ευκολότερο για μένα είναι να, να μου στέλνετε καταγγελίες προκειμένου να μπορώ να ερευνώ και να, και να ρωτώ το Συμβούλιο για ποιο λόγο στην κάθε ε, στην εκάστοτε περίπτωση έχουν αρνηθεί να δώσουν πληροφορίες και στη συνέχεια θα μπορέσω να αξιολογήσω πιο συνολικά την εκάστοτε περίπτωση για να δω αν πράγματι υπήρχαν λόγοι για τη μία αποκάλυψη πληροφοριών ή όχι. Αν δεν υπάρχει καταγγελία είναι πολύ δύσκολο να το κάνω. Σε μια άλλη, ε, ε, μια, ε, μια άλλη μέθοδος είναι να ερχόμαστε σε επαφές, σε συζητήσεις, σε ένα πιο άτυπο πλαίσιο προκειμένου να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε, σε κάθε περίπτωση καθώς αυτή θα ανακύπτει. Όπως είπα, το επιτελείο μου, η υπηρεσία μου είναι στη διάθεσή σας. Για μένα λοιπόν ε, όταν ε, συνέταξα την ομιλία που ήθελα να εκφωνήσω εδώ και βλέποντας ότι δεν υπάρχουν καταγγελίες παρά το γεγονός ότι υπάρχει δυσαρέσκεια από την πλευρά σας για το γεγονός ότι δεν προστατεύονται επαρκώς ε, τα δημόσια συμφέροντα ε, τονίζω ξανά αυτό, καταγγελίες. Ευχαριστώ κύριο Ντελάγκη. Κυρία Ντελάγκη από το ΕΛΚ παρακαλώ. Ευχαριστώ. Και ζητώ συγγνώμη που έχασα την εισαγωγή σας. Θα ήθελα να μάθω από την εμπειρία σας, γιατί σίγουρα γνωρίζετε την πρωτοβουλία ΚΟΣΑΚ και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Μπορεί να κάτι στην εισαγωγή σας, δεν το γνωρίζω. Ε, σύμφωνα με τη δική σας εμπειρία, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ενημέρωση που έχουν κάποια κράτη-μέλη όπου γίνεται έντονη συζήτηση για ευρωπαϊκά νομοθετικά θέματα και όπου οι υπουργοί στις εθνικές συζητήσεις λαμβάνουν κάποια θέση. Και από τη δική μου πείρα, πρακτικά την τελευταία δεκαετία έχω δει ότι υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης και αντιπαράθεσης και αντιπαραβολής αυτών που λένε οι υπουργοί στα κράτη-μέλη και ε, με την ενημέρωση που έχουμε εμείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο συχνά άτυποι ε, για το πώς συμπεριφέρονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για τη δική μου χώρα που είναι κάτω χώρες μπορώ αυτό να το κάνω γιατί παρακολουθώ τη συζήτηση στο Εθνικό Κοινοβούλιο και συχνά άτυπα παρακολουθώ τα τεκτενόμενα εδώ. Όπως είπατε δεν ε, κρατάνε και πρακτικά. Αλλά μαθαίνω τι συμβαίνει στο Συμβούλιο και πώς τοποθετεί τη χώρα μου. Και σε αρκετά νομοθετικά θέματα, όπου ήμουν ας πούμε εισηγήτρια, παρακολούθησα τι έγινε σε διάφορα κράτη-μέλη και ξέρω ποια είναι τα κενά. Φυσικά που δεν είχα ποτέ την ευκαιρία να έχω πλήρη εικόνα για τα 28 κράτη, για τα 27, αλλά είμαι πεπισμένη ότι υπάρχει αυτή η εικόνα. Σύμφωνα λοιπόν με τη δική σας εμπειρία, πώς μπορείτε να μας συμβουλεύσετε εμάς να εργαστούμε καλύτερα με τις πληροφορίες και την ενημέρωση που υπάρχει σε εθνικό επίπεδο, για να είναι πιο πλήρης η εικόνα και για τη δουλειά που κάνουμε εδώ για φορολογικά θέματα από αυτό αυτό που γίνεται τώρα σε σύγκριση με την περιορισμένη ενημέρωση που θα δεήσει να μας δώσει το Συμβούλιο, που ουσιαστικά είναι μηδενική. Τι μας συμβουλεύετε να κάνουμε. Το είπα και προηγουμένως, όταν είναι ευαίσθητο το θέμα, χρειάζεστε πολιτική υποστήριξη, κάποιος να λάβει αυτή την ευθύνη, το λάβαρο και να το προχωρήσει. Συγγνώμη, δεν αναφέρθηκα στην Κόζα και ιδιαίτερα στους Ολλανδούς που πραγματικά ανέλαβαν εδώ την πρωτοβουλία και ε, στην Προεδρία οπωσδήποτε την Ολλανδική έγινε πολύ μεγάλη δουλειά για τη διαφάνεια. Πόσες χώρες ήταν που υπέγραψαν, νομίζω 20, 20 εθνικά κοινοβούλια. Αυτό είναι μια καλή αρχή, αλλά σε τέτοιο επίπεδο θα πρέπει να γίνει. Στη δική μου δουλειά καμιά φορά δυσκολεύομαι να <laughs> τους κάνω να ενδιαφερθούν για κάποιες ε, συστάσεις. Αν δεν υπάρχει πολιτική υποστήριξη και συνένεση από την κοινωνία των πολιτών, διαφόρους πολιτικούς, κοινοβούλια, ΜΚΟ, ε, που εργάζονται όλοι προς την διακατεύθυνση και όταν το θέμα είναι ευαίσθητο είναι δύσκολο. Βεβαίως κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά η ΚΟΣΑ και τα Εθνικά Κοινοβούλια, ζωτική σημασία. Και ε, μας βοηθάει πάρα πολύ και αντίστροφα η δική μας δουλειά βοήθησε πολύ τους Ολλανδούς για να πιέσουν από τους τριμερείς διαλόγους και τη διαφάνεια και τις προτάσεις που κάναμε. Δεν είναι αυτή η επίσημη προφανώς συνεργασία, είναι άτυπη αλλά πολύ ε, βοηθάει. Αυτό που χρειάζεται είναι πραγματικά να αναλάβει κάποιος να το προωθεί αυτό το θέμα και να καταλάβει ο κόσμος πόσο σημαντικό είναι. Σας είπα, διάβασα την έκθεση της τελευταίας επιτροπής και ως πολίτης συνειδητοποίησα πόσο εκτεταμένο είναι αυτό το φαινόμενο και για ποια τάξη μεγέθους ε, πρόκειται και τι σημαίνει αυτό σε πραγματικούς όρους για τη ζωή των πολιτών. Βεβαίως έχει κάνει σπουδαία δουλειά και η χώρα σας και η ΚΟΖΑΚ και από πλευρά μου αυτό που μπορώ να κάνω είναι ότι θα, θα δώσω συνέχεια. Συνεχίζεται, βεβαίω συνεχίζεται, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα αυτή η προσπάθεια. Ευχαριστώ. Η κυρία Γοζιέγα από του Σοσιαλιστέ και Δημοκράτε, σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ καταρχά για τι συστάσει σα, οι οποίε είναι προφανώ πολύ σημαντικέ για το Κοινοβούλιο. Βλέπουμε ότι υπάρχει έλλειψη διαφάνεια στο Συμβούλιο, το οποίο παρεμποδίζει το έργο μα, ιδίω στα πλαίσια της ομάδας του κώδικα δεοντολογίας που επικρίθηκε και από την έκθεση τάξη 1 και τάξη 2. Η δική σας τώρα η έρευνα θα έλεγα ότι είναι κάπως γενική στη φύση της. Προβλέπετε να κάνετε μια ειδική έρευνα όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας του κώδικα δεοντολογίας προκειμένου να έχουμε συγκεκριμένες πλέον συστάσεις για τη συγκεκριμένη αυτή ομάδα εργασίας του Συμβουλίου που ασχολείται με ζητήματα φορολογικής ισότητας και μήπως θα σας βοηθούσε και μια επίσημη καταγγελία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πέρα από αυτό θα ήθελα να ασχοληθώ με την υπόθεση και την απόφαση Καπιτάνη σε σχέση με την πρόσβαση στα έγγραφα των τριμερών διαλόγων. Μετά την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστεύετε ότι έχουμε πλέον στα χέρια μας νέα πιο ισχυρά επιχειρήματα για να ζητήσουμε περισσότερη διαφάνεια από το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη. Κοιτάξτε, όπως έχετε συνειδητοποιήσει όλοι στην Επιτροπή αυτή, το ζήτημα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο από πολιτικής πλευράς. Κατά την προετοιμασία μου για την σημερινή ακρόαση, διάβαζα τα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την πολιτική διαφάνειας όσον αφορά την φορολογία και μία από τις φράσεις που πρόσεξα είναι αυτό το οποίο λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ένα γραφό ότι η φορολογία αγγίζει την ίδια την κυριαρχία, την εθνική κυριαρχία. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καταλαβαίνετε για ποιο λόγο τα φορολογικά ζητήματα είναι τόσο ευαίσθητα από πολιτική πλευρά. Από την άλλη, βέβαια, υπάρχουν όλε οι συστάσει που είχε κάνει και η δική σα επιτροπή και ανησυχίε που έχουν εκφράσει και άλλε κοινοβουλευτικέ επιτροπέ. Εγώ πραγματικά προσπαθώ να δω πώς μπορώ να εμπλακώ με τον πιο αποτελεσματικό και παραγωγικό τρόπο. Δεν με ενδιαφέρει απλώ να έρθω και να επαναλάβω την εργασία που έχουν ξεκινήσει άλλα θεσμικά όργανα, τα οποία μπορεί να είναι πολύ καλύτερα τοποθετημένα από μένα προκειμένου να κάνουν το έργο αυτό. Σίγουρα θα με βοηθούσαν οι καταγγελίες όπως σας είπα και ενδεχομένως και κάποια στιγμή θα μπορούσαμε να είχαμε και ένα πιο συλλογικής καταγγελίας. Πάντως θα ήταν πραγματικά χρήσιμα έστω και μία μεμονωμένη καταγγελία να υποβληθεί προκειμένου να μπορέσω να ασχοληθώ περισσότερο με τη συγκεκριμένη αυτή ομάδα εργασία του Συμβουλίου στην οποία αναφερθήκατε. Σα ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε αρκετά αποτελεσματικοί στη διαχείριση του χρόνου. Μα παραμένει λίγο χρόνο ακόμα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διαδικασία Catch the Eye εφόσον κάποιο άλλο θέλει να πάρει το λόγο. Δεν βλέπω κανέναν. Δεν ξέρω λοιπόν αν οι συγητέ θα θέλουν να ξαναπάρουν το λόγο για να πούνε κάτι σε αυτή τη φάση. Α, σα ζητώ συγγνώμη, δεν σα είχα δει, κυρία Αναγκόμε. έχετε το λόγο και μετά θα ακούσουμε τους υπόλοιπου τον κύριο Κόφοντ. Ευχαριστώ κύριε Ορέιλε, για τη θέση σας. Και πραγματικά εκτιμάμε την υποστήριξή σας. Μιλήσατε για την αδιαφάνεια την οποία επιβάλλει το Συμβούλιο ότι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί κακοδιαχείριση και στρεβλή διοικητική πρακτική. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι το 1 εκατομμύριο στο οποίο αναφερθήκατε, αλλά γνωρίζουμε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι τουλάχιστον 50 δισεκατομμύρια χάνονται από ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα κράτη-μέλη, ε, στις ενδομιλικές συναλλαγές που είναι ε, τρόπος χρηματοδότησης εγκληματικών οργανώσεων και τρομοκρατικών τύπου ISIS και al qaeda Αυτά τα λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή δεν είναι απλώς κακή διαχείριση και στρεβλή διοικητική πρακτική. Είναι υποβοήθηση οργανωμένου εγκλήματος και τρομοκρατικών ε, οργανώσεων για να συνεχίσουν το έργο τους ας πούμε στην απάτη με το ΦΠΑ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ και ένα χρόνο και πλέον έχει προτείνει δράσεις στα κράτη-μέλη και το αποτέλεσμα είναι μηδενικό. Τι λέτε, ε, κατανοώ ότι μπορεί κανείς να αγανακτεί για την εμπλοκή των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε επίπεδο Συμβουλίου, όχι μόνο για τα φορολογικά. Αλλά σωστά αναφερθήκατε ε, ε, ε και τη βαρύτητα του προβλήματος και η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, το ξέπλυμα χρήματος δηλαδή, είναι πραγματικά μεγάλο πρόβλημα. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα γνωρίζει και φυσικά το Συμβούλιο. Και την έκταση και το βάθος και το εύρος αυτού του προβλήματος. Και αυτό δείχνει ότι η δική σας Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να δρά και, να λειτουργεί απρόσκοπτα. Και οι συστάσεις να έχουν κάποια συνέχεια. Έχετε δίκιο. Και πάλι από την εμπειρία μου ως διαμεσολαβητρία εδώ και στη χώρα μου. όταν τα πράγματα είναι δύσκολα, πολιτικά, ευαίσθητα, φορτισμένα, όσο πιο συντονισμένη είναι η προσπάθεια, όσο περισσότερες μικρές ομάδες ε, ενώνουν ε, τις δυνάμεις τους για να αγωνίζονται προς την ίδια κατεύθυνση, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να το επιτύχουν. Γι' αυτό θα πρέπει ο κόσμος να ενημερώνεται σωστά και κάνουμε και τις συστάσεις. είμαστε και εμείς, αλλά κυρίως να ενημερώνουμε τους πολίτες για να πιέσουν προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ κύριο Σκόφωτ. Ευχαριστώ και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την ε, διαμεσολαβήτρια για τις ενδιαφέρουσες και πολύ καλές απαντήσεις της. Πρώτον, όπως είπατε αρχικά, εμείς ως ειδική επιτροπή που εξετάζει ζητήματα που σχετίζονται με ζητήματα φορολογικά, επιχειρήσεων, φοροαποφυγής κτλ. κτλ. Ε, όπως είπατε και εσείς, ε, το, το θέμα αυτό άπτεται τον ε, ε, οικονομικών εγκλημάτων, αλλά άπτεται και των δημόσιων θεσμών και της ικανότητάς τους να λογοδετούν, να είναι διαφανή και να μπορούν να, είναι κατανοητά κατανοητό προς τους πολίτες τι ακριβώς κάνουν. Γι' αυτό και είναι τόσο σημαντική η συνεργασία μας, θεμελιώδους σημασία θα έλεγα. Γιατί αν θέλουμε πραγματικά να οικοδομήσουμε μια δίκαιη ενιαία αγορά στην Ευρώπη, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχουν ε, ε, δυνατότητες σε μεγάλες, ε, μεγάλη επιχειρηματική όμιλη να φοροαποφεύγουν, να φοροδιαφεύγουν ε, τις τις προάλλες διαπιστώσαμε ότι η McDonald's για παράδειγμα δεν πληρώνει σχεδόν ούτε ευρώ φόρους στην Ευρώπη γιατί ε, τοποθετούν τα κέρδη τους εκτός Ευρώπης και φορολογούνται εκτός Ευρώπης δηλαδή. Γι' αυτό και πρέπει να εξασφαλίσουμε αυτή τη διαφάνεια και να κάνουμε να ε, ε, ε, ασκήσουμε πίεση ώστε οι κυβερνήσεις μας, τα κράτη-μέλη μας να λογοδοτήσουν γι' αυτά. Είναι καθήκον μας ως νομοθέτης και τουλάχιστον θα πρέπει να έχουμε εικόνα ποια είναι η στάση που τηρεί η χώρα του καθενός στο Συμβούλιο ώστε να μπορούμε να την κάνουμε και να λογοδοτήσει ε, κάτι αντίστοιχο θέμα αντιμετωπίσαμε και με το απόρριτο το τραπεζικό. Αυστρία, Λουξεμβούργο για παράδειγμα. Καταφέραμε ακόμη και να καταλήξουμε σε συμφωνία με την Ελβετία για να άρει το τραπεζικό απόρριτό της. Είναι σημαντικό είναι, είναι εφικτό να σημειωθεί πρόοδο, αλλά για να, για να σημειωθεί πρόοδο πρέπει να ασκηθεί πίεση στι κυβερνήσει μα, στα κράτη-μέλη μα. Και αυτό ε, θα έχει ε, τις, τα επιθυμητά αποτελέσματα και στο Συμβούλιο. Πάντω, αν δεν αλλάξουμε συμπεριφορά τώρα, θα υπάρξουν αρνητικότατες επιπτώσεις και στη μελλοντική συνεργασία μας. Και όπως είπα και αρχικά, δεν είναι δυνατόν να έχουμε ενιαία αγορά όπου έχουμε άρει όλα τα εμπόδια στην κυκλοφορία κεφαλαίων για παράδειγμα και ταυτόχρονα να επιτρέπουμε να υπάρχουν ε, αδιαφανείς φορολογικές συνεργασίες μεταξύ ε, ευρωπαϊκών χωρών με τρίτες χώρες ή μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών. Γι' αυτό και είναι σημαντικό ναι, τα ζητήματα που άπτονται των φορολογικών θεμάτων είναι ευαίσθητα και σημαντικά, αλλά υπάρχει και ένα ζήτημα που σχετίζεται με τη λογοδοσία των ε, θεσμικών οργάνων. Γι' αυτό και σας καλώ να συνεργαστούμε σε μεγαλύτερο βάθος για να ξέρουμε τι κάνει το Συμβούλιο, τι κάνει το ΕΚΟΦΗΝ, να, είμαστε, να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια ε, στα φορολογικά ζητήματα γιατί ε, υπάρχουν συγκεκριμένε χώρες οι οποίες έχουν λειτουργήσει στο παρελθόν και εξακολουθούν να το κάνουν ως ε, φορολογική παράδειση. Γι' αυτό και ε, όταν καταρτίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάλογο για τρίτες, για, για, τρίτες χώρες θα μπορούσαν σε αυτόν τον κατάλογο να ενταχθούν και ευρωπαϊκές χώρες, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί οι πρακτικές που ακολουθούν στο εσωτερικό τους προσυδειάζουν προς την πρακτική που ακολουθούν η φορολογική παράδειση. Γι' αυτό και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ και θέλω πάρα πολύ και εγώ να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας. Ευχαριστώ. Θέλω να επανέλθω στο, στην απάντησή σας ε, σχετικά με την διαφάνεια ε, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα. Χαίρομαι πολύ για την, για την ισορροπημένη θέση ε, που εκφράσατε. Εγώ έχω εμπειρία από κεντρικές τράπεζες και η διαφάνεια έχει ενισχυθεί πολύ στις κεντρικές τράπεζες, κάτι που έχει ενισχύσει και την αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής. Και νομίζω ότι οι αποφάσεις ε, πολιτικής που λαμβάνονται βεβαίως από κυβερνήσεις είναι λίγο διαφορετικές, αλλά παρόλα αυτά θέλω να μου πείτε τι πιστεύετε σχετικά με τη δυνατότητα αυξημένης διαφάνειας από το Συμβούλιο στο, στα θέματα της φορολογίας. Βεβαίως είναι πολύ ευαίσθητο το ζήτημα, είναι εθνική αρμοδιότητα κτλ. Αλλά κατά τη γνώμη σας υπάρχει ε, πιθανότητα να εξευρεθεί συμβιβασμός σε αυτό το θέμα ε, μπορούμε να βελτιώσουμε τον τρόπο λήψης αποφάσεων. Um, Κοιτάξτε, μαγική σφαίρα δεν έχω μπροστά μου. Δεν μπορώ λοιπόν να σας πω ακριβώς πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Όπως σας είπα, μου έκανε εντύπωση πραγματικά η σοβαρότητα του ζητήματος και πόσο διευρυμένο είναι το φαινόμενο αυτό. Και πώς ε, ουσιαστικά επηρεάζεται η ίδια η ζωή των πολιτών, πολλές φορές οι δημόσιες πολιτικές σε επίπεδο κρατών μελών από τα όσα αποφασίζονται. Σαφώς λοιπόν είναι προς το δημόσιο συμφέρον, υπάρχουν συμφωνίες και συμβασμοί όσον αφορά τη φορολογία σε επίπεδο συμβουλίου, αλλά θα πρέπει εν μη τι άλλο να γνωρίζουμε ποιε είναι οι παράμετροι τη συζήτηση, ποιε είναι οι διαφορετικέ τοποθετήσει των κρατών μελών. Εγώ θα ήθελα να γνωρίζω ποια είναι η στάση τη Ιρλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, των κάτω χωρών. Και πολύ συχνά όταν υπάρχει μία μυστικοπάθεια έτσι στο Συμβούλιο, δεν είναι ότι ε, το Συμβούλιο ουσιαστικά προσπαθεί να αποκρύψει κάποιες πληροφορίες από άλλες ομάδες στα πλαίσια του Συμβουλίου, αλλά από αρμόδιες άλλες ομάδες σε εθνικό επίπεδο. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε μια εύκολη απάντηση στα ζητήματα αυτά. Σαφώς θα πρέπει να υπάρχει μια συνειδητοποίηση πλέον του κοινού, μια ευαισθητοποίηση των πολιτών, γιατί αυτό θα ασκήσει πίεση και σαφώς θα πρέπει και η δική σας η Επιτροπή να συνεχίσει να ασκεί πίεση και περισσότερη διαφάνεια και εγώ αν μπορώ να σας βοηθήσω, σας είπα ότι μέσω συγκεκριμένων καταγγελιών θα μπορούσα να απευθυνθώ στο Συμβούλιο σε σχέση με τη συμμόρφωσή του, τη μη συμμόρφωσή του με συγκεκριμένους κανόνες. Σας ευχαριστούμε, ο κύριος Τελάνγκη έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ για την προθυμία σας να βοηθήσετε για να επιτευχθεί μεγαλύτερη διαφάνεια. Τώρα η ομάδα για τον κώδικα δεοντολογίας μας είπε η πρόεδρος στην Επιτροπή Πάναμα ότι δεν είναι επίσημο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά διακυβερνητικό όργανο. Και η δικαιολόγηση για την άρνηση ενημέρωσης είναι ότι δεν είμαστε ευρωπαϊκό όργανο και δεν είμαστε υπόλογοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εσείς τι λέτε. Σύμφωνα με τη δική σας εντολή μπορείτε να παρακαλείτε και διακυβερνητικά όργανα ε, να είναι πιο διαφανή και να αλλάξουν συμπεριφορά. Γιατί με αυτή την δικαιολογία όλα τα κείμενα ήταν μαυρισμένα, σβησμένα με μαύρο τα πάντα, εκτός από την ημερήσια διάταξη. Και η δικαιολογία ότι δεν σας οφείλουμε τίποτα να λογοδοτούμε, διότι δεν είμαστε ε, κοινοτικό ή ευρωπαϊκό όργανο, αλλά διακυβερνητικό. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό. Ευχαριστώ πολύ τη διαμεσολαβήτρια, λέει ο Πρόεδρος, για τη συνεισφορά τη αυτή. Έκανα μια ερώτηση, λέει ο κύριο Λάγκεν. μήπω να απαντήσει, κυρία Ρέιλι. Ναι, σε σχέση με αυτό. Ελπίζω να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία. Κατανοώ απολύτω τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις διαπραγματεύσεις, ιδιαίτερα σε επίπεδο συμβολίου κτλ. αλλά δικαιούνται να ενημερώνονται και οι πολίτες για τις συζητήσεις που γίνονται και με ποιο, σε ποιο πλαίσιο και με ποιο τρόπο. Και όταν υπάρχει ένα κενό ενημέρωσης, αυτό δίνει έδαφος σε ψευδείς ειδήσει και fake news και μπορεί να καλύψει το κενό αυτό πληροφόρηση κάποιο με τρόπο επιζήμιο για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή δεν θα πρέπει κανείς να φοβάται ε, να δημοσιεύονται τα πραγματικά γεγονότα και τα πραγματικά περιστατικά. Γιατί αυτό είναι και δικαίωμα των Ευρωπαίων πολιτών. Yes, well, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ και πάλι κύριε Ορέιλη. Ελπίζω να απαντήσει σύντομα το Συμβούλιο στις συστάσεις σας και να απαντήσει και επικοδομητικά. η διαφάνεια των εργασιών τους ελπίζω να αυξηθεί προς όφελος και των υπόλοιπων θεσμικών οργάνων, αλλά κυρίως του κοινού, των πολιτών. Βεβαίως και εμείς θα εξετάσουμε το δεχόμενο να κάνουμε επίσημες καταγγελίες ε, στην κυρία Ρέιλι. Θα το δούμε αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Ρέιλι για την παρουσία σας, τις απαντήσεις σας και την πάγια προσπάθειά σας να αυξηθεί η διαφάνεια. Ευχαριστώ πολύ. So this us to the second panel. Λοιπόν, περνάμε στο δεύτερο πάνελ της σημερινής ακρόασης. Ευρωπαϊκός κατάλογος μη συνεργαζόμενων χωρών. Υπάρχει κάποιο περιθώριο βελτίωσης. Θα ήθελα πολύ σύντομα να σας παρουσιάσω τους ομιλητές που έχουμε στο πάνελ αυτό. Καταρχάς ο κύριος Βαλέρ Μουταγλιέ, Διευθυντή στη Διεύθυνση ΔΕΛΤΑ, άμεση φορολόγηση, φορολογικό συντονισμό, οικονομικέ αναλύσει και αξιολόγηση από την DG Taxu της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έπειτα η Έλλη Βαν Ντεβέλντε, καθηγήτρια φορολογικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Χάσελ του Βελγίου, Άλεξ Κόπχαμ, εκτελεστικός επικεφαλής του Δικτύου Φορολογικής Δικαιοσύνης και ο κύριος Γιώχαν Λάγκερόκ, ο οποίος είναι σύμβουλο σε ζητήματα κοινοτική πολιτικής όσον αφορά τη φορολογία και την ανισότητα εξ ονόματος της Oxfam την ίδια διαδικασία θα ακολουθήσουμε στους γύρους ερωτήσεων που θα γίνουμε πέντε λεπτά ερώτηση για την υποβολή της ερώτησης και την απάντηση και θα ξεκινήσουμε με μία σύντομη παρουσίαση, σύντομη παρέμβαση από τους ομιλητές. Πρώτος θα πάρει το λόγο ο κύριος Βαλέρ Μουταρλιέ και καθότι μιλάμε για διαφάνεια μέρα Ο κύριος Βαλιάχ Μουταγλιά έχει τα γενέθλιά του, επομένω έχει γίνει ένα χρόνο ακόμα πιο σοφός. Το ευχόμαστε χρόνια πολλά και κύριε Βαλιάχ Μουταγλιά σας δίνω και το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχει καλύτερο τρόπος να περάσει κανείς ε, το απόγευμα το γενεθλίων του από το να βρίσκεται εδώ στη δική σας την Επιτροπή. Με χαρά λοιπόν είμαι εδώ για να σας ενημερώσω για τη στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τον κοινό αυτό κατάλογο. Τον Ιανουάριο του 2016 ξεκίνησε αυτή η πρώτη στρατηγική για την κατάρτιση του καταλόγου αυτού και έπειτα τον Δεκέμβριο του 2017 τα κράτη-μέλη ενέκριναν τον πρώτο τέτοιο κατάλογο σε ευρωπαϊκό επίπεδο αφού κάνανε μια διεξοδική ανάλυση και έλεγχο 92 φορολογικών επικρατιών παντού στον κόσμο. επικεφαλίσταν το Συμβούλιο με την τεχνική υποστήριξη της Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Ο συντονισμός επικεντρώθηκε και βασίστηκε και στην πολιτική βούληση αναγνώρισης του καταλόγου αυτού και κυρίως υπόθηκε ότι μέσω της διαδικασίας αυτής η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφερε να κάνει τους διεθνούς της, διεθνούς της εταίρους να ακούσουν περισσότερο ποιες είναι οι προσδοκίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα φορολογικά θέματα. Είδαμε ότι οι περισσότεροι εταίροι συμμετείχαν επικοδομητικά Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατάρτισης του καταλόγου αυτού, οι περισσότερες δικαιοδοσίες, οι περισσότερες χώρες ανέλαβαν πολιτική δέσμευση προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις που είχαν ε, ε, εντοπιστεί στα πλαίσια της έρευνας αυτής. Το βασικό κριτήριο το οποίο χρησιμοποιήθηκε όσον αφορά τη διαφάνεια ήταν αρκετά ευρύ προ... προκειμένου να καλύπτονται όλε οι πιθανέ ελλείψει. Δηλαδή, όχι μόνο η διαφάνεια που ήταν το βασικό κριτήριο, αλλά και οι βλαβερέ φορολογικέ πρακτικέ, καθώ επίση και οι κίνδυνοι που έχουν να κάνουν με τι δικαιοδοσίε εκείνε που χρησιμοποιούν μηδενική φορολόγηση. Περίπου 100 λοιπόν τέτοιες ε, φορολογικές επικράτειες θα έπρεπε να αναλάβουν δράση μέχρι το τέλος του έτους. Άλλες πάλι ανέλαβαν δράση για να βελτιώσουν το φορολογικό τους καθεστώς, το φορολογικό τους σύστημα. Και έπειτα οι επικράτειες εκείνες οι οποίες έχουν μηδενική φορολογία υποχρεώθηκαν να προβλέψουν αλλαγές στην εσωτερική τους νομοθεσία. Μέχρι το τέλος του έτους καλούνται οι χώρες αυτές μέχρι το τέλος του 2019 όσον αφορά τις αναπτυσσόμενες χώρες προβλέπεται ότι οι χώρες αυτές θα πρέπει να επιφέρουν τι απαραίτητες αλλαγές. Τις βοηθά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Έχουμε ξεκινήσει έναν ευρύ διάλογο με τις χώρες αυτές, εξηγώντας τους πώς έχουν τα πράγματα, στηρίζοντάς τους από τεχνική πλευράς και αυτό που μας ενδιαφέρει να διασφαλίσουμε ότι κάθε χώρα συνειδητοποιεί τι πρέπει να κάνει. Οποιαδήποτε χώρα από την άλλη δεν συνεργάζεται και δεν εφαρμόζει τις δεσμεύσεις της θα πρέπει να αντιμετωπίσει επιπτώσεις. Διαφορετικά δεν έχει καμία βαρύτητα ο κατάλογος αυτός. Η απειλή αυτή των κυρώσεων θα πρέπει πραγματικά να χρησιμοποιηθεί για τις χώρες εκείνες οι οποίες δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα. Και θα ήθελα τώρα να αναφερθώ στην εργασία αυτή την πολύ σημαντική βρίσκεται εν εξελίξη που έχει να κάνει με τα μέτρα άμυνα. Εμεί έχουμε πει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε αποτελεσματικά, αποτρεπτικά μέτρα αμυντικά, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα κράτη-μέλη κατά των φορολογικών αυτών επικρατιών. Η άποψη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι υπάρχει ακόμα ένα περιθώριο βελτίωση προτού πετύχουμε το στόχο αυτό. Οι φυστάμενε πρακτικέ αποδεικνύουν ότι τα αμυντικά αυτά μέτρα, αμυντικέ πρακτικέ δεν είναι αρκετά συντονισμένε ούτε αρκετά αποτελεσματικέ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη δική της την πλευρά έχει καταβάλει προσπάθειες προκειμένου να κάνει τον κατάλογο αυτό πιο ισχυρό. Προβλέπουμε πλέον συγκεκριμένα μέτρα στα πλαίσια της κοινοτική νομοθεσίας προκειμένου να υπάρχουν πραγματικά επιπτώσεις για τις χώρες εκείνες που συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και που δεν λαμβάνουν μέτρα για να συμμορφωθούν και ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να χρησιμοποιηθεί από δικαιοδοσίες οι οποίες χρησιμοποιούν πρακτικές για την παράκαψη της φορολογίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει άμεση διασύνδεση πλέον ανάμεσα στην κοινοτική χρηματοδότηση και τις χώρες εκείνες αποδέκτες της χρηματοδότησης αυτής οι οποίες προωθούν πρακτικές φορολογικής ε, αποφυγής, φορολογικής παράκαμψης. Η στάση μας αυτή συνάδει με τη γενικότερη δέσμευση που έχουμε να είμαστε απόλυτα σαφείς, διαλλακτικοί και να μπορούμε να συνεργαζόμαστε με όλους τους ε, εταίρους μας που προβλέπονται ε, στη λίστα αυτή. Συνεργαζόμαστε και με τη Διαμεσολαβήτρια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τονίσει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό διαδικασία που θα χρησιμοποιηθεί για τον κατάλογο αυτό να είναι απόλυτα διαφανή και ανοιχτή. Οι τρίτε χώρε θα πρέπει να δουν, όπω και οι πολίτε οι ίδιοι, ότι υπάρχουν συγκεκριμένα αντικειμενικά διαφανή κριτήρια που χρησιμοποιούνται στον κατάλογο αυτό. Επίτροπο Μοσκοβισή άσκησε πίεση στου εταίρου στα πλαίσια του ΕΚΟΦΗΝ προκειμένου να δημοσιοποιηθεί η επιστολή που έχουν στείλει τρίτες χώρες στην ομάδα του κώδικα δεοντολογίας πάνω από το ίμιση των δεσμεύσεων των τρίτων αυτών χωρών έχουν ήδη κοινοποιηθεί και περιμένουμε ότι η κοινοποίηση θα υπάρξει και για τις υπόλοιπες δεσμεύσεις των υπολείπων τρίτων χωρών που βρίσκονται σε αυτόν τον κατάλογο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτός ο βαθμός διαφάνειας γιατί κατά αυτόν τον τρόπο ασκείται μεγαλύτερη πίεση στις χώρες αυτές. Θα πρέπει προφανώς ο κατάλογος αυτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεχίσει να εξελίσσεται προκειμένου να έχει κάποια σημασία και κάποια βαρύτητα. Αποφασίσαμε πέρυσι ότι θα πρέπει να έχουμε περισσότερα κριτήρια όσον αφορά τον πραγματικό δικαιούχο και όσον αφορά την εφαρμογή των ελάχιστων προτύπων BEPS για την ε, καταπολέμηση δηλαδή τη διάφορη φορολογική βάση και τη μετατόπιση των κερδών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει προφανώ να υποστηρίζει τη στρατηγική αυτή για τον κατάλογο αυτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση η νέα αυτή στρατηγική προφανώς έχει ένα περιθώριο βελτίωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί μια πολύ σημαντική πηγή έμπνευση και νέων ιδεών σχετικά με τον κατάλογο αυτό και εκτιμούμε όλος ιδιαιτέρως τη συμβολή των μη κυβερνητικών οργανώσεων που συμμετέχουν στην πλατφόρμα χρηστής φορολογικής διοίκησης από την οποία προέκυψε και αυτός ο κατάλογος. Είμαστε στη διάθεση όλων αυτών των εταίρων για να ακούσουμε τις περαιτέρω ιδέες που ενδεχομένω να έχουν και προκειμένου να καταφέρουμε με τη δική τους τη βοήθεια να διαμορφώσουμε καλύτερα αυτόν τον κατάλογο. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ε, Ήδη το επίτευγμα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ότι καταφέραμε να θεσπίσουμε τον κατάλογο αυτό. Προσβλέπουμε σε μια επικοδομητική συνεργασία με το Κοινοβούλιο και με εξωτερικούς φορείς και είμαστε πεπισμένοι ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να βασιζόμαστε στη δική σας την υποστήριξη και στην πίεση που εσείς μπορείτε να ασκήσετε στα κράτη-μέλη για να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους. Ευχαριστώ κύριε Βαντεβέλτε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, πρόσκληση. Είχα προσέλθει και σε εργαστήρια των Επιτροπών Τάξη 1 και 2 και θέλω να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόοδο που έχει σημειώσει και τις προτάσεις που έχει υποβάλει. Μου ζητήσατε να απαντήσω σε δύο ερωτήματα σήμερα. Πρώτον, ποια είναι η δική μου αξιολόγηση σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο των μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών σε φορολογικά ζητήματα όσον αφορά τη διαδικασία. Αν θεωρώ ότι η διαδικασία αυτή είναι αξιόπιστη και ποιε θα ήταν οι δικέ μου συστάσει για, για βελτίωση τη διαδικασία. Και δεύτερον, αν πιστεύω ότι ο κατάλογος αυτός πρέπει να περιλαμβάνει και κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προσφέρουν επιθετικές φορολογικές πρακτικές και δυνατότητες. Θέλω να απαντήσω και στα δύο ερωτήματα με μία απάντηση, γιατί θεωρώ ότι διασυνδέονται αυτά τα δύο θέματα. Κατανοώ ότι ένας μαύρος κατάλογος φορολογικών παραδείσων είναι ένα εργαλείο, όχι πανάκιο, προκειμένου να ασκηθεί πίεση σε συγκεκριμένους φορολογικούς παραδείσους ώστε να εφαρμόζουν σε συγκεκριμένα πρότυπα και κανόνες που βεβαίως θα πρέπει να δεσμεύουν και τα ίδια τα κράτη-μέλη. Και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ και την ε, υπηρεσία έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που κατέληξε στο, στο συμπέρασμα ότι αυτή τη στιγμή ε, δεν περιλαμβάνονται κράτη-μέλη που δεν σημαίνει όμως ότι έχουν ασυλία όσον αφορά την κριτική. Γι' αυτό και ε, όσον αφορά την, ε, τον ε, εντοπισμό και τον προσδιορισμό επιθετικών φορολογικών πρακτικών που χρησιμοποιούν μεγάλες πολυεθνικές και επιχειρηματικοί όμιλοι ε, είναι ένα θέμα το οποίο βεβαίως ε, εμφανίζεται και στα κράτη-μέλη και δεν αφορά μόνο ε, τις εταιρείες θηρίδες. Ως ακαδημαϊκός λοιπόν θέλω να επικεντρωθώ σε κάποια ζητήματα και να κάνω κάποιες προτάσεις. Κατά τη γνώμη μου, ο φορολογικός σχεδιασμός, ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός και οι απάτες στον τομέα της φορολογίας από την άλλη πλευρά δεν ε, έχουν το ίδιο, την, την, ίδια σημασία. Στον φορολογικό, ο φορολογικός σχεδιασμός αφορά το να εκμεταλλευτεί κανείς κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά ή παραθυράκια ή αναντιστοιχίες που υπάρχουν μεταξύ διαφόρων φορολογικών ε, συστημάτων και η Κομισιόν ε, ορίζει τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό ε, ως προσπάθεια να εκμεταλλευτεί κανείς. Αυτός ο ορισμός είναι ασαφής. Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς εννοεί η Κομισιόν με τον όρο επιθετικός. Πότε ένας φορολογικός σχεδιασμός είναι επιθετικός και πότε είναι ο υπερβολικός φορολογικός σχεδιασμός απλά υπερβολικός, δεν είναι απαραίτητα κακός και ακόμη και ο επιθετικός φορολογικός ε, σχεδιασμός δεν είναι παράνομος σε πολλές χώρες γιατί δεν παραβιάζεται η νομοθεσία. Κατά τη γνώμη μου ο φορολογικός σχεδιασμός γίνεται επιθετικός όταν υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη νομική μορφή και την οικονομική ουσία. Θεωρώ ότι είναι μια αναγκαστική ε, ανισορροπία μεταξύ του πνεύματος και του γράμματος του νόμου. Όσο περισσότερο υπάρχει ε, έλλειψη σεβασμού προς το, πνεύμα του νόμου, ε, τόσο περισσότερη απόκληση υπάρχει και από το γράμμα του. Δεν πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες, αλλά στην ουσία γίνεται κατάχρηση του γράμματος του νόμου από αυτές τις πρακτικές και στη συνέχεια ε, ε χρειάζονται κανόνες για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής. Είναι όμως πιθανό για εταιρικούς λόγους τα κράτη-μέλη να επιτρέπουν να υπάρχουν εταιρείε θηρίδες που δεν έχουν καθόλου οικονομική δραστηριότητα στην επικράτειά τους. Αυτό όμως είναι κάτι διαφορετικό, διότι αυτό αποτελεί εθνική αρμοδιότητα, επιλογή των κρατών μελών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δικά τους καθεστώτα όσον αφορά την έδρα των εταιριών και τις μεταβιβάσεις ε, των, των εδρών. Ε, αυτό είναι σύμφωνο με την ελευθερία εγκατάστασης και με την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Το να ε, πληρώνει κανείς φορούς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία βεβαίως είναι σύνομο. Πρόβλημα υπάρχει όταν δεν υπάρχει πραγματική μεταφορά έδρας και ε, όταν υπάρχει απλά μια ε, ε, μεταφορά ως «ή». Όταν δηλαδή πλήττεται το κράτος μέλος όπου μια εταιρεία έχει την πραγματική της έδρα αλλά εμφανίζεται να την έχει αλλού. Αυτό βεβαίως δεν αφορά μόνο την, τον απλό φορολογικό σχεδιασμό και γι' αυτό χαρακτηρίζεται επιθετικός. Γι' αυτό και κάποιες φορές αυτά τα κράτη-μέλη που προσφέρουν αυτές τις δυνατότητες χαρακτηρίζονται ως φορολογική παράδειση. Για τις νομικές λοιπόν ε, πλευρές έχω τοποθετηθεί και στην απάντηση που σας έχω αποστείλει ακόμα και ο νομοθέτης ε, ε, ενθαρρύνει το φορολογικό σχεδιασμό αφού δίνει φοροπολογίες τι ακριβώς, ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον, σε κάποιες συγκεκριμένε φοροαπαλλαγές, όπως για παράδειγμα αν κάνεις αποταμίευση σε κάποιο συνταξιδοτικό ταμείο, στο Βέλγιο, που υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα, και, ή όταν για παράδειγμα φορολογείς την κατανάλωση ζάχαρης, ε, και τον φορολογικό σχεδιασμό. Είναι και αυτό μια μορφή φορολογικού σχεδιασμού, η οποία μάλιστα έχει και τη βούλα τη της κυβέρνησης. Και αυτό βεβαίω το λαμβάνουν υπόψη του οι φοροτεχνικοί που συμβουλεύουν πολυεθνικές εταιρείε και μεγάλου επιχειρηματικού ομίλους. Υπάρχει μάλιστα φορολογικό ανταγωνισμό ο οποίο οργανώνεται από τι κυβερνήσει και που, διευκολύνει τι πολυεθνικές εταιρείε, αλλά και άτομα μεμονωμένα προκειμένου να εκμεταλλεύονται αυτόν τον φορολογικό ανταγωνισμό. Και αυτά τα ζητήματα βεβαίω έχουν και ένα διασυνοριακό χαρακτήρα οι φορολογικέ, ε, βεβαίω, ε, ο φορολογικό σχεδιασμό δεν αφορά όμω μόνο το διασυνοριακά ε, τι δραστηριονομικές δραστηριότητε, αλλά και τι δραστηριότητε μια εταιρεία εντός στο, στο πλαίσιο μια συγκεκριμένη χώρα. Υπάρχει λοιπόν ένα φορολογικό ανταγωνισμό, επιζήμιο, ο οποίο συνδέεται με τη φοροαποφυγή, φοροδιαφυγή και πρέπει να δούμε αν πρόκειται για αντιμετώπιση ή καταπολέμηση ε, ή αν θέλουμε να, να τον, ε, τις παραβίασεις των, το, αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε τους κανόνες που υπάρχουν ή την παραβίαση των κανόνων. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι ο κατάλογος των φορολογικών παραδείσεων μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο για την καταπολέμηση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού που οργανώνεται από τρίτες χώρες. Θέλω λοιπόν στην, παράμβα, στην παρέμβασή μου να αναφερθώ στην ανάλυση που, είχα, ε, που είχε συντάξει ο κύριος Τζέφρι Owens από το Πανεπιστήμιο της Βιέννης για την ε, Επιτροπή Tax 1, όπου εντόπισε συγκεκριμένες φορολογικές ε, διαφορές μάλλον στη φορολογική πολιτική των κρατών μελών τα επόμενα 10 χρόνια η συμφιλίωση και ο συμβιβασμό των φορολογικών πολιτικών των κρατών μελών είναι μία από τι βασικότερε προκλήσει που αντιμετωπίζουμε. Πρέπει αφενό να προσελκύσει κάθε χώρα ε, επενδύσεις. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να σταθεί στον διεθνή ανταγωνισμό και επίσης οι μικρές χώρες ε, χρησιμοποιούν συγκριτικούς ε, δείκτες για τα φορολογικά τους συστήματα που βασίζονται στους ανταγωνιστές τους. Έτσι λοιπόν εμφανίζονται επιζήμιες φορολογικές πρακτικές. Η απάντηση του κυρίου Οέντς στην παγκοσμιοποίηση είναι καλύτερη συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει κάποιο να εκχωρήσει ένα μέρος της κυριαρχίας του. Για τις τρίτες χώρες αυτό βεβαίως σημαίνει να τους ασκηθούν πιέσεις ώστε να ενισχύσουν τη φορολογική τους ε, διαφάνεια και τη δικαιοσύνη των φορολογικών τους συστημάτων. Και αυτό θεωρώ και εγώ ότι είναι το βασικό ζήτημα που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή και που αποτελεί το κεντρικό, το κομβικό στοιχείο για την αντιμετώπιση των επιθετικών ε, φορολογικών πρακτικών φορολογικού σχεδιασμού. Αλλιώς θα υπάρχει μια, ένας ανταγωνισμός προς τα κάτω για το ποιο θα ζητάει από τις εταιρείες το, τους λιγότερους φόρους. εφόσον λοιπόν τα κράτη-μέλη επιμένουν στην εθνική τους κυριαρχία όσον αφορά τα φορολογικά τους ζητήματα, μόνο οι εκθέσεις της ομάδας για τον κώδικα διοντολογίας, οι εκθέσεις του Κοινοβουλίου και μπορούν να αποτελέσουν ε, πηγή άσκησης πίεσης. Στο παρελθόν έχουν ε, συνταχθεί τέτοιου είδους ε, κείμενα και τέτοιου είδους εκθέσεις έχουν αποβεί πολύ χρήσιμες. Γνώμη μου λοιπόν είναι ότι οι τελικές εκθέσεις σχετικά με τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό είναι πολύ χρήσιμο, χρήσιμες και θα μας βοηθήσουν στην καταπολέμηση των, του επιθετικού φορολογικού ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών. Ωστόσο, λόγω του καθεστώτος που ισχύει, η επιβολή κυρώσεων στα, στα κράτη-μέλη και στις πολυεθνικές που επιδίδονται σε, μια τέτοια, ένα τέτοιο επιθετικό φορολογικό ανταγωνισμό είναι ε, η παρακολούθηση των, ε, των, της επιβολής των, των ε, κανόνων που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις. Καθηγήτρια, σας παρακαλώ, μπορείτε να ολοκληρώσετε για να μπορέσετε και να απαντήσετε στις ερωτήσεις των μελών. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι, τα, ότι τρίτες χώρες και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να τοποθετηθούν στον ίδιο κατάλογο μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών, αλλά του υπάρχει ενιαία αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, ο φορολογικό σχεδιασμό και ο επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό πολλέ φορέ συνάδουν με το ευρωπαϊκό δίκτυο εφόσον δεν υπάρχει διάκριση ει βάρο συγκεκριμένων εταιριών των κρατών μελών. Επίση, οι εθνικέ νομοθεσίε, αλλά και οι διοικητικέ πρακτικέ των κρατών μελών πρέπει πάντοτε να συνάδουν με τι οδηγίε της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη φορολογική διαφάνεια κτλ. Ό,τι αφορά για τα κριτήρια, για ένα κατάλογο ε, φορολογικών παραδείσων, και εδώ τελειώνω, ε, διαφάνει για τα φορολογικά, δίκαιη φορολόγηση και εφαρμογή μέτρων anti-BEPS, ε, θα πρέπει να υπάρχουν πιο συγκεκριμένα κριτήρια και νομικής φύσεως να περιχαρακωθούν κάποια καθεστώτα που προστατεύουν την εθνική οικονομία Ε, ε, τι γίνεται με τη φορολόγηση των ε, διαμενόντων των στη χώρα και των μη Αυτά ήταν τα κριτήρια του ΟΣΑ του 1998. Τι γίνεται με τους φορολογικούς ελέγχους σε τρίτες χώρες. Τι γίνεται με τα προγράμματα συμμόρφωσης των εταιρικών φόρων. Τι γίνεται με τα συστήματα των tax rulings των φορολογικών συμφωνιών. Τι γίνεται με την προσφυγή στη δικαιοσύνη. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να τα εφαρμόσουν όλα αυτά για να ε, αντιμετωπίσουν την επιθετική φορολογική ε, πρακτική και σχεδιασμό των πολυεθνικών. Ε, των πολυεθνικών. Χαίρομαι για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω εδώ και για τη δουλειά σας είναι πάρα πολύ σημαντική ε, για τον έλεγχο ε, αυτό σε αυτό τον τομέα που όπως ακούσαμε ε, θα πρέπει να μαθαίνουν πολύ περισσότερα οι πολίτες σχετικά με τη λήψη των αποφάσεων σε αυτό τον τομέα. Εμείς είμαστε εδώ ως κοινωνία των πολιτών, λέει ο κύριος Άλεξ Κόφαμ από το δίκτυο για φορολογική δικαιοσύνη. Ε, εμείς θεωρούμε το φόρο όχι απλώς έσοδο αλλά και ε, στοιχείο αναδιανομής. Ε, θα πρέπει να φορολογείται σωστά ο καπνός ή οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα που βλάπτουν το περιβάλλον με σωστό τρόπο και θα πρέπει να υπάρχει και αντίστοιχη διακυβέρνηση και να φορολογούνται οι επιχειρήσεις εκεί που έχουν κέρδη. Γιατί υπάρχουν θέματα και διακυβέρνηση και θέματα ε, διαφθοράς ε, και θέματα λογοδοσίας. Ε, γι' αυτό δημιουργήθηκε το δίκτυό μας. Η φόροι είναι πολιτικό θέμα. Τέθηκε το θέμα και της εθνικής κυριαρχία και της φορολογική κυριαρχία δεν είναι απλώς το θέμα ότι έχουν το δικαίωμα οι πολίτες να γνωρίζουν τι γίνεται με τη φορολογία, αλλά γιατί ε, τα φορολογικά ζητήματα μπορούν να επηρεάσουν την κυριαρχία των κρατών μελών και τη διακυβέρνησή τους. Σε ποιο βαθμό η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν είναι πρόθυμη να παρακάμπτει την κυριαρχία αλλού για να την προστατεύει εδώ και σε άλλες χώρες. Ακόμα αυτά τα πράγματα δεν είναι σαφή ε, ούτε προς τη μία κατεύθυνση ούτε προς την άλλη. 500 δισεκατομμύρια δολάρια είναι το διαφυγόν κέρδος μάλλον από τις πολυεθνικές ε, και από τις offshore. Ε, και αυτά υποσκάπτουν βαθιά την κυριαρχία των κρατών τη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλού και ε, προέρχονται από κάποιες χώρες ε, που με μυστικοπάθεια και με μεγιστοποίηση κέρδους ευνοούν κάποιες πολυεθνικές εταιρείες για την ε, απόκρυψη αυτών των εσόδων. Χρειάζεται ένας μηχανισμός λοιπόν για να αλλάξει αυτό και να ευθύγραμμεστεί κάπως στα πλαίσια της πολιτικής λήψης, αποφάσεων, λήψης πολιτικών αποφάσεων. Ας πούμε ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επιβάλλει κάποια πράγματα στην Αμίμπια που δεν έχει φορολογική συμπεριφορά τέτοια ώστε να επηρεάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη, για τις Ηνωμένε Πολιτείες Αμερικής μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να τις πειθαναγκάσει. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη απειλή από το φορολογικό απόρριτο και το οικονομικό απόρριτο. Έχουμε απαντήσει γραπτός στις ερωτήσεις και έχουμε μπει σε κάποια στοιχεία που δεν θα επαναλάβω. Ε, πάντως το βασικό που ακούσαμε και προηγουμένως είναι ότι η λίστα, ένας κατάλογος θα πρέπει να είναι αντικειμενικά επαληθεύσιμος. Και ακούσαμε και από την ομάδα ε, επαφής, η ε, ομάδα μάλλον για τον κώδικα δεοντολογίας, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι οι πολίτες δεν τα γνωρίζουν και δεν μπορούν να ε, ζητήσουν από τις κυβερνήσεις να λογοδοτήσουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ως διεθνής ε, πρωταγωνιστής δεν μπορεί να, να αναλάβει δράση ε, με ετεροδικία. Τι μπορεί να γίνει βραχυπρόθεσμα, να παραμείνει ως έχει κατάθεση. Το θέμα είναι να είναι πλήρως ε, διαφανείς όλες οι αποφάσεις και ε, όλες ε, οι συζητήσεις για τις χώρες αυτές. Τους επόμενους μήνες θα δούμε μια κατάσταση όπου θα εμφανιστούν οι Ηνωμένε Πολιτείε ως χώρα που πρέπει να εγγραφεί στο συγκεκριμένο κατάλογο βάσει των κριτηρίων του Και εδώ θα υπάρξει ένα θέμα αν, ε, αντιπίνων, ε, αντιμέτρων. Ας πούμε, όταν οι πολυεθνικές κάνουν την έκθεση αναχώρα και αναφέρεται η χώρα, ως χώρα αυτή οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θα αναλάβουμε δράση εναντίον των Ηνωμένων Πολιτείων ή μόνο κατά της Ναμίμπια και άλλων τέτοιων χωρών. Βεβαίω καλωσορίζουμε αυτή την εξέλιξη. Πιο μακροπρόθεσμα τώρα σε μια διετία ή τριετία και μπορεί η δική σας επιτροπή να συνεισφέρει προς την κατεύθυνση αυτή. Πώς βγαίνετε από μια θέση όπου αναπόφευκτα είναι μια θέμητη ε, πρακτική πλουσίων χωρών να επιβάλλει ε, την άποψή της σε κάποιες άλλες χώρες σε κάτι που ισχύει παγκοσμίω και τι θα γίνει με τι Ηνωμένε Πολιτείε. Πώς θα τις πιθαναγκάσουμε ε, και να μην είναι αυτό μια σύγκρουση μόνο Ευρωπαϊκής Ένωσης Ενωμένων Πολιτειών αλλά ευρύτερη. Αυτό έχει συζητηθεί επανειλημμένα και σε ένα συνέδριο για τη φορολογική διαφάνεια και φορολογική κυριαρχία που είναι αλληλένδετα. Και εκεί υπόθηκε ότι ε, πρέπει να γίνει αυτή η πλατφόρμα το 2003 η αλφαβήτα είναι αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών με τις εταιρείες, όχι με τους φίλους σας ή τις μεγάλες εταιρείες, με όλες τις δικαιοδοσίες. Και η Ελβετία να ανταλλάσσει πληροφορίες και ενημέρωση, όχι μόνο με τη Γερμανία, αλλά και με το Μαλάουι, ας πούμε. Να γνωρίζουμε απολύτως ε, ποιος είναι ο τελικός δικαιούχος, ο, ο, ο ιδιοκτήτης μιας εταιρείας και οι πολυεθνικές να αναφέρουν τα κέρδη και τις δραστηριότητες αναχώρα είδαμε πώς άλλαξαν τα πράγματα. Πριν από 15 χρόνια θα μας είχαν χλεβάσει αν κάναμε αυτές τις προτάσεις. Τώρα υπάρχει ευκαιρία να ε, βρεθεί συνένεση, ε, απουσία των Ηνωμένων Πολιτειών μάλλον, και να κάνουμε ένα βήμα ακόμα περισσότερο προς ε, την πολυμερή συνεργασία και να ενισχύσουμε την κυριαρχία όλων των κρατών μέλων. Όχι μόνο να υπερασπιζόμαστε τον χώρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα φέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολύ ε, ισχυρότερη θέση και μοίρα και επίσης η ε, αηφόρος και βιώσιμη ανάπτυξη θα είναι ένας από τους σημαντικούς στόχους τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λάγκεροκ. Γεια σας. Πρόεδρε, αντιπρόεδροι, αγαπητοί βουλευτές. Ε, χρόνια πολλά, κύριε ε, Μουχτάνια, για τα γενέθλιά σας. Ε, σας ευχαριστώ που με καλέσατε εδώ ε, για να σας δώσω τις απόψεις της Oxfam για το κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μη συνεργάσιμες χώρες. Είναι η περίφημη μαύρη λίστα. Εγώ θα την έλεγα γκρίζα. Στο τέλος ομιλίας μου θα σας αναφέρω και κάποιες συστάσεις για να γίνει καλύτερη αυτή η λίστα και πιο αποτελεσματική. Και αυτή ήταν και η ερώτηση βασική που ε, μας κάνατε. Σε πάνω από 90 χώρες είναι παρούσα η Oxfam για την πολέμηση της φτώχειας και την προογωγή της ε, ισότητας. Ασχολούμαστε με φορολογικά θέματα εδώ και χρόνια. Η φορολογική παράδειση είναι ε, το απόγειο της φορολογικής κούρσας προς τα κάτω και αυτό δημιουργεί πάρα πολλές ε, φτωχές χώρες στον κόσμο. Γι' αυτό ε, έχουμε ασχοληθεί και πέρσι τον Νοέμβριο εκδώσαμε τη μαύρη λίστα μας με νέα κριτήρια που ελέγχουμε τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κοιτάμε ποια θα ήταν μια σωστή δίκαιη μαύρη λίστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ήταν κάτι επαναστατικό υπό την έννοια ότι επιτέλους λαμβάνουν υπόψη ότι επιζήμιες φορολογικές ε, πρακτικές και η μηδενική φορολόγηση είναι ε, κάτι το οποίο προκαλεί μεγάλες απώλειες και ε, εμείς στην Oxfam χαιρετήσαμε αυτή την απόφαση της μαύρης λίστας αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει τα κριτήρια να είναι αντικειμενικά και χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις και χωρίς συμφέροντα γιατί από εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα ε, θα δείτε λοιπόν ότι δεν είναι πάρα πολύ μεγάλος ο ενθουσιασμός μου για τη μαύρη λίστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς αυτά τα τρία που σας είπα δεν έχουν γίνει σεβαστά. Ε, ε, κυρίως οι μικρές χώρες είναι αυτές που βρίσκονται οι Βερμούδες, οι Βρετανικές Παρθένες νήσι κτλ και βλέπουμε και χώρε φτωχέ και μεσαίου εισοδήματο που αναφέρονται μόνο και μόνο επειδή δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπα του ΩΣΑ που δεν συμμετέχουν. Ενώ άλλες χώρες ε, εκφεύγουν από μια μαύρη ή γκρίζα λίστα όπως είναι Βραζιλία. Και τέλος η διαδικασία που οδήγησε σε αυτή τη λίστα ήταν πάρα πολύ αδιαφανής. Και ο τρόπο με τον οποίο καταρτίστηκε παρόλο που ε, έχουν ε, γίνει κάποιες καλέ κινήσει, όπω είπε και ο κ. Μορταλιέ. Και ασχολείται μόνο με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό βλάπτει πάρα πολύ την αξιοπιστία, διότι οι κάτω χώρες, ε, η Μάλτα, η Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο δεν ε, ανταποκρίνονται σε κριτήρια δίκαιης φορολόγησης. Πάντως είναι χρήσιμο αυτό το εγχείρημα της μαύρης λίστας γιατί γίνεται μια συζήτηση ε, για μεδενικό φορολογικό συντελεστή που δεν γινόταν μέχρι τώρα. Επίση, και τι γίνεται με τις επιζήμιες πρακτικές εξετάζει και μπορούν οι χώρε στην κρίζα λίστα να αλλάξουν την ομοδοσία του. Αλλά και πάλι εδώ είμαστε επιφυλακτικοί. Η ομάδα για τον κώδικα δεοντολογίας 20 χρόνια ήδη ελέγχει όλες αυτές τις χώρες. Ε, υπάρχουν κάποια καθεστώτα που έχουν ε, κάποιες χώρες που έχουν αλλάξει νομοθεσία τους, αλλά το Βέλγιο ε, χρησιμοποιεί ε, φορολογικά κίνητρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα πεδίο ε, με ίδιους κανόνους ε, παιχνιδιού, αλλά αυτό δεν θα καταργήσει ε, τους φορολογικούς παραδείσους. Χρειάζονται επιγόντως αλλαγές. Έρχομαι τώρα στην απάντηση που πρέπει να δώσω. Πώς μπορεί να βελτιωθεί αυτός ο κατάλογος για να αντιμετωπιστούν καλύτερα επιζήμιες πρακτικές. Θα πρέπει να αναθεωρηθούν τα κριτήρια της ομάδας για τον κώδικα δεοντολογίας γιατί δεν συμπεριλαμβάνει όλες τις φορολογικές πρακτικές. Επίσης, οικονομικοί δείκτες θα πρέπει να ενισχυθούν ε, η Γενική Διεύθυνση Ταξούτ στα τέλη του 2017 έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη για το ευρωπαϊκό εξάμεινο όταν αξιολογούσαν τα 7 κράτη-μέλη που έχουν επιζήμιες ε, τέτοιες φορολογικές πρακτικές. Άλλη σύσταση, να βελτιωθεί ο μαύρος κατάλογος με μεγαλύτερη διαφάνεια, αποτελεσματικότητα, αλλά και παγκόσμια αντιμετώπιση στα πλαίσια του ΟΗΕ. Η σύσταση θα ήταν να ζητήσουμε από το Συμβούλιο να κοιτάξουν πώς μπορεί να γίνουν πραγματικές αλλαγές στις χώρες αυτές. Να υπάρχουν διάφορες κυρώσεις επίσης ε, που να επιβάλλονται ανάλογα με το ποιο κριτήριο δεν γίνεται σεβαστό, ας πούμε. Επειδή η Μογγολία δεν έχει επιβάλει τα ελάχιστα πρότυπα ε, του BEPS, δεν θα υποστεί τις κυρώσεις. Αλλά οι Βερμούδε, α πούμε, που είναι από τους μεγαλύτερους φορολογικούς παραδείσους. Για μά σημαντικότερη σύσταση, η μαύρη λίστα δεν θα πρέπει να είναι μια πρόφαση για να μην γίνουν βαθιές φορολογικές μεταρρυθμίσεις για τη φοροαποφυγή. οι ε, Ηνωμένε Πολιτείε έχουν ένα το φορολογικό συντελεστή, εμεί γιατί δεν το έχουμε κάνει. Ή η έκθεση αναχώρα, ε, γιατί έχει ε, μπλοκαριστεί στο Συμφούλιο. Και τελικά η ενοποιημένη κοινή βάση φορολόγηση επιχειρήσεων, το CCCTV. Γιατί όλα αυτά δεν έχουν εφαρμοστεί, να μην χρησιμοποιείται η μαύρη λίστα ως πρόφαση για να γίνονται κάποια πασαλήματα στα θέματα των φορολογικών πρακτικών. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε όλους τους ομιλητές. Μπορεί να ξεκινήσει η συζήτηση με τους βουλευτές. Πέντε λεπτά αναερώτηση κάθε φορά, όπου θα έχουμε την παρέμβαση, την ερώτηση μάλλον του βουλευτή και έπειτα την απάντηση του ομιλητή. Σας ζητώ να είστε σύντομοι με τις ερωτήσεις προκειμένου να ακούσουμε και τις απαντήσεις και να καλύψουμε και τους δώδεκα ομιλητές. Πέντε λεπτά λοιπόν αναερώτηση. Ο συνηγητή εξ του ΕΛΚΟ, κύριο Νίντερ Μάιερ, έχει πρώτο το λόγο. Σα ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ σήμερα. Εγώ δεν θα επικεντρωθώ τόσο πολύ στον κατάλογο αυτό, στου άλλου καταλόγου. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι ο απότερο στόχο. Ο απότερο στόχος είναι να ενθαρρύνουμε την αλλαγή συμπεριφορά των χωρών εκείνων που δεν συνεργάζονται αυτή τη στιγμή προκειμένου να αρχίσουν να συνεργάζονται πιο υπεύθυνα σε φορολογικά ζητήματα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο δημιουργήθηκε και η μαύρη λίστα και πιστεύω ότι προκειμένου να είμαστε πιο αποτελεσματικοί το να εισάγουμε ή να βγάζουμε κάποιον από τη λίστα θα πρέπει να γίνεται με τρόπο διαφανή και με τρόπο αποτελεσματικό. Θα πρέπει να είναι σαφή τα κριτήρια επίσης ε, ένταξης μιας χώρας στη μαύρη την κρίζα λίστα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο έγγραφο συζήτηση, στο έγγραφο προβληματισμού μάλλον του 2016 εξηγεί ποιες θα ήταν οι πιθανές κυρώσεις που θα μπορούσαν να ισχύσουν, οι επιπτώσεις ε, όπως θα μπορούσε να πει κανεί. Θεωρώ πάντως ότι οι επιπτώσεις αυτές, οι κυρώσεις είναι αρκετά περιορισμένες. Νομίζω ότι ε, από το να συμπεριλαμβάνουμε τελικά μία χώρα στο κατάλογο αυτό, καταλήγουμε πολύ συχνά στο να υπάρχει απλώς ένας συντονισμός των εθνικών αρχών. Και το πρόβλημα είναι ότι ακόμα και μετά την ένταξη στο κατάλογο αυτό δεν είναι οι επιπτώσεις. Αυτό δεν αποδυναμώνει την αποτελεσματικότητα του ίδιου του καταλόγου. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, αν υπάρχουν ε, σημαντικές ε, διακυμάνσεις ως προς την αντίδραση των ε, κρατών που συμμετέχουν στον κατάλογο αυτών, που έχουν ενταχθεί μάλλον στον κατάλογο. Ξέρετε ότι κάποιες χώρες μπορεί να αντιδράσουν πολύ έντονα και αρνητικά, πάλι όχι. Αυτό δεν θα επηράσει και τις ίδιες τις φορολογικές πολιτικές γιατί καταλαβαίνετε ότι ακόμα και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί τελικά στα πλαίσια μιας αρνητικής αντίδρασης κράτους μέλους να έχουμε από το κράτος αυτό μια πιο θετική συνεργασία με φορολογικό παράδεισο τελικά. Αυτό από μόνο του θα αποδυναμώσει τον κατάλογο. Ευχαριστούμε πολύ. Ποιος θέλει να απαντήσει μόνος, πρώτος, με συγχωρείτε, ο κύριος Μηταγρία έχει το λόγο. Θα ξεκινήσω εγώ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, Επ' αυτού όντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα περίμενε πιο ταχεία αποτελέσματα και καλύτερη πρόοδο. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να κινητοποιήσουμε την κοινοτική χρηματοδότηση. Ας μην υποτιμούμε την επίπτωση αυτής της χρηματοδότησης. Ήδη έχουμε πετύχει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ήδη αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, υπάρχουν δύο επίπεδα κυρώσεων νομοθετικά και διοικητικά, αυτά είναι πολύ σημαντικά για τη βιωσιμότητα της όλης διαδικασίας. Βραχυπρόθεσμα τώρα, μόνο και μόνο το πλήγμα στη φήμη μιας χώρας, του να συμμετέχει στον μαύρο, στον γκρι κατάλογο τελικά. Ήδη αυτό από μόνο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ουσιαστικό ασκούμε πίεση κατά αυτόν τον τρόπο τώρα πρόθεσμα, τον έχουμε μία συντονισμένη προσέγγιση με κάποιες ελάχιστες κυρώσεις και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για ποιο λόγο? Γιατί υπάρχει κάτι το οποίο δεν θέλουμε να διακινδυνεύσουμε. Η ελευθερία που προέβλεπουν οι συνθήκες και η εσωτερική αγορά. Υπάρχει όμως διαφορά ανάμεσα στο να είμαστε πάρα πολύ απόλυτοι όσον αφορά τις ελευθερίες που προβλέπουν οι συνθήκες και η κατάχρηση έπειτα των ελευθεριών αυτών όσον αφορά την φορολογική πολιτική. Αν λοιπόν πραγματικά θέλουμε να διατηρήσουμε την πίεση και έπειτα να καταφέρουμε παράλληλα με την πίεση αυτή που ασκούμε στις χώρες αυτές να έχουμε και τις ελευθερίες που προβλέπονται από τις συνθήκες για την ελευθερία εγκατάστασης, κινητικότητας κτλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μια κοινή στάση από τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη αποφάσισαν όσον αφορά το πρώτο στάδιο να υποβάλουν αιτήσει στην ομάδα του κώδικα δεοντολογίας κάποιες χώρες μας είπαν ότι θέλουν να δούνε πώς χρησιμοποιούν τον κοινοτικό κατάλογο και τον εθνικό κατάλογο στα αντίμετρα τα οποία θα υιοθετήσουν και αναμένουμε να δούμε πραγματικά τις εκθέσεις αυτές από τα κράτη-μέλη για να δούμε πώς χρησιμοποιούν τους καταλόγους αυτούς. Σας ευχαριστούμε πολύ, ο κύριος Κόμπεν. Εφόσον έχουμε κατάλογο βάση κριτηρίων, προφανώς ε, ε υπάρχει ε, επικέντρωση στις χώρες χαμηλότερου εισοδήματος. Γι' αυτό και είμαστε επιφυλακτικοί. Γι' αυτό όμως πρέπει όμως να, είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά ε, την αντίδραση που θα, ε, που θα προκύψει από αυτές τις χώρες χαμηλού εισοδήματος. Γιατί αυτό δεν θα φέρει και τα επιθυμητά αποτελέσματα. Αντίθετα, πρέπει να ενθαρρύνουμε μεγαλύτερη φορολογική διαφάνεια από τους φορολογικούς και να τους αναγκάσουμε αν δεν, τους, αν δεν το κάνει ε, η χώρα στην οποία έχουν τις δραστηριότητες τους και την έδρα τους. Άρα πρέπει να δώσουμε κίνητρα για μεγαλύτερη διαφάνεια και ταυτόχρονα να προκαλέσουμε πολιτικές αντιδράσεις ε, στην ίδια την ε, χώρα, στην τρίτη χώρα. Κατά τη στοιχεία η ΕΠΑ αναγκάζουν όλες τις χώρες να έρχονται σε διαπραγμάτευση μαζί τους προκειμένου να μπορούν να, οι εκάστοτε εταιρείε που έχουν την έδρα τους σε τρίτες χώρες να μπορούν να δραστηριοποιούνται στις ΗΠΑ. Κάτι τέτοιο λοιπόν πρέπει να γίνει και εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να εξασφαλιστεί το επίπεδο διαφάνειας και συμμόρφωσης με την νομοθεσία που επιθυμείται. Αυτό το ζήτημα λοιπόν του σχεδιασμού ε, ως προς τη χάραξη της ευρωπαϊκής πολιτικής είναι ζωτική σημασίας. Ευχαριστώ και τους ομιλητές. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι παρεμβάσεις. Ξέρω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο, οπότε θα ξεκινήσω με την αντίθετη σειρά. Το κύριο Λάγκεροκ. Είπατε για, τους, για το CCTV, για, την, για τις εκθέσεις αναχώρα. Είπατε ότι όλα αυτά πρέπει να εφαρμοστούν πλήρως για να αντιμετωπιστεί η φοροποφυγή. Όμως, κατά τη γνώμη σας, είναι εφικτό αν θέλετε, να μιλήσουμε για αποτελεσματική καταπολέμηση της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής χωρίς να υπάρχει δημόσια ε, υποβολή εκθέσεων αναχώρα. Και τονίζω το δημόσια. Ε, ε, χρειαζόμαστε ένα τέτοιο εργαλείο θεμελιωδώς προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει συνεργασία ώστε να, να αναγκάζονται οι πολυεθνικές να ε, δηλώνουν τα κέρδη τους και πού τα έχουν ε, πραγματοποιήσει. Κύριε Κόμπαν, βάσει της αξιολόγησής σας, ε, έξι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κύπρος, Μάλτα, Λουξεμβούργο, κάτω χώρες, Ενωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία ανήκουν κανονικά ή θα έπρεπε να ανήκουν στον μαύρο κατάλογο αν είχαν εφαρμοστεί σε αυτές τα ίδια κριτήρια. Επομένως, αν ο ισχύων μαύρος κατάλογος, ο οποίος βεβαίως δεν περιλαμβάνει ε, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν λοιπόν τώρα το, Ευρω... το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει της δικής αξιολόγηση δεν θα πρέπει να προσθεθεί στο μέλλον σε αυτό το μαύρο κατάλογο. Ε, θα είναι και ένα, μία από τις, ε, τις ε, επιπτώσεις αυτό, μια τέτοια εξέλιξη εν του Brexit ή μάλλον μετά το Brexit. Επίσης, είπατε ότι η Κομισιόν έχει κάποια εργαλεία στη διάθεσή της όσον αφορά την επιβολή κυρώσεων σε μη συνεργάσιμε δικαιοδοσίε. Μπορείτε όμως να δώσετε περισσότερες πληροφορίες για το τι είδου εργαλεία μπορεί κανείς να εφαρμόσει ω ε, ως Κομισιόν έναντι τρίτων χωρών που βρίσκονται στο μαύρο κατάλογο. Μπορείτε να αναλάβετε δράση και εναντίον εταιριών ή προσώπων που βρίσκονται σε αυτές τις τρίτες χώρες. Ε, δηλαδή σε αυτό το μαύρο κατάλογο, αυτός ο μαύρος κατάλογος σας επιτρέπει να, να αναλαμβάνετε δράση ε, ενάντια σε χώρες ή και σε εταιρείε. Ευχαριστώ. Ε, μία συμφωνία είναι αυτή που μας προτείνεται δηλαδή με δύο λόγια. Για την ε, υποβολή εκθέσεων αναχώρα. Είναι θεμελιώδης ε, ε θεμελιώδες αυτό το στοιχείο για την λογοδοσία τόσο των ε, τρίτων χωρών όσο και των μεγάλων πολυεθνικών και έχει αποδειχθεί στο παρελθόν ότι μια τέτοια διαδικασία βοηθά και τις χώρες στο να αλλάζουν, να αλλάζουν τις φορολογικές πρακτικές. Γι' αυτό και δεν καταλαβαίνω γιατί το Συμβούλιο επιμένει στη στάση στην οποία έχει τηρήσει μέχρι στιγμής. Όσον αφορά τις ελαρμονισμένους ε, κανόνες για την ενοποιημένη φορολογική βάση των εταιριών. Μπορούμε πάντα να μιλούμε για στοχευμένε κυρώσει κτλ. Μα υπάρχει ήδη ο, κανον, ο CFC που προβλέπει ότι που προβλέπει ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, εναρμονισμένος τρόπο ε, εφαρμογής αυτών των κανόνων. Πρέπει λοιπόν ε, να υπάρχει εναρμόνιση και από εκεί και πέρα θα υπάρχει ένα ενοποιημένος ελάχιστο φορολογικό συντελεστή για κέρδη που έχουν επιτευχθεί στο εξωτερικό. Να πω πρώτον ότι λυπάμαι για το Brexit. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα υποφέρει. Ήδη βλέπουμε ότι υφίσταται σημαντικές οικονομικές συνέπειες και άλλες ε, προφανώς μάλλον. Εμείς ε, ως το δίκτυό μας ήμασταν αντίθετοι. Τώρα προσπαθούμε να βρούμε τη χρυσή τομή. Το Ηνωμένο Βασίλειο ε, θα φύγει, το Ηνωμένο Βασίλειο που μπλοκάρει σε πολλά θέματα και στα φορολογικά. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να ε, προχωρήσει περισσότερο και αυτό θα είναι προς όφελος και του λαού του Ηνωμένου Βασιλείου. Και σε τελική ανάλυση υπέρ της χώρας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα κριτήρια, αν είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, προφανώς θα ήταν ε, στη λίστα. Αλλά η έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση μειώνει και την ελκυστικότητα του Ηνωμένου Βασιλείου ως ε, τόπου μεταφοράς των κερδών και γενικότερα ως οικονομική δραστηριότητα. Ε, Κύριε Μοχτάλια, ε, σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις που ρωτήσατε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμείς ουσιαστικά τι έχουμε περισσότερο νομοθεσία, νομοθεσία ε, αυτό τον καιρό που εκπονείται για τις δημόσιες εκθέσεις αναχώρα για περισσότερη και βαθμια ε, και ε, νομιμοποίηση χωρών που είναι τώρα σε φορολογικούς παραδείσμα εταιρεών Έχουμε την οδηγία ΜΥΦΙΤ. Ελπίζω οι δύο συνεισηγητές να μας βοηθήσουν για τον κανονισμό αυτό. Ε, έχουμε επίσης την ανάλυση για την δυστυχία ε, και ε, την ευρωπαϊκή οικονομική υποστήριξη. Αυτή είναι οριζόντια, εγκάρσια νομοθεσία. Βεβαίως, όταν πρόκειται για συμμετοχή στα συμβούλια τα διοικητικά διεθνών οργανισμών όπου θα έχουμε λόγο για το ε, εάν και κατά πόσο μια χώρα ή μια, μια εταιρεία συμμορφώνεται ως εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουμε λάβει, θα λάβουμε μάλλον αποφάσεις που θα επηρεάσουν συγκεκριμένες επιχειρήσεις, συγκεκριμένα πρόσωπα. Αλλά εμείς δρούμε μέσω της νομοθεσίας, μέσω της παρακολούθησης και της υλοποίησης της νομοθεσίας. Αυτή είναι η δική μας δράση. Ευχαριστώ. Ο Μάρκους Φέρμπερ από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ και καιρό το συζητούμε αυτό το θέμα των μαύρων ε, καταλόγων και χαρήκαμε πάρα πολύ που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατήρθησε και υπέβαλε μια μαύρη λίστα η οποία ε, όπως και να το κάνεις από 210 κράτη που υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο καταλαβαίνετε και τα γερμανικά μου ή να τα πω σε κακά αγγλικά όχι, καλύτερα στα γερμανικά. Έλεγα λοιπόν ότι από τα 200 τόσα κράτη που υπάρχουν στον κόσμο, 17 αναγράφονται, <laughs> καταφέρατε να συγκεντρώσετε στη μαύρη λίστα. Και σε σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε το Συμβούλιο να φέρει σε 8 κράτη. Σήμερα διάβασα στην ε, τοπική μου εφημερίδα ότι μια μεγάλη επιχείρηση fast food έχει τέτοια κατακαιρματισμένα ε, ε, ε, παραρτήματα, πώς να το πω, σε χώρες που έχουν αφαιρεθεί από τον κατάλογο, που δεν θα πληρώνει φόρο καθόλου. Και ποια είναι αυτά τα κριτήρια για να βγεις από τη λίστα. Και έχω μια πολύ απλή ερώτηση. Το σύστημα αυτό είναι αποτελεσματικό της μαύρης λίστας ή μήπως να το καταργήσουμε καλύτερα. Δηλαδή 17 μείον 8 κάνω μέσω μέσω στην αφαίρεση 9, 9 κράτη από τα 210 του κόσμου τούτου. Έχουμε διαδικασίε ελέγχου και παρακολούθησης. Ποιε είναι αυτές οι χώρες, οι δικαιοδοσίε έχει αλλάξει τίποτα εκεί. Σχέδια έχετε εσείς. Και αυτό απευθύνεται προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να επιβάλλετε κυρώσεις για τι χώρε που γράφονται στον κατάλογο αυτό ή μήπω υπάρχει, ε, υπάρχει μέθοδος να προσθεθούν και άλλες χώρες. Τι πρέπει να κάνεις για να μπει στη λίστα. Γιατί από ό,τι φαίνεται μάλλον η μόνη δυνατότητα που υπάρχει να φερούνται χώρες από τη λίστα. Και αυτά που ζήσαμε ε, στα τέλη του περασμένου και αρχές του τρέχοντος δεν αύξησαν την ε, εμπιστοσύνη στη μαύρη λίστα. Αλλά φαίνεται ότι και η μεγαλύτερη φορολογική αμαρτωλοί, ας πούμε, θεωρούνται σεβαστά κράτη από πλευρά Συμβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και ε, θα ήθελα να μάθω πώς φαντάζεστε ότι θα εξελιχθούν όλα αυτά μακροπρόθεσμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε να απαντησουμε πως Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ενδεχομένω και κάποιο άλλο μετά, η κυρία Βάντεν Βέλτεν, ενδεχομένω θα μπορούσε να απαντήσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντω πρώτη. Σα ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις αυτές. Κοιτάξτε, σε ένα βαθμό μπορώ να καταλάβω την έκπληξη ορισμένων ενδιαφερομένων οι οποίοι βλέπουν πώς διακυμμένονται τα πράγματα και πώς έχει εξελιχθεί η λίστα αυτή με την πάρδο του χρόνου. Αυτό έχει να κάνει με συγκεκριμένε επιλογέ που έκανε το Συμβούλιο να βγάλει κάποιες χώρες από τον κατάλογο βάσει των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει. Και νομίζω ότι αυτό είναι κατανοητό, τουλάχιστον στην αρχή της διαδικασίας, το είπε αυτό και ένας ομιλητής πριν από λίγο. Ο απότερος στόχος είναι να δώσουμε κίνητρα προκειμένου να αλλάξει φορολογική συμπεριφορά και να καταλήξουμε σε μια δέσμευση για αλλαγή βασικά, για μεταρρυθμίσεις. Η επιλογή λοιπόν του ΕΚΟΦΗΝ ήταν να περάσει κάποιες δικαιοδοσίες, κάποιες χώρες από τη μαύρη λίστα σε έναν άλλο κατάλογο που τις παρακολουθούμε περισσότερο σε σχέση με τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, ιδίως στην αρχική φάση, τα πρώτα χρόνια δηλαδή, και αναφέρομαι εδώ πέρα σε αυτά που είπε και ο συνάδελφος από την Oxfam. Σε καμία περίπτωση δεν γλιτώνει κάποια χώρα από τίποτα. Ουσιαστικά ανέλαβαν δεσμεύσεις, αυτό έγινε και εξακολουθούν να βρίσκονται υπό επιτήρηση μέχρι τα τέλη του έτους για να δούμε τελικά αν όντως θα τηρήσουν και σε ποιο βαθμό τις δεσμεύσεις τους. Αν θέλετε να συγκρίνουμε αριθμητικά δεδομένα πόσες χώρες βρίσκονται στον κατάλογο του δικτύου φορολογικής δικαιοσύνης, 92 έχουμε εμείς. Εμείς αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε την κατάσταση 92 χωρών. Ορισμένες δεν δεσμεύτηκαν, άλλες πάλι ανέλαβαν δεσμεύσεις και εμείς ε, εξακολουθούμε και τις επιτηρούμε με πάρα πολύ μεγάλη αυστηρότητα. Και από την άλλη ο πρόεδρος του ΕΚΟΦΗΝ πριν από μερικές εβδομάδες έστειλε μια επιστολή στον ΩΣΑ ζητώντας το φόρουμ για τις επιβλαβείς φορολογικές πρακτικές του ΩΣΑ να διασφαλίσει ότι τα νέα στοιχεία της φορολογικής μεταρρύθμισης των Πολιτειών θα τύχουν ε, επιτήρηση στα πλαίσια του φόρουμ αυτού για τις επιβλαβείς πρακτικές. Λοιπόν, θα πρέπει να είμαστε σαφείς. Η παρακολούθηση, η επαγρύπνηση εξακολουθεί και υφίσταται για τις 92 αυτές χώρες και κάθε φορά λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός στον οποίο ανέλαβαν δεσμεύσεις και ο βαθμός στον οποίο τηρούν και εκπληρούν αυτές τις δεσμεύσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει την εργασία, την παρακολούθηση των δεσμεύσεων αυτών. Στέλνουμε τακτικές εκθέσεις στην ομάδα κώδικα δεοντολογίας, ο οποίος πριν το καλοκαίρι θα συντάξει μια ενδιάμεση έκθεση όπως έχουν ζητήσει οι Υπουργοί στα συμπεράσματα του Δεκεμβρίου Κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί για κάποιες από τις χώρες αυτές να κινητοποιηθεί η διαδικασία της έγκαιρης προειδοποίησης και ενδεχομένως να χρειαστεί για κάποιες από αυτές να ληφθούν και διορθωτικά μέτρα. Επομένως, αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι έχουμε ένα δέντρο το οποίο κρύβει το δάσος. Σαφώς έχουμε ένα συγκεκριμένο κατάλογο Βλέπουμε ποιες είναι οι χώρες οι οποίες δεν θέλουν να συνεργαστούν και αυτές βρίσκονται στον κατάλογο. Για όλες οι υπόλοιπες που έχουν αναλάβει δεσμεύσεις παρακολουθούμε τις τάσεις τους και τις μεταρρυθμίσεις τους μέχρι το τέλος του έτους. Η κυρία Βέλντε. Ένας μικρός μαύρος κατάλογος μπορεί να αποτελέσει ένα είδος άσκηση πολιτικής πίεσης και μπορεί να αποβεί τελικά πιο αποτελεσματικός από κάποια άλλα μέτρα. Και όντω, όπως υπόθηκε, είναι πάρα πολύ σημαντικό εν συνεχεία να βλέπουμε ακριβώ αν τηρούν τις δεσμεύσεις τους τα κράτη. Και εγώ θα μιλήσω γερμανικά. Πρώτα απ' όλα, κατανοούμε όλη την πολιτική κατάσταση στην οποία βρίσκεστε και αν όπως ο συνάδελφος Κόφωτ και εγώ ε, συμμετέχει κανείς από την πρώτη Εξεταστική Επιτροπή τάξη 1 και όταν ε, ε, έχει λάβει γνώση βεβαίως και τη κατάσταση που επικρατεί εντό αυτή τη ομάδα για το Code of Conduct, καταλαβαίνουμε τι δυσκολίε που αντιμετωπίζει Κομισιόν και τα αναγνωρίζουμε αυτά. Αναγνωρίζουμε επίση όλοι ότι πρόκειται για μια ευφυή διαδικασία. Οι χώρε που δείχνουν κάποια προθυμία να αλλάξουν κάποια πράγματα στα φορολογικά του συστήματα να λαμβάνουν κάποια κίνητρα προκειμένου να είναι πιο συνεργάσιμα. Ε, γι' αυτό και είναι, είναι, είναι κατανοητή αυτή η προσέγγιση της κατάρτισης και ενός γκρίζου καταλόγου. Επίσης χαιρετίζω το γεγονός ότι είπατε ότι, θα, ότι έχετε σκοπό να, να δημοσιεύετε εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο που σημειώνουν συγκεκριμένε χώρες που έχουν δηλώσει την προθυμία τους να είναι πιο ε, συνεργάσιμες. Όμως αυτό που μου λείπει εμένα ως κοινοβούλιο είναι ποια είναι, ε, ποια είναι ακριβώς η δομή, μια διαφάνεια ως προς τη δομή. Τι ακριβώς δηλαδή αναμένω, περιμένω, τι συγκεκριμένα περιμένω από, ένα, ε, από μια χώρα που έχω εντάξει στο μαύρο κατάλογο για να την βγάλω από το μαύρο κατάλογο. Εδώ ε, ε, εγώ έχω εργαστεί πάρα πολλά χρόνια στα διορθωτικά ταμεία κτλ. Είστε πραγματικά πρωταθλητές παγκόσμιοι στο να αξιολογείτε και να ε, ε, παρουσιάζετε με διαφάνεια όλα τα στοιχεία. Και σε αυτόν τον τομέα έχουμε μηδέν πληροφορίες, τίποτα, σχετικά με την μεθοδολογία και το συγκεκριμένο ερώτημα δηλαδή σε ποιο σημείο ποιο, ποιου κριτηρίου, ποια χώρα εκπληρώνει τι και τι δεν εκπληρώνει. Αυτό νομίζω ότι ήταν, είναι το, το α και το ω κάθε αξιολόγηση κανονικά. Και γι' αυτό θέλω το να θέσω το ερώτημα προς εσάς. Η Κομισιόν είναι διατεθειμένη ή έχοντας υπόψη μας και τη σχέση σας με, την Code με το Code of Conduct Group μπορείτε να επιτύχετε αυτή τη μορφή διαφάνειας ή να μην περιμένουμε κάτι τέτοιο. Γιατί είναι τόσο σημαντικό να λάβουμε αυτή τη διαφάνεια σε αυτή την έκταση. Διότι όσο δεν υπάρχει αυτή η διαφάνεια θεωρεί ο καθένας ότι πρόκειται απλά για πολιτικές προφάσεις. Ε, μπορεί και να μην είναι έτσι τα πράγματα. Ε, αλλά όσο τα πράγματα είναι μη κατανοητά τότε αυτή η υποψία δεν πρόκειται να διασκεδαστεί ποτέ αυτό. Ένα ερώτημα προς, προς την Oxfam. Είπατε ε, να καταρτιστεί και ένας κατάλογος φορολογικών παραδείσων που θα περιλαμβάνει και ευρωπαϊκές χώρες. Συγκεκριμένα πώς ακριβώς πιστεύετε ότι μπορεί αυτό να γίνει. Πρακτικά, τελευταίο ερώτημα προς, προς τον συνάδελφο από την Κομισιόν. Κατανόησης. Βγήκα λίγο έξω από την αίθουσα, δεν ξέρω αν το είπατε. Για ποιο λόγο φορολογική παράδοση, όπως για παράδειγμα η Σιγκαπούρη, που λειτουργούν ως αγωγή φορολογικών παραδείσων, δεν τοποθετήθηκαν, δεν ε, εντάχθηκαν σε αυτό το μαύρο κατάλογο. Ευχαριστώ. 1,5 λεπτό για τις απαντήσεις έχουμε πλέον. Η Κομισιόν και η Oxfam. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα γιατί έχω ένα λεπτάκι μόνο. Βεβαίως πάντα είναι δυνατές οι πρόοδοι. Και από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής εμείς ανέκαθεν πιέζαμε όσο γινόταν περισσότερο για τη διαφάνεια. Ε, δημοσιεύσαμε το βαθμολόγιο μας, ε, γνώρισε αυτό μεγάλες αντιδράσεις και δυσφορίες. Όπως σας είπα, ο Επίτροπος Μοσκοβισή ε, επέμεινε να είναι δημόσιες οι αναφορές και αναχώρα και, και μάλλον οι δεσμεύσεις αναχώρα. Υπάρχουν κάποια κριτήρια γιατί αναγράφεται η χώρα στον κατάλογο, γιατί έχει πρόβλημα διαφάνιση, γιατί έχει ένα ε, καθεστώτα και συστήματα που επιτρέπουν κάποιες καταστάσεις. Είναι δημόσιες λοιπόν αυτές οι επιστολές που έχουμε στείλει σε όλα αυτά τα κράτη και δημόσιες οι πληροφορίες γιατί αναγράφονται στο συγκεκριμένο κατάλογο ή τουλάχιστον ε, ποια είναι τα ε, θέματα στα οποία τους ζητούμε να δεσμευθούν. Ξέρουμε λοιπόν γιατί έχουν δεσμευτεί και εκεί μπορείτε να μας ζητήσετε το λόγο και να λογοδοτήσουμε για τον έλεγχο και την παρακολούθηση αυτών των δεσμεύσεων και των υποσχέσεων. Και η κοινή γνώμη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίξουν το ρόλο τους πιέζοντας αυτές τις χώρες για να κάνουν τις μεταρρυθμίσεις. Ε, λοιπόν, πιέζουμε μάλιστα έτσι ώστε... να γίνουν γνωστά και δημόσια και οι λόγοι ε, που μας κάνουν να ανησυχούμε αλλά και οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν οι χώρες αυτές. Μόνο έτσι θα βεβαιωθούμε ότι θα πληρωθούν αυτά όλα. Σιγκαπούρη και κάτω χώρες, έτσι έχω να απαντήσω εγώ. Ε, Μάλτα, Λουξεμβούργο και Ιρλανδία κλπ. Για τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη χαιρόμαστε που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τελευταίο ευρωπαϊκό εξάμεινο το ε, ανέφερε αυτό και το κατέδειξε. Είναι καλό, σωστό βήμα. Δεν χρειάζεται να αναθεωρηθεί μόνο ο κώδικας διαντολογίας και η αντίστοιχη ομάδα, αλλά και ο τρόπος λειτουργίας. Ε, γιατί δεν έχουν εντοπίσει αυτές ε, τις χώρες, ε, ως χώρες που έχουν ε, patent boxes όπως είναι η Ιρλανδία και οι κάτω χώρες, θα πρέπει να σταματήσουν αυτές οι διευκολύνσεις και η μειωμένη φορολόγηση των κερδών από ό,τι στο παρελθόν. Γιατί η Σιγκαπούρη ως αγωγός για φορολογικούς παραδείσους ναι, θα μπορούσε να είναι στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον κατάλογο, αλλά το κριτήριο 2.2 είναι πάρα πολύ ασαφές, το οποίο επιγράφεται ε, προσέλκυση κερδών που έχουν ε, παραχθεί εκτός offshore. Αυτό χρειάζεται μεγαλύτερη διευκρίνηση ως προς τον ορισμό, γιατί είναι πολύ ασαφές και γενικόλογο. Τι θα πει attracting offshore profits. Ευχαριστώ πολύ. Το ECR ο πρώτος αντιπρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω καταρχάς ομιλητές. Σας ζητώ συγγνώμη που έφτασα με καθυστέρηση. Ήμουνα στην Επιτροπή Μεταφορών, στην οποία εργάστηκα για πολλά χρόνια συντονιστή και το αναφέρω αυτό γιατί και στα πλαίσια τη αεροναυτιλία ξέρετε ότι υπάρχει ένα μαύρο κατάλογο όσον αφορά τι αεροπορικέ εταιρείε αν ενταχθεί κανείς στον κατάλογο αυτό, ουσιαστικά δεν μπορεί καμία πτήση να γίνει στον ενέριο χώρο σας. Ή ξέρετε ότι σε ορισμένε περιπτώσεις, ορισμένες χώρες υπολείπονται των δεσμεύσεων που έχουν σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Αεροναυτιλίας. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή οι εταιρείε οι οποίε φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτε χώρε είναι εταιρείε οι οποίε πληρούν τα κριτήρια τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτέ οι οποίε συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια τη Αεροναυτιλία. Και ξέρετε ότι ανατακτά χρονικά διαστήματα παρακολουθούμε την τήρηση των κανόνων αυτών και αναλόγω ο μαύρο αυτό κατάλογο επικαιροποιείται. Το αναφέρω αυτό σε σύγκριση με τον κατάλογο τον οποίο συζητάμε εμεί αυτή τη στιγμή. Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να έχουμε και κάποιου εμπειρογνώμονε όσον αφορά τον φορολογικό μαύρο κατάλογο τον οποίο εμεί χρησιμοποιούμε. Διαφορετικά είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσουμε στου πολίτε πώς ακριβώς λειτουργεί ο κατάλογος αυτός. Είχα πάει σε μια αντιπροσωπεία σε χώρες της Μέσης Ανατολής, οι οποίες βρισκόντουσαν στον κατάλογο αυτό των μη συνεργαζόμενων επικρατιών. Πολλές από τις χώρες αυτές θέλανε να βγουν από τον κατάλογο αυτό και μία από αυτές, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, θέσπισαν πλέον ένα φόρο προστιθέμενης αξίας της τάξης του 5%, το οποίο δεν υπήρχε στο παρελθόν. Αλλά ξέρετε ότι η χώρα αυτή, όπως και άλλες χώρες, στις οποίες δεν καταβάλλονται σημαντικές φορολογικές συνεισφορές, μπορεί να έχουν βγει ένα από κάποιο μαύρο κατάλογο, αλλά βρίσκονται σε έναν γκρίζο κατάλογο και γι' αυτό το λόγο βρίσκονται υπό την επιτήρηση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριε Μουταγλιέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ε, εξηγήσεις τις οποίες μας δώσατε, για το πώς παρακολουθείτε τις 92 αυτές χώρες αλλά μήπως μπορούμε να κάνουμε και πιο σημαντικά πράγματα σε πολιτικό επίπεδο. Πρόσφατα η χώρα μου, η Λετωνία, προσπάθησε να επικαιροποιήσει την νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις. Προφανώς υπάρχει μια κοινοτική οδηγία την οποία εφαρμόζουμε και έπρεπε να καλύψουμε και τις offshore εταιρείε. Και χρειάστηκε να ασχοληθούμε βέβαια και με κάποιες εταιρείε του λεγόμενου μαύρου καταλόγου. Και Κάποιοι δικηγόροι μας είπανε ότι ε, πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί γιατί εδώ πέρα καλείστε να εφαρμόσετε την κοινοτική οδηγία. Επομένω, δεν μπορείτε εσεί στα πλαίσια του μαύρου καταλόγου να δημιουργήσετε ένα επιμέρου πιο σύντομο κατάλογο με φορολογικέ επικράτειε με τι οποίε θα μπορούσατε να συνεργαστείτε και προ οποίε θα μπορούσατε να αναθέσετε δημόσιε συμβάσει. Γιατί εδώ πέρα ουσιαστικά διακυβεύονται τα χρήματα των φορολογουμένων. Θα μπορούσατε όμως να με εξηγήσετε στις περιπτώσεις αυτές τι θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς ως πολιτικοί θύνοντες Και θα ακούσουμε και την άποψη φαντάζομαι μη κυβερνητικών οργανώσεων. Θα απαντήσω στο πρώτο μέρο του ερωτήματο. Χαίρομαι που είπατε για τα καθεστώτα μηδενική φορολόγηση, γιατί το πρόβλημα αυτό δεν αντιμετωπίζεται επαρκώ αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι και το Συμβούλιο δεν γνωρίζει πώ ακριβώ μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα των δικαιοδοσιών με μηδενικούς φορολογικούς ε, ε, συντελεστέ. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν αυτέ οι επιζήμιε φορολογικέ πρακτικέ που είναι εύκολο να το αντιμετωπίσει κανεί. Ε, μπορεί να του πει φτιάξει αυτό και αυτό κτλ. Ε, κτλ. Με τους μηδενικούς φορολογικούς συντελεστές δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Γιατί δεν ξέρουμε πώς να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Δεν υπάρχει συντελεστής, δεν υπάρχει φορολογική αρχή. Τι κάνουμε λοιπόν με αυτά τα καθεστώτα μηδενική φορολόγηση ώστε να εξασφαλίσουμε ότι δεν προκαλούν ε, αποτελέσματα spillover σε άλλες χώρες κυρίαρχε οι οποίε θέλουν να, να διαμορφώσουν φορολογικά του συστήματα όπω θέλουν. Πρότασή μου θα ήταν να μην αρχίσουμε ε, να, προσθέτουμε κάποιες, ε, ε, κάποια κριτήρια, κάποιε διατάξει, Για παράδειγμα το να έχει δύο υπαλλήλου στι βερμούδε. Μια χαρά θα μπορούσε να το κάνει αυτή η, η Coca-Cola για παράδειγμα. Όχι, να εξασφαλίσουμε ότι τα κέρδη που πραγματοποιούνται στις Βερμούδες θα φορολογούνται με σοβαρές ε, ε, ε, διατάξεις καταπολέμησης φοροαποφυγής για να μπορεί να φορολογούνται τα κέρδη παντού. Δεν ξέρω βέβαια, μπορεί και να κάνω λάθος. Μπορεί οι Βερμούδες να προτίθενται και να, είναι διατεθειμένες να αλλάξουν ε, τις φορολογικές πρακτικές. Αυτό όμως ε, βεβαίως εξαρτάται από τις διαπραγματεύσεις στις οποίες θα προβεί το Συμβούλιο. Για τις δημόσιες προμήθειες προφανώς υπάρχει μια ενεργή διαδικασία, ε, συζήτηση γύρω από αυτή τη λετονική υπόθεση και το τι ακριβώς σημαίνει. Νομίζω ότι θα καταλήξουμε κατά πάσα πιθανότητα στο να πούμε ότι αντί να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα στο κατά πόσο αυτή η δικαιοδοσία αφορά το αν ήταν εξωτερικό, στο εξωτερικό η δραστηριότητα ή το κέρδος ε, πρέπει να το, να το ε, αντιμετωπίσεις στο πλαίσιο της κάθε, της, κάθε, της κάθε χώρας. Αλλά για να μπορείς να συμμετέχεις σε διαγωνισμούς ε, δημόσιων, δημόσιων προμηθειών θα πρέπει να εμφανίζεις ένα δεδομένο, ένα συγκεκριμένο επίπεδο διαφάνειας ώστε να εξασφαλίσουμε ότι όποια και αν είναι η δικαιοδοσία χωρ, εταιρείας η οποία συμμετέχει σε, σε κάποιον διαγωνισμό για δημόσιες προμήθειες θα πρέπει τουλάχιστον να εξασφαλίζεται ότι κάθε εταιρεία που συμμετέχει σε αυτό το διαγωνισμό να πληρεί κάποια ελάχιστα βασικά κριτήρια διαφάνειας. Θέλω να πω, εντάξει, δημόσιες προμήθειες, αλλά δεν μπορείτε να ελέγξετε από το, το, το, το Δήμο ε, ο Δήμος δηλαδή που κάνει τον κάθε διαγωνισμό δεν μπορεί να ελέγχει που, που, που έχει κάθε χώρα, την, κάθε εταιρεία την, την έδρα της. Okay, so the next... Λοιπόν, από τους Πρασίνους η Αντιπρόεδρο μας, η κυρία Ευαζολή. Ε, μια πρώτη ερώτηση. Προς τον κύριο Μουταχλιέ το Κοινοβούλιο στην σύσταση 187 της έκθεσης ΠΑΝΑ ζητεί να χρησιμοποιηθεί το άρθρο 116 για να καταθετεθεί νομοθετική πρόταξη και για να αλλάξει ο κώδικας δεντολογίας που θεωρούμε ότι δυσλειτουργεί σφόδρα. Εσείς είπατε ότι δεν πιστεύετε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν ε, αποτελεσματικός τρόπος μεταρρύθμισης. Θα μπορούσατε να μου δώσετε μια συμπληρωματική εξήγηση. Για ποιο λόγο το θεωρείτε αυτό τελέσφορο για την ε, μεταρρύθμιση του κώδικα δεντολογίας. Στη συνέχεια, έχω μια ερώτηση προς τον κύριο Λάγκεροκ. Στα αγγλικά. Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι η Oxfam κατατάσσει 35 ε, ε, χώρες στο μαύρο κατάλογο, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο 9. Θα μπορούσατε να μας δώσετε τη δική σας ανάλυση για ποιο λόγο η Βραζιλία δεν συμπεριλαμβάνεται στο συγκεκριμένο κατάλογο. you... Και ποιες είναι οι βασικές βελτιώσεις που θα συνιστούσατε στους ηθήνοντες και εκείνους που λαμβάνουν τις ευρωπαϊκές αποφάσεις για τη διαδικασία του μαύρου καταλόγου. Κύριος Μεταγλιέ πρώτος. Κύριε Ζολή, σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Μια ερώτηση που έχει μια έντονα πολιτική φύση Επομένως, δεν μπορώ παρά να επαναλάβω αυτό που είπε ο Επίτροπος Μοσκοβισή στο παρελθόν εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δύο ουσιαστικά είναι τα ζητήματα στο πλαίσιο της ερώτησής σας. Πρώτον, θα πρέπει να μεταρρυθμίσουμε ένα μέσο, το οποίο είναι ένα μέσο τελικά συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών, που και να γίνει αυτό το μέσο νομοθετικό τελικά. Και αν ναι, ποια θα είναι η κατάλληλη νομική βάση τότε γιατί αυτή τη στιγμή γίνεται μια νομοθετική πρόταση, τίθεται και το ζήτημα της νομικής βάσης. Προκειμένου τώρα να εξετάσουμε αν πραγματικά είναι σκόπιμο να αλλάξουμε νομοθετικό περιβάλλον, το πρώτο θέμα το οποίο θέτουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο οποίο πρέπει να απαντήσουμε είναι αν θα αυξηθεί τελικά η αποτελεσματικότητα του κώδικα διοντολογίας αν αλλάξει νομικό καθεστώς. Και όπως έχουμε πει ήδη στο Κοινοβούλιο, στο παρελθόν, έχουμε ξεκινήσει μια σφαιρική αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το φορολογικό ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά και του τρόπου με τον οποίο συμβάλλει η ομάδα του κώδικα διοντολογίας προκειμένου να δούμε αν τελικά το έργο της ομάδας αυτής τα τελευταία 20 χρόνια όντως έχει συμβάλει στο να εγκριθούν μέτρα τα οποία βάλουν κατά του φορολογικού ανταγωνισμού. Αυτό όντω έγινε. Καταφέραμε επίσης να συνεργαστούμε με χώρες όπως το Λίχτενστάιν, η Ελβετία. Κάναμε λοιπόν πρώτα μία αξιολόγηση των ζητημάτων αυτών για να δούμε τελικά αν χρειάζεται να αλλάξουμε νομικό καθεστώς, αν πρέπει να υποβληθεί μια πρόταση για να συσταθεί ένα άλλο μέσο και όπως είπε και ο Επίτροπος το άρθρο 116 της συνθήκης θέτει συγκεκριμένε προϋποθέσεις νομοθετικής φύσης ή και προϋποθέσεις όσον αφορά συγκεκριμένες πρακτικές στο πλαίσιο των κρατών μελών οι οποίες δεν μπορούν να αντικατασταθούν από τον κοινοτικό συντονισμό. Και αυτές οι προποθέσεις λοιπόν θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και στα πλαίσια της αξιολόγησης αυτής, η οποία θα πρέπει ουσιαστικά να επιτύχει τους στόχους της, το είπε και ο κύριος Μοσκοβισή, το πιο σημαντικό να καταλήξουμε τελικά σε ένα μέσο το οποίο θα είναι πιο αποτελεσματικό και όχι αναγκαστικά να αντικαταστήσουμε το μέσο αυτό. Ένα μέσο το οποίο έχει δώσει συγκεκριμένα αποτελέσματα μέχρι σήμερα. Να απαντήσω και εγώ στα ερωτήματα αυτά για ποιο λόγο υπάρχει διαφορά μεταξύ ΜΟΝ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοιτάξτε, εμείς δεν περιμέναμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα θέσπιζε και έναν γκρι κατάλογο. Αυτό άλλαξε τα δεδομένα. Εμείς δημιουργήσαμε τον δικό μας τον μαύρο κατάλογο χρησιμοποιώντας αντικειμενικούς οικονομικούς δείκτες, αξιολογώντας τελικά ποια χώρα είχε επιζήμιες φορολογικές πρακτικές. Και στη δική μας την έκθεση βάσει των κριτηρίων αυτών των αντικειμενικών μπορούμε πραγματικά να δούμε ποιοι προωθούν επιζήμιες πρακτικές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε σε μια πρώτη φάση να έχει μαύρο κατάλογο, έπειτα θέσπισε και τον γκρίζο κατάλογο και έπειτα αποφάσισε να έχει διαφοροποιημένη στάση απέναντι στις χώρες εκείνες οι οποίες μπορεί να μεν είχαν ενταχθεί στους καταλόγους αυτούς αλλά εν συνεχεία αποφασίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι πρακτικές τους δεν ήταν τελικά επιζήμιες. Τώρα η Βραζιλία εντελώς ειδική και ξεχωριστή περίπτωση. Δεν κατονομάζω ούτε κατηγορώ κάποια χώρα. Η Βραζιλία πάντως έχει καθεστώτα τα οποία θα μπορούσαν να υπαχθούν στο κριτήριο 2 που έχει να κάνει με την φορολογική δικαιοσύνη. ενδεχομένως να υπάρχει κάποια χώρα στο Συμβούλιο που να έχει αντιταχθεί τελικά στη συμπερίληψη της Βραζιλίας στο μαύρο ή τον γκρι κατάλογο. Μπορεί και αυτό να εξηγεί τελικά την απουσία της χώρας αυτής. Ο κύριος Μουταγλία πάλι έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, πρέπει πραγματικά τώρα να αντιδράσω σε σχέση με τις δηλώσεις αυτές που ακούσαμε. Και ειλικρινά πρέπει να επιμείνω στο ότι η καζόμενη αυτή πολιτικοποίηση της διαδικασίας θέσπισης του καταλόγου πραγματικά είναι υπερβολική. Όσον αφορά τη διαδικασία ανάλυσης και διεξοδικού ελέγχου των ε, φορολογικών επικρατιών κατά τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2017 όσον αφορά την εργασία των εμπειρογνωμόνων που εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταφέραμε εκ του σύνεγγυς να δούμε γιατί υποστηρίζαμε τους εμπειρογνώμονες αυτού. Πρέπει να σας πω ότι όλες, όλοι αυτοί οι φορείς δεν επηρεάστηκαν από πολιτικούς λόγους ε, κατάφεραν να λειτουργήσουν εντελώ αντικειμενικά λόγου για τον οποίο κάποιε χώρε δεν εμφανίζονται ούτε στο μαύρο ούτε στον γκρι κατάλογο είναι το ότι η ανάλυση που έγινε βάσει των κριτηρίων που έχουμε, που ενδεχομένω ορισμένα θεωρούν ότι δεν επαρκή, πάντω με βάση τα κριτήρια αυτά έγινε η ανάλυση, κατέληξε σε ένα συγκεκριμένο συμπέρασμα βάσει του οποίου οι συγκεκριμένε χώρε δεν εντάχθηκαν στου καταλόγου αυτού. Σε καμία περίπτωση το αποτέλεσμα αυτό δεν ήταν αποτέλεσμα πολιτική πίεση που ασκήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσω μιλώντα ω μη κυβερνητική οργάνωση, βλέποντα τι συμβαίνει στην κοινωνία και στα μέσα ενημέρωση. Για μένα αυτό που αντιλαμβάνεται κανεί αντι, αντι, αντιστοιχεί και στην πραγματικότητα. Αν λοιπόν η διαδικασία δεν ήταν διαφανή, είναι προφανέ το συμπέρασμα ότι η διαδικασία αυτή ήταν ε, πολιτικοποιημένη. Ακού, διαβάζαμε άρθρα κάθε εβδομάδα ε, ότι οι Βερμούδε ασκούν πίεση προκειμένου να μην μπουν στο μαύρο κατάλογο. Ε, και το έλεγαν μάλιστα δημοσίω. Δεν θέλουμε. Λοιπόν, ε, προφανώ ε, ε, εμά αυτό μα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η διαδικασία αυτή ήταν πολιτικοποιημένη. Αφού υπήρχαν σχετικέ αναφορέ στα μέσα ενημέρωση. Αν το Συμβούλιο λοιπόν θέλει να νομίζουμε ότι η διαδικασία αυτή δεν ήταν πολιτικοποιημένη, τότε θα πρέπει να είναι διαφανέ όσο γίνεται και βεβαίω από εκεί και πέρα εμεί είμαστε απόλυτα διατεθειμένοι να σα πιστέψουμε. Ευχαριστώ η κυρία Λόπε από την ΚΟΥΑ. Bueno. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λόπεθ Μπερμέχο. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ και τα μέλη του πάνελ για τις ε, παρεμβάσεις και για το χρόνο που μας αφιερώνετε σήμερα. Λυπάμαι που η πρόεδρος ε, της ομάδας του κώδικα δεοντολογίας δεν θεώρησε σημαντικό να έρθει στη συζήτηση αυτή. Ελπίζω πραγματικά να μην είναι προφάσεις όλα αυτά για να μην συμμετέχουν άλλα θεσμικά όργανα. Δυστυχώς τι διαπιστώνουμε σταδιακά και βαθμιά απομειώνεται ε, αυτός ο κατάλογος. Και δυστυχώς φαίνεται ότι αν χρησιμοποιήσουμε τα ίδια κριτήρια με το Συμβούλιο, το Συμβούλιο έχει κάνει ένα κατάλογο 17 χωρών που έχουν γίνει 9 και μάλλον την Παρασκευή θα μείνουν 7 και το δίκτυο φορολογικής ε, δικαιοσύνης καταλήγει σε 41 χώρες, ενώ η Oxfam σε 35, σε αντίστοιχους καταλόγους. Εγώ δεν θα επιμείνω, έχουν ε, γίνει πολλές εξηγήσεις και δοθεί, αλλά δεν ε, είναι πολιτική διαδικασία λέτε, αλλά έτσι φαίνεται μάλλον. Και χειρότερα ο κόσμος αυτό πιστεύει, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει σε αυτό το πολιτικό παιχνίδι και δεν χρησιμοποιεί αντικειμενικά κριτήρια για την κατάρτιση αυτών των καταλόγων. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα ε, έχει ορίσει κάποιους δείκτες ε, φορολογικής, ε, επιθετικής σχεδίας και πολιτικής για την Ιρλανδία, τη Μάλτα, το Βέλγιο, την Κύπρο, το Λουξεμβούργο, την Ουγγαρία κλπ είναι χώρες που εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες που είναι φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή. Ας μην γελιόμαστε και χωρίς κοσμητικά επίθετα. Ο ίδιος ο Επίτροπος Μοσκοβισή είπε εδώ στο Κοινοβούλιο ότι είναι σε συνομιλίες λέει με τα κράτη-μέλη και ότι ορισμένα θεωρούσαν ότι άδικα έχουν συμπεριληφθεί σε ένα τέτοιο κατάλογο. Παρόλα αυτά πρόκειται για τις ίδιες χώρες πάνω κάτω που καταλήγουν σε όλες τις λίστες των υπόπτων. Και έχω δύο ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν πιστεύετε ότι με τα στοιχεία αυτά είναι πάρα πολύ ρήψο κίνδυνο να αφαιρέσετε χώρες από τον κατάλογο ε, μόνο και μόνο για να υπάρχει μια δέσμευση, μάλλον όταν υπάρχει μια δέσμευση και όχι ουσιαστική πρόοδος και δεύτερη ε, ερώτηση που συνδέεται με αυτό. Πόσα περισσότερα κίνητρα πια χρειάζονται αυτές οι χώρες οι οποίες κατ' εξακολούθηση ε, πέφτουν στις ίδιες πρακτικές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μουταγλιέ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Έχω την αίσθηση ότι είναι δύο διαφορετικά τα ερωτήματα. Το πρώτο έχει να κάνει με το πώς θα βεβαιωθούμε ότι οι χώρε που εγγράφονται στην κρίζα λίστα δεν ξεφεύγουν. Το δεύτερο είναι το γεωγραφικό πεδίο και η σχέση τους με τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη. Στην πρώτη ερώτηση, όπως σας ανέφερα γίνεται σχολαστικότατη ανάλυση και παρακολούθηση των δεσμεύσεων και σε βάθος. Όταν βγεις από ένα κατάλογο δεν σημαίνει ότι τη γλίτωσες. Σημαίνει ότι ε, υφίστασε πίεση για να ε, έχεις αποτελέσματα. Μπορώ να σας διαβεβαίωσω ότι οι συνομιλητές μας αρχίζουν αυτό να το αντιλαμβάνονται, να το καταλαβαίνουν και να αισθάνονται ότι τα λέμε σοβαρά αυτά. Και θα πρέπει τελικά να έχουν αποτελέσματα. Για το δεύτερο ζήτημα που ρωτήσατε, όπως ανέφερα στην εισαγωγή μου, Το εγχείρημα αυτό σχεδιάστηκε και προωθήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2016 ε, στην ανακοίνωση για την εξωτερική μας στρατηγική ως εργαλείο ε, άσκησης πολιτικής και σχέσεων με τρίτες χώρες. Ε, δηλαδή αυτός ο ευρωπαϊκός κατάλογος ανέκαθεν ε, θεωρείται ότι περιορίζεται σε τρίτες χώρες. Αυτό τι σημαίνει ότι δεν ανησυχούμε για τη χρηστή διακυβέρνηση στα φορολογικά και τι σημαίνει αυτή για την εσωτερική αγορά. Όχι βέβαια, αλλά έχουμε άλλα μέσα και εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και χρησιμοποιούμε στην εσωτερική αγορά. Το πρώτο που ομολογώ ότι είναι το ε, πιο προσφυλές μέσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η νομοθεσία και έχουμε πάρα πολλές νομοθετικές προτάσεις που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο. Δεν χρειάζεται να τα απαριθμίσω όλα αυτά τα νομοθετήματα. Ε, και η νομοθεσία είναι πάρα πολύ ισχυρό μέσο. Για ποιο λόγο είναι ισχυρό. Γιατί έχουμε την νομοθεσία, έχουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι θεματοφύλακα των συνθήκων και βεβαιώνεται ότι γίνεται σωστά η μεταφορά και η εφαρμογή και μετά έχουμε και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεύτερο μέσο, συντονισμός και ε, ε, πίεση ομοτήμων για όσα δεν είναι νομοθεσία, που είναι ο κώδικας διοντολογίας. Βεβαίως χωράει βελτίωση και στη διαφάνεια. Εντάξει, το έλαβα το μήνυμα και ηχηρό ήταν από πλευρά σας, αλλά για να ε, προχωρήσουμε και να καλύψουμε αυτά που δεν καλύπτονται από την νομοθεσία. Και το τρίτο, στο οποίο αναφερθήκατε, έχει να κάνει με το διάλογο που έχουμε με τα δικά μας κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση της οικονομικής, τους πολιτικής δια του οικονομικού εξαμήνου. Και υπάρχουν και συστάσεις για την Ευρωζώνη. Είναι πάρα πολύ ισχυρό αυτό το μέσο και το εργαλείο και για τη φορολόγηση και από την αρχή ασχολούμαστε με αυτό και είναι γεγονός ότι θα τα δείτε στι συστάσει αναχώρα φέτο για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, θα γίνει τη δική αναφορά και μνήμα ε, σε θέματα φορολογικής, επιθετικής φορολογικής πολιτικής. Δεν θέλω να επικεντρωθώ στις αδυναμίες σχετικά με την ένταξη χωρών στον Μαύρο Κατάλογο, αλλά θέλω να πω το εξή. Εφόσον υπάρχουν αδυναμίες, προφανώς δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί στα σοβαρά ο κατάλογος αυτός, ανεξάρτητα από το ποιος είναι, ποια είναι τα κριτήρια που έχουν χρησιμοποιηθεί. Πρώτον, ποια είναι αυτά τα, ποιες είναι αυτές οι αδυναμίες. Για τα δημόσια κριτήρια, που είναι δημόσια και αντικειμενικά, έχουμε πει ότι τα κριτήρια αυτά ενισχύουν διακρίσεις εις βάρος χωρών χαμηλότερου εισοδήματο. Δεύτερον, τα, τα κριτήρια που δεν είναι αντικειμενικά επαληθεύσιμα ε, δυστυχώς ε, αξιοποιούνται από χώρες οι οποίες είναι διαβόητες για το ότι αποκρύπτουν σοβαρά αφορολογικά τους στοιχεία. Είναι σημαντικό λοιπόν να, να έχουμε καθαρή εικόνα για το τι γίνεται μέχρι στιγμή και τι θα κάνουμε και από εδώ και πέρα. Τι γίνεται σε αυτή την ομάδα για τον κώδικα ε, δοντολογίας. Είναι χρήσιμη αυτή η συζήτηση. Η ανάλυση που δημοσιεύσαμε στο περιοδικό Διεθνής Ανάπτυξη φέτος δείχνει ότι οι αμερικανικές πολυεθνικές το μερίδιο των παγκόσμιων κερδών που δηλώνουν για φορολογικούς σκοπούς σε δικαιοδοσίες πέραν των, ε, των χωρών όπου έχουν την οικονομική δραστηριότητα από το 1980 έχει ανέβει από το 5% στο 20-25% και το μεγάλο μέρος αυτής της ε, μεταφοράς των κερδών κατευθύνθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα Ιρλανδία, κάτω χώρες και Λουξεμβούργο. Άρα, αν δούμε τις δραστηριότητες αυτών των πολυεθνικών που μετέφεραν τα κέρδη τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εύλογα οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι κάποιες χώρες ε, ε, λειτουργούν ως φορολογική παράδειση. Και αυτό ε, είναι ένα στοιχείο που πρέπει, μας οδηγεί και στην ανάγκη να μεταρρυθμιστεί η λειτουργία αυτής της ομάδας για τον κώδικα διοντολογίας. Ευχαριστώ. Λέω Πρόεδρος. Ο Μπέρναντ Μόνοτ από την ομάδα INF. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Όσον αφορά τις μη συνεργάσιμες δικαιοδοσίες, πιστεύετε ότι υπάρχει ένα περιθώριο βελτίωσης, θεωρώ πως ναι. Σαφώς μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση, όχι όμως χάρη στην Ομοσπονδιακή Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει προκαλέσει η ίδια τα φαινόμενα φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής. Η φορολογική αυτή αιμορραγία λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθότι το άρθρο 63 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ελεύθερη εγκατάσταση των επιχειρήσεων. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο ακούμε ότι χώρες όπως η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο και άλλες χώρες μπορούν να προσελκύουν ευρωπαϊκές ε, επιχειρήσεις και επιχειρήσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ας μην ξεχνάμε από την άλλη ότι ε, ασχολούμεθα τελικά πολύ περισσότερο με επικράτειες όπως ε, το Τρενιδάδ και ε, το Πάγκο ή Σαντα Λουτσία, αντί ουσιαστικά να ασχολούμεθα με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακούσαμε εδώ πέρα ότι είναι εκατοντάδες δισεκατομμύρια τα ευρώ τα οποία ξεφεύγουν από τα δημόσια ταμεία και δυστυχώς εδώ πέρα δεν βλέπουμε να λαμβάνονται τα σωστά μέτρα, όπως για παράδειγμα το ότι θα έπρεπε να λαμβάνονται κυρώσεις κατά των ίδιο των πολυεθνικών εταιριών, αλλά και κατά χωρών όπως η Μάλτα, το Λουξεμβούργο, η Ιρλανδία, που τελικά καταχρώνται τους ευρωπαϊκούς κανόνες προκειμένου να επωφελούνται οι ίδιες. Επίσης, ξεχνάμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα των ΗΠΑ. Αν πραγματικά θέλουμε φορολογική διαφάνεια, θα πρέπει να ασχοληθούμε και με τι ΗΠΑ, οι οποίε εσκεμμένα καλλιεργούν ένα είδο φορολογική αδιαφάνεια. Είναι η μόνη χώρα του ΩΣΑ η οποία αποφάσισε να μην συνεργαστεί με την υποχρέωση υποβολή εκθέσεων όσον αφορά τα φορολογικά ζητήματα. Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν χώρες που αυτή τη στιγμή εμπλέκονται στο Panama Papers, οι οποίες έχουν γίνει πολύ πιο διαφανείς τελικά από τις ίδιες τις Ηνωμένε Πολιτείε. Οι πολιτείες ε, του Delaware, της Νεβάδα και της Νότιας Δακότα αυτή τη στιγμή φιλοξενούν πολύ περισσότερες εταιρείες οι οποίες φοροδιαφεύγουν απευθυνόμενο στο πάνελ και κυρίως στον κύριο Λάγκεροκ, θεωρείται ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε ή τουλάχιστον οι πολιτείε των Πολιτειών, στις οποίες αναφέρθηκα θα μπορούσαν να ενταχθούν σε ένα μαύρο κατάλογο μη συνεργάσιμων φορολογικών επικρατιών. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας, Πρόεδρος. Ο εκπρόσωπο τη Oxfam, ο κύριο Λαγκερόκα. Κοιτάξτε, για τι ΗΠΑ είναι σαφή τα κριτήρια. Πρώτον, φορολογική διαφάνεια και υπάρχουν κάποια επιμέρου κρατήρια. Τι γίνεται με το CBRS, με την υποβολή εκθέσεων. Ξέρετε ότι υπάρχουν, όπως σας είπα, τα κριτήρια και τα υποκριτήρια φορολογικής διαφάνειας. Μέχρι το 2019 θα πρέπει ουσιαστικά οι Ηνωμένε Πολιτείε να τηρήσουν τα κριτήρια του ΩΣΑ. Αν δεν το κάνουν αυτό θα πρέπει να ενταχθούν και αυτές, θεωρητικά τουλάχιστον, στον μαύρο κατάλογο. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει μέχρι το 2019, μέχρι τον Ιούνιο του 2019 για την ακρίβεια ο κύριος Μουταγλιέ. Σας ευχαριστώ κύριε Μονό. Να κάνω κι εγώ με τη σειρά μου μια παρατήρηση. Δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο στόχο για μια συγκεκριμένη χώρα προφανώς. Έχουμε, όπως σας είπα, 92 χώρες, 92 φορολογικές επικράτειες τις οποίες τις παρακολουθούμε σε βάθος χρόνου, γιατί όπως σας εξήγησα τροποποιούνται και τα ίδια τα κριτήρια και θέλουμε να δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση των χωρών αυτών. Πιο συγκεκριμένα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν κάποιοι υπερπόντια εδάφοι των Ηνωμένων Πολιτειών τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια τα οποία έχουμε θέσει και αυτό το λόγο βρίσκονται στο μαύρο κατάλογο. Αυτή τη στιγμή οι πυρωτικές τουλάχιστον Ηνωμένε Πολιτείες ακολουθούν τα κριτήρια του Συμβουλίου θα πρέπει όμως να καταβληθούν κάποιες περαιτέρω προσπάθειες από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι τον Ιούνιο του 2016 και η φορολογική μεταρρύθμιση των Ηνωμένων Πολιτειών θέτει εκ νέου κάποια ζητήματα όσον αφορά τα νέα προβλεπόμενα φορολογικά καθεστώτα τα οποία θα εγκρίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πρέπει να δούμε δηλαδή αν θα συνάδουν τελικά με τα διεθνή κριτήρια. Αλλά η εξέταση αυτή ήδη προβλέπεται να γίνει το φθινόπωρο από τον ΩΣΑ. Πρόεδρος, υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να πάρει το λόγο, να προσθέσει κάτι. Αναφέρομαι στα μέλη του πάνελ. Ναι, κύριε Κόμπαμ. Για να υπερασπιστώ το νομοσπιδιακό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αξίζει να αναγνωρίσει κανείς ότι τα πρότυπα του ΩΣΑ για την υποβολή εκθέσεων, η ε, πολυμερής ε, δυνατότητα ανταλλαγής προφοριών που είναι το μεγαλύτερο ε, βήμα για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής έχει την αφετηρία του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίς αυτά δεν θα είχαν γίνει ούτε τα υπόλοιπα βήματα στη ΣΥΠΑ κτλ. κτλ. Αυτό, το ότι είμαι κατά του μαύρου καταλόγου δεν σημαίνει ότι, είμαι κατά όλων όσων έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. αυτό θέλω να το τονίσω. Ευχαριστώ. Κύριε ε, Κύριε Πρόεδρε, έχω ένα ερώτημα για τα κριτήρια. Ε, το έχουμε συζητήσει ήδη εκτενώς. Γι' αυτό και οι γνώσεις μου είναι βαθύτερες στον τομέα αυτό. Θέλω όμως να λάβω μια πιο συγκεκριμένη απάντηση για τον τρόπο με τον οποίο τα κριτήρια χρησιμοποιούνται, εφαρμόζονται και για το ποια θα είναι τα επόμενα βήματα αυτής της διαδικασίας. Βλέπω ότι υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις που εκφράστηκαν σε σχέση με τα κριτήρια όσον αφορά τον ποιοτικό έναντι του ποιοτικού τους, ποσοτικού του χαρακτήρα είναι πολύ δύσκολα κάποια από αυτά τα πράγματα που προβλέπονται στα κριτήρια να μετρηθούν, να ποσοτικοποιηθούν και με ενδιαφέρει ε, πραγματικά να μάθω πώς η Κομισιόν με αντικειμενικό και αμερόληπτο τρόπο αξιολογεί τι ακριβώς τελικά αποτελεί δίκαιο και τι άδικο φορολογικό σύστημα. Γιατί πολλές φορές υπάρχει και αυτό που αναφέρεται ως φορολογικό dumping που κατά τη γνώμη μου είναι απλά ένας όρο προπαγάνδας που δεν σημαίνει τίποτα, είναι κενός περιεχομένου. Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα λοιπόν. Πώς θέλει η Κομισιόν να εξασφαλίσει ότι η αξιολόγηση βάσει των κριτηρίων πράγματι είναι απαλλαγμένη από ε, αξιολογικές ε, αδυναμίες. Δεύτερον, όσον αφορά τη διαδικασία, σε ποιο βαθμό η διαδικασία αυτή είναι αυτοματοποιημένη. Είπατε ότι δεν πρόκειται για... δεν υπάρχει βάση δικαίου για τη διαδικασία αυτή. Αυτό σημαίνει ότι τα κίνητρα αυτής της διαδικασίας είναι πολιτικά, υπάρχουν δηλαδή πολιτικές αξιολογήσεις και εκτιμήσεις στη βάση των κριτηρίων που πραγματοποιούνται και στη βάση και άλλων ενδεχομένω διαθέσιμων πληροφοριών προκειμένου να καταλήξει κανείς στην απόφαση για το αν μια χώρα θα πρέπει να μπει ή να βγει από το μαύρο κατάλογο. Ποια είναι η διακριτική ευχέρεια δηλαδή ε, και ποια είναι, ε, είναι οι αυτόματοι μηχανισμοί που εφαρμόζονται προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι διατηρείται ένα ελάχιστο επίπεδο διαφάνειας και ώστε το κοινό να γνωρίζει πώς ακριβώς τελικά λαμβάνονται οι αποφάσεις. Ευθύνομαι προφανώ τώρα στον κύριο Μουταγλιέ, αλλά μπορεί ενδεχομένω και άλλοι να θέλουν να πάρουν τον λόγο επ' αυτού. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρωσάτη. Για τα κριτήρια που ρωτήσατε. Πρέπει να πω ότι είτε μας αρέσει είτε όχι. Ο κώδικας δεοντολογίας έχει μια διάρκεια 20 ετών και εφαρμόζει πάρα πολύ λεπτομερή κριτήρια για να αξιολογήσει τι εστί επιζήμιο φορολογικό καθεστώς. Επί μία 20 ετία, δηλαδή έχουμε συσσωρευμένη πάρα πολύ εμπειρία ε, ε, και ε, εμπειρικά καθαρά πώς εφαρμόζονται αυτά τα κριτήρια είναι πάρα πολύ ακριβή, πάρα πολύ τεχνικά και συγκεκριμένα. Ε, ε, η συνολική έννοια είναι επιζήμιες φορολογικές πρακτικές και καθεστώτα. Αλλά είναι πάρα πολύ τεχνικά τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για να αξιολογηθεί αυτή ή ε, ένα ειδικό φορολογικό καθεστώς. Κατανοώ τι επιφυλάξει σας, ορισμένων από εσάς, γιατί δεν έχετε πρόσβαση στη συζήτηση και το επιθυμείτε, αλλά για εμά, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν κάνουμε μία αξιολόγηση ενός συστήματος, δεν έχουμε παρά μόνο ελάχιστο, αυτά, ή να μην πω καθόλου περιθώρια ελιγμών για το εάν ευθυγραμμιζόμαστε με τα κριτήρια ή όχι. Είναι πάρα πολύ τεχνική αυτή η δουλειά που γίνεται στον κώδικα δεοντολογίας. Με χαρά θέλετε να σας δώσω μια πιο λεπτομερή εξήγηση για τον τρόπο με τον οποίο ε, αξιολογούμε με βάση πέντε κριτήρια. Ναι, να απαντήσετε γραπτός, λέει ο κύριος ε, για τη δεύτερη ερώτησή σας. Αυτό γίνεται αυτόματα. Τι θα πει αυτόματα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε μια αξιολόγηση ε, εάν θέλουμε να υπάρξει μια κοινή απόφαση, περιμένουμε την απόφαση, την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δική μας εντολή είναι εμείς να προετοιμάζουμε σε τεχνικό επίπεδο την απόφαση και την αξιολόγηση την κάνει ε, η Επιτροπή του Κώδικα Διοντολογίας. Είτε πρόκειται για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε για τρίτες χώρες. Το αυτόματο δεν γίνεται έτσι κάτι με, με τρόπο αυτόματο μηχανικό. Για αυτό που λέτε. Υπάρχει μια υποψία εδώ και μια καχυποψία ότι γίνεται πάρα πολύ πολιτική η συζήτηση. Αυτή δεν είναι βάσιμη. Εγώ έχω αυτή την αίσθηση. Θα μου πείτε ότι έχω το προνόμιο να συμμετέχω στις διαδικασίες. Ε, ενώ εσείς δεν το έχετε. Δεν σας ζητώ να με, Αλλά δεν είπαμε ότι η αντίληψη είναι η πραγματικότητα. Ο καθένας αντιλαμβάνει την πραγματικότητα όπως τη βλέπει. Ε, κοιτάξτε, Το 1997 ε, τα κριτήρια αυτά που ορίστηκαν δεν είναι καθόλου ατυχή, είναι πάρα πολύ φιλόδοξα. Τα καλύπτουν όλα και τα, το, το, τους μηδενικούς φορολογικούς συντελεστές και τις επιζημιες πρακτικές κτλ. Και, αλλά το κείμενο αυτό τότε δεν ε, γνώρισε συνέχεια ούτε το άλλο του ΩΣΑ του 1998 γιατί δεν υπήρχε πολιτική βούληση στη δεκαετία του 2000 για να αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή που εντάσσεται ε, στο πεδίο εφαρμογής αυτό. Και τι συμβαίνει με το, την ομάδα του κώδικα διοντολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν πολλά τεχνικά και πολλοί δικηγόροι ε, και ε, ε, οι οποίοι κινητοποιούνται για να φροντίσεις ότι η χώρα σου δεν θα ενταχθεί σε αυτό τον κατάλογο. Αν όλα ήταν καλά και άγια δεν θα ήμασταν εδώ σήμερα εμείς. Η κατάσταση ήταν πάρα πολύ διαφορετική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Άννα Γκόμες, αντιπρόεδρος μας. Ευχαριστώ. Δεν με εκπλήσουν όλα αυτά. Ε, ότι ε, ε, γνώρισε όλη αυτή, όλο αυτό το, το σκάνδαλο και την καταγραφή ο μαύρος κατάλογος αυτός. Ούτε αποτελεσματικός είναι επειδή έχει γνωρίσει τέτοια αντίδραση και τέτοια φασαρία. Ποια είναι τα συγκεκριμένα μέτρα που θα αναλάβετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δεσμευτούν τα κράτη, ε, τα κράτη θα τα τηρήσουν αυτά. Βεβαίως ήταν πολιτική η απόφαση. Και όταν γύρισα στη χώρα μου, μου είπανε, μα πόσο ξαδιάνθρωποι είναι αυτοί που βγαίνουν και, και και κιόλας ότι στην Πορτογαλία α, βγάλαμε το Μακάο από τη μαύρη λίστα και, και θριαμβολογούσαν κιόλα. Και είμαι βέβαια ότι και σε άλλε χώρε το έκαναν αυτό. Και επανέρχομαι στο θέμα των μηδονικών φορολογικών συντελεστών. Μα αυτά ε, πώς θα τα καταπολεμήσουμε όταν τα δεχόμαστε στην ίδια μας την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι η ίδια μου χώρα από την οποία κατάγεται αυτός ο κύριος που είναι τώρα ε, πρόεδρος του Eurogroup και έχει μηδενικό φορολογικό συντελεστή ε, για ε, διαμένοντες κατοίκους που δεν είναι επίκοοι Πορτογαλίας, που είναι τεράστια κατάφορη αδικία εις βάρος των Πορτογάλων φορολογουμένων. Μα πώς μπορούμε να ακούναμε το δάχτυλο στους άλλους όταν δεν βλέπουμε τι γίνεται στην ίδια μας την αυλή. Έλλειψη των κυρώσεων που είπατε. Χαίρομαι κύριε Μουταρλιέ που λέτε ότι θα αναλυφθεί κάποια δράση και σύντομα κατά των ΗΠΑ. Ναι, πώς όμως θα γίνει αυτό. Αφού το σύστημα δεν προβλέπει κυρώσεις. Εντάξει, το σημαντικότερο είναι η πολιτική βούληση. Και δεν έχει καμία σχέση το ομοσπονδιακό αυτό που ακούσαμε. Μα ακριβώς εδώ είτε θα προχωρήσουμε προς μια ομοσπονδιακή λύση είτε θα κολλήσουμε και θα πνιγούμε σε αυτή τη φορολογική ζούγκλα των εθνικών κυριαρχιών. Φυσικά θα πρέπει να ζητήσουμε ε, κυρώσεις και αποτελεσματικές. Και πού βρισκόμαστε σε αυτή την ιδέα να προχωρήσουμε προς ένα φορολογικό σώμα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει, να ηγηθεί όπως έχουμε ζητήσει ε, σε εκθέσεις μας. Ε, θα κάνει πολύ μεγάλη διαφορά. Το 2011 15 μάλλον, είχαν αναλάβει δράση οι αναπτυσσόμενες χώρες για τις παράνομες ροές κεφαλαίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπλόκα. Τι κάνει για όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι κάνει κύριε Μουτέλνια? Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Γκόμε. Κοιτάξτε, όσον αφορά την πρώτη σα ερώτηση, όπως και εσείς έτσι και εγώ διάβασα ενδεχομένω κάποιες ε, υπερβολικές λίγο ερμηνείε που δόθηκαν στην απόφαση του ΕΚΟΦΗΝ αλλά όπως σας είπα δεν διαφεύγουμε από τίποτα όταν βρισκόμαστε στον γκρίζο κατάλογο. Αυτό σας το λέω με απόλυτη βεβαιότητα σήμερα. Ερχόμαστε σε επαφή με τις χώρες αυτές, έρχονται αυτές σε επαφή με εμά. Πολλές φορές πηγαίνουμε εμείς στα πλαίσια αντιπροσωπιών στις χώρες αυτές γιατί πραγματικά ασχολούμεθα έπειτα με πάρα πολλές λεπτομέρειες του φορολογικού τους καθεστώτος και θέλουμε να δούμε τελικά αν οι προτινόμενες από αυτές μεταρρυθμίσεις όντως αντιστοιχούν στις δικές μας προσδοκίες. Και ορισμένες τότε αρχίζουν και σκέφτονται αν έκαναν καλά που άρχισαν τη συνεργασία αυτή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί συνειδητοποιούν ότι οι δικές μας προσδοκίες είναι πάρα πολύ αυστηρές, ότι είμαστε πάρα πολύ απαιτητικοί δεν νομίζω λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλέ χώρες οι οποίες θα περηφανεύονταν τόσο πολύ γιατί βρέθηκαν σε έναν κατάλογο στα πλαίσια του οποίου χρειάζεται να καταβάλουν φοβερές προσπάθειες. Εμείς πάντω, παρακολουθούμε όπω σα είπα πάρα πολύ στενά το πώς οι χώρες αυτές τηρούν τις δεσμεύσεις τους και προσπαθούμε να καταβάλουμε, να υποβάλουμε έπειτα στα μέσα του έτους και στα τέλη του έτους μια αντικειμενική έκθεση προκειμένου πραγματικά να φαίνεται αν και κατά πόσο χώρες στηρούν τις δεσμεύσεις τους. Εν συνεχεία αναφερθήκατε σε ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται στην Ευρώπη αλλά και εκτός Ευρώπης τα καθεστώτα εκείνα όπου σας δίνουμε την υπηκότητα μιας χώρας με αντάλλαγμα επενδύσει στη χώρα αυτή και με αντάλλαγμα φορολογικά κίνητρα. Το φαινόμενο αυτό υφίσταται. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μια κάποια ανησυχία αντιμετωπίζουμε το φαινόμενο αυτό σε σχέση με τα ζητήματα δηλαδή φορολογικού ανταγωνισμού και φοροαποφυγής. Αυτό το οποίο συμβαίνει όμως είναι ότι πολύ συχνά έχουμε να κάνουμε με την φορολογία ατόμων, σε επίπεδο δηλαδή φυσικών προσώπων. Και το ερώτημα το οποίο που τίθεται είναι το όργανο το οποίο έχουμε εμείς για τη φορολογία των επιχειρήσεων στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής του μπορεί να καλύψει όλα αυτά τα φαινόμενα, ακόμα και όταν έχουμε να κάνουμε με φορολογία ιδιωτών, δηλαδή. Θέσατε διάφορα ερωτήματα, είπαμε ότι θα απαντήσουμε στα ερωτήματα αυτά. Θέσατε επίσης και το ζήτημα της μεταρρύθμισης του κώδικα της δεντολογίας, Πολλές φορές ως προς αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πει ότι θα πρέπει να δούμε το πεδίο εφαρμογή αυτού του κώδικα και έπειτα τη μέθοδο εργασίας του κώδικα αυτού και αν όντω λειτουργεί με διαφάνεια. Απαντήσεις πιο συγκεκριμένες προς αυτό θα σας δώσουμε γραπτός μετά το τέλος αυτής της ακρόασης. Τώρα, ένα ακόμα ζήτημα. Απουσία διακυβέρνηση σε παγκόσμιο επίπεδο για το ζήτημα αυτό είναι κάτι με το οποίο ασχολήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην διάσκεψη της Άντι Σαμπέμπα. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι ξεκινήσαμε από ένα επίπεδο το οποίο δεν ήταν ικανοποιητικό και νομίζω ότι όλοι λυπούμαθα τελικά που η διεθνής κοινότητα δεν συμμετείχε τελικά στη διαμόρφωση των προτύπων και των κριτηρίων, αλλά αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ότι η διεθνής κοινότητα έρχεται να ενταχθεί τελικά στο γενικότερο πλαίσιο του BEPS, όπου έχουμε πάνω από 100 χώρες πλέον. Επομένως, στο πλαίσιο αυτό μπορούμε να καταφέρουμε να διαμορφώσουμε περαιτέρω κριτήρια, να ενισχύσουμε τα κριτήρια αυτά. Έχουμε εκεί και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ως προς αυτό δεν έχω εγώ σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή περαιτέρω σχόλια να κάνω. Ευχαριστώ και Βέρνερ Λάγκεν και κλείνω τον κατάλογο ομιλητών και θα ολοκληρώσουμε με τους συζητές. Ναι, δεν ήσασταν στον κατάλογο των ομιλητών. Αλλά εντάξει, τώρα στο HDI θα προσπαθήσω να σας δώσω λίγο το χρόνο. Βέρνερ Λάγκεν και μετά ο κ. Κόμπαν. Yeah. Okay. Ε, Σύντομα. Μέχρι στιγμής, και αυτό είναι και το αποτέλεσμα της σημερινής συζήτηση η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το εργαλείο του ανταγωνισμού προκειμένου να αντιμετωπίζει ε, παραβιάσεις ε, των, ε, πολιτικής και των κανονισμών για το, του ανταγωνισμού. Μήπως λοιπόν θα μπορούσαμε και σε αυτή τη βάση να καταρτήσουμε έναν κατάλογο για τις διεθνείς εταιρείες και χώρες που ε, χρησιμοποιούν ή αξιοποιούν αυτές τις δυνατότητες επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Είναι μια εφικτή δυνατότητα αυτή που θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε. Είπατε ότι οι διεθνείς συμφωνίες κινούνται σε σωστή κατεύθυνση αλλά δεν υπάρχει βούληση επιβολής τους. Το δεύτερο που αφορά την ηθαγένεια και τα εξατομικευμένα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από αυτήν είναι, είναι ένα θέμα το οποίο δεν, είναι, δεν το έχουμε συζητήσει επαρκώς. Το είπε και ένα ακόμα. Πρέπει να το συζητηθεί αυτό. Τρίτον, φορολογική μεταρρύθμιση ΣΥΠΑ. Εξακολουθούν να κυκλοφορούν εσφαλμένα στοιχεία και πληροφορίες. Στη ΣΥΠΑ 11 ε, πολιτείες ε, ε, υπάρχουν μεταξύ των 5 50 που δεν έχουν φορολογική ε, δεν έχουν φορολογήσει των εταιρεών. Το Delaware δεν ανήκει. Ήμασταν εκεί και το διαπιστώσαμε. Αλλά η φορολογική μεταρρύθμιση του Τραμπ ε, θα οδηγήσει στο να υπάρξει ε, αμνηστία για όλες τις πολιτείες και όλες τις εταιρείες για τα τελευταία χρόνια με αυτή τη φορολόγηση του 21%. Άρα μετά την ε, φορολογική μεταρρύθμιση δεν θα μπορείς να τσιμπήσεις εταιρείες όπως ε, η Apple και γι' αυτόν τον λόγο κατά πάσα πιθανότητα είπα δεν πρόκειται ποτέ να καταλήξουν σε αυτό, σε αυτό το μαύρο κατάλογο. Θα ήθελα να το σχολιάσετε αυτό. Να κατηγορουποιήσουμε λιγάκι τις... Ε, να ακούσουμε πρώτα μαζί όλες τις ερωτήσεις. Ε, οπότε θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο όσο σαγηνευτική και αν είναι αυτή η συζήτηση για να τοποθετήσουμε τη ΣΥΠΑ σε ένα μαύρο κατάλογο ε, πρέπει να πω ότι μόλις φτάσουμε στο Brexit θα, ε, θα μπούμε και εμείς σε αυτό το μαύρο κατάλογο αλλά εγώ προσβλέπω σε, αυτό το, σε αυτή τη χρονική στιγμή επιτέλους να βγούμε ο φορολογικός ανταγωνισμός όμως κυρίες και κύριοι είναι υγιής Ακριβώς γιατί ε, καταπολεμά τη δαπάνη, την κατασπατάληση μάλλον των χρημάτων των φορολογωμένων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να διασπείρει θεσμοθετημένο σοσιαλισμό σε όλο τον κόσμο. Εγώ διαφωνώ απολύτως με την Αναγκόμες ε, θέλω την φορολογική ζούγκλα μεταξύ κυρίαρχων εθνών και κρατών που θα προσελκύουν τις εταιρείε. Δεν θέλουμε θεσμοθετημένο σοσιαλισμό κρατικό, το είχαμε με τη Σοβιετική Ένωση, με την Ανατολική ε- ε- Ευρώπη, εγώ διαφωνώ, εσείς θέλετε να τον επαναφέρετε. Τόμας Μαν, για να μας ακούνε και προσκεκλημένοι, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν υπάρχει ε, συνεδρίαση που να μην θέλει ο κύριος Κόμπουρ να κάνει το σόου του. Εμείς τα ξέρουμε αυτά, η παράσταση είναι, μην τρομάξετε. Μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είδατε τι γίνεται με τον κώδικα διοντολογίας. Βεβαίως και υπάρχει. 20 χρόνια ναι. Δεν αρκεί. Συμφωνώ. Είπατε ότι θέλετε να έρθετε και να μας τα εξηγήσετε. Τι φτάνει αυτό. Ε, ε, ε, δεν πρέπει να βγείτε στην κοινή γνώμη και να πείτε ότι έχουμε κάποια εργαλεία, έχουμε δυνατότητες παρακολούθησης. Και ο κώδικας διοντολογίας για μας δεν είναι ευκαταφρόνητο, είναι σημαντικό. Και θέλω να συγχαρώ τους συναδέλφους για την επιμονή τους, ε, για ε, το μαύρο κατάλογο, ναι ε, να το δημοσιεύουμε και ο, ο γκρίζος κατάλογος δεν σημαίνει ότι απαλλάσσει εσείς είσαι από παρακολούθηση. Αναφερθήκατε σε 92 κράτη, αλλά δεν τα ξέρει αυτά ο κόσμος. Δεν θα μπορούσαμε να τα πούμε. Ότι κοιτάξτε, σας παρακολουθούμε, αλλά όχι με τρόπο ε, πολιτικό και φιλικό, αλλά με αντικειμενικά κριτήρια για να δούμε πώ μπορεί να λειτουργήσει αυτό ο έλεγχο. Αν γίνουν όλα αυτά θα προχωρήσουμε και για τι κυρώσει Μέχρι τώρα δεν προβλέπονται καθόλου. Σε άλλου τομεί έχουμε προσφυγή επί παραλήψη, εξαγγελίε, αλλά για τι κυρώσει δεν είναι και εδώ απαραίτητο να πούμε ότι μέχρι εδώ και μη παρέκει. Αυτό περιμένει και ο κόσμο να ακούσει από εμά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λάνχεροκ. Ευχαριστώ. Να απαντήσω στην πρώτη ερώτηση ε, του κύριου Λάγκεν. Ένας κατάλογος που θα παρακολουθούμε τις εταιρείες που κάνουν ε, ε, φοροδιαφυγή. έχουμε την έκθεση ένα χώρα που αυτό είναι αποτελεσματικό για τις εταιρείε. Εκεί θα έχουμε όλα τα στοιχεία των εταιριών για να παρακολουθούμε και να αξιολογούμε εάν ε, έχουν σωστή πρακτική ή όχι φορολογικά. Και ιδιαίτερα για τους Γερμανούς εδώ θέλω να πω ότι ζητήστε από την, την κυβέρνησή σας να είναι θετική απέναντι ε, στις εκθέσεις αναχώρας. Στις 23 Μαΐου που συνεδριάζει αυτή η Επιτροπή, παρακαλώ πείτε στην κυβέρνησή σας να έχει επικοδομητική στάση και να απαντήσω στο θεσμοθετημένο σοσιαλισμό. Μπορείτε να χαίρεστε που υπάρχει μεγάλη φορολογική κούρσα και ανταγωνισμός. Για μένα δεν είναι καθόλου θεσμοθετημένο σοσιαλισμός αυτό ε, που ε, προσβλέπω. Ο Πρόεδρος. Δεν ξέρω αν θέλουν οι υπόλοιποι να απαντήσουν να κάνω ένα σχόλιο τελικό. Ε, κύριε ε, Μουταχλιέ, ευχαριστώ Πρόεδρε και για την ευκαιρία ε, για τη συζήτηση αυτή για να επανέλθω σε κάτι που είπε ο κύριος Μαν. Βεβαίως, δεν θα πρέπει να έχουμε έμονες ιδέες. Έχουμε ένα πρόγραμμα για να δούμε τα θέματα μιας φορολόγησης αποτελεσματικής, δίκαιας και σωστής είναι πάρα πολλά τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Η νομοθεσία που προτείναμε και εγκρίθηκε, όπως είπαμε, η νομοθεσία που προτείνουμε και πρόκειται να εγκριθεί ε, και ε, ε, την δημόσια έκθεση αναχώρα, το CCCTB με την ενιαία κοινή βάση φορολόγηση των επιχειρήσεων, η φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας επίσης και ο κώδικας διατολογία και η λίστα είναι συμπληρωματικά εργαλεία. Θα παρακαλούσα λοιπόν και με όρους επικοινωνίας ε, κύριε Μαν, προσπαθώ να σας πείσω ότι από την αρχή της θητείας ε, της Επιτροπής Juncker εργαζόμαστε ε, σε όλα αυτά τα επίπεδα και με τις κρατικές ενισχύσεις που σε κάθε περίπτωση αφορούν μία επιχείρηση, αλλά σε σχέση ε, με την πολιτική συγκυρία βοηθάει για να πάρουμε μια απόφαση για συστηματική νομοθεσία. Δεν θα είχαμε προχωρήσει αν δεν ε, ε, υπήρχε αυτή η δυνατότητα με τις κρατικές ενισχύσεις. Για το Μητρό Επιχειρήσεων τώρα δεν είναι αυτή η πρωτοβουλία την οποία προτιθέμεθα να αναλάβουμε. Η, δημόσια έκθεση αναχώρα είναι πολύ σημαντική όπως ακούσαμε. Θέλω να σε επιστήσω την προσοχή και στην τελευταία αναθεώρηση της οδηγίας για τη διοικητική συνεργασία, για τη διαφάνεια και τη διάθεση των πληροφοριών που έχουν οι εφορίες ε, για ε, αυτά τα κατασκευάσματα ε, της επιθετικής φορολογικής πολιτικής κάθε Αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να διαβιβάζονται έτσι ώστε να είναι σε γνώση όλων. Η λίστα λοιπόν και ο κώδικας είναι δύο μόνο εργαλεία από ένα κατάλογο πολλών μέσων και εργαλείων που έχουμε για την εσωτερική αγορά αλλά και για να γίνει πιο στιβαρό το διεθνές σύστημα που έχει τα όρια του. Αυτή είναι η φιλοδοξία του μας και τα όρια που έχουμε έχουν να κάνουν και με την ανάγκη να είμαστε αποτελεσματικοί. Ο πρόεδρος Γιούνκερ θέλει αποτελέσματα. Καμιά φορά μας επικρίνουν γιατί κάνουμε ε, πολιτική των μικρών βημάτων σταδιακά, βαθμιαία, να εδραιώσουμε την πρώτη φάση για να περάσουμε στη φαίνεται. Αυτό, ε, Αυτό μπορεί να φέρεται σε κάποιους ε, ανεπαρκές και σας ευχαριστώ για αυτό γιατί θέλετε περισσότερα αποτελέσματα αλλά έτσι θα προχωρήσουμε στο γενικότερο οικοδόμημα της δίκαιης φορολόγησης αλλά η βάση θα πρέπει να είναι πάρα πολύ γερή και σε αυτή θα εξακολουθούμε να χτίζουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Βάντεβέλτε Πολύ σύντομα παρακαλώ πολύ. Ο κύριος Κόμπαν πρώτος. Κοιτάξτε, αν είμαστε αισιόδοξοι μπορούμε να περιμένουμε νέα δεδομένα και νέα μέτρα στο μέλλον προκειμένου να παρακολουθούμε καλύτερα την εξέλιξη των καθεστώτων αυτών. Έχουμε τους βιώσιμους στόχους των Ηνωμένων Εθνών στα πλαίσια των οποίων υπάρχουν και συγκεκριμένοι στόχοι για τη μείωση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. Χρησιμοποιούνται επίσης και συγκεκριμένοι δείκτες. Προβλέπεται για κάθε επικράτεια να προβλέπονται ακριβώς ποια είναι τα κέρδη μιας πολυεθνικής επιχείρησης τα οποία δεν δηλώνονται σε ένα συγκεκριμένο τόπο, στον οποίο όμως εμφανίζεται η πολυεθνική αυτή επιχείρηση και για την φοροδιαφυγή πάλι θέλουμε να γνωρίζουμε τα παρουσιακά στοιχεία που έχει κάθε εταιρεία σε συγκεκριμένες φορολογικές επικράτειες στοιχεία τα οποία δεν είναι αντικείμενο ανταλλαγή πληροφοριών. Ήδη λοιπόν υπάρχουν κάποια μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενδεχομένως θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε και κάποια νέα μέτρα προκειμένου να υπάρχει μια μεγαλύτερη διαφάνεια. Ενδεχομένω και αυτά θα μπορούσαν να απασχολήσουν ω νέε ιδέε λίγο τη συζήτηση που κάνει η ενδεχομενω θα μπορουσαμε να δημιουργησουμε και καποια νεα μετρα προκειμενου να υπαρχει μια μεγαλυτερη διαφανεια ενδεχομενω και αυτα θα μπορουσαν να απασχολησουν ω νεε ιδεε λιγο τη συζητηση που κανει η επιτροπη σα. Η κυρία Βαντεβέλτ έχει το λόγο. Εν κατακλείδη θα ήθελα να πω ότι ο κατάλογος αυτός ασχολείται με ελάχιστα πρότυπα. Αν θέλει κανείς να προχωρήσει ακόμα περισσότερο, αν θέλει κανείς να δημιουργήσει ένα μεγαλύτερο κατάλογο, τότε θα πρέπει να ενσωματωθούν και περισσότερα κριτήρια. Προσβλέπουμε πάντως όλοι όλα αυτά τα πολύ πιο λεπτομερή και τεχνικά κριτήρια τα οποία θα θεσπιστούν για τα επόμενα χρόνια, αυτά τα οποία ακούσαμε δηλαδή. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Υπάρχει κάποιος από τους συνεισηγητές που θέλει να πάρει το λόγο. Ο κύριος Νέντερμαν ή ο κύριος Κόφοντ. Αν όχι, τότε θέλω να ευχαριστήσω όλους τους καλεσμένους μας. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που διεξήχθη. Είναι σαφές ότι ο κοινοτικό αυτός κατάλογος αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα πρόοδου. Εξακολουθεί όμως να εκκρεμεί το ερώτημα αν όντως χρησιμοποιείται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, αν χρησιμοποιούνται τα καλύτερα δυνατά κριτήρια και ακόμα πιο σημαντικό χρησιμοποιούνται ορθά τα κριτήρια αυτά. Τα κριτήρια θα πρέπει να είναι αντικειμενικά επαληθεύσιμα και κατά τη χρήση τους ενσωματώνοντας ή αφαιρώντας χώρες από τον κατάλογο δεν θα πρέπει να επηρεάζονται από πολιτικές προτιμήσεις. Στα λόγια βέβαια αυτό είναι πολύ πιο εύκολο από ότι στην πράξη. Ξέρουμε ότι και στα πλαίσια των εξοδότηση πράξεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις πιο επικίνδυνες χώρες στον τομέα του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος, δεχθήκαμε και εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αρκετή πίεση από τα λόμπι. Και ενώ γενικότερα υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο διαφάνειας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για διάφορα ζητήματα, επ' ασκήθηκε πάρα πολύ σημαντική εξωτερική πίεση. Λοιπόν, η αυξημένη διαφάνεια είναι η μόνη δυνατή λύση που έχουμε και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να διαμορφώσουμε ακόμα καλύτερα τα κριτήρια, να τα συγκεκριμενοποιήσουμε περισσότερο. Πάντως ε, είμαι πεπισμένος ότι στην τελική μας έκθεση θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα αυτά και βέβαια θα δούμε αν και κατά την έγκρισή της θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες θα υπάρχουν ακόμα στον κατάλογο. Πιστεύω ότι κατά την έγκριση της έκθεσής μας θα υπάρχουν χώρες ακόμα στο μαύρο κατάλογο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας σήμερα.